la silla. <laughs> Siempre tienes bastante espacio por lo que se Buonasera, un saluto Καλησπέρα. Ε, θα ήθελα να χαιρετήσω όλους και όλες τη συνάντηση αυτή με το πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Θα πρέπει να το εγκρίνουμε αυτό το πρώτο σημείο και σήμερα το απόγευμα Έχω μια συνάντηση που έχουν να κάνουν με ειδικά δύο σημεία, τα θεμελιώδη δικαιώματα, βασικά δικαιώματα για άτομα με αναπηρίε και το θέμα θα μας το παρουσιάσει μια πρώην αντιπρόταση επιτροπής μας αναφορών κάτι σύνοτ και από το Φόρουμ για τις Αναπηρίες στο Ευρωπαϊκό 1,5 περίπου εκατομμύρια άτομα έχουν προσυπογράψει αυτήν την αφορά και με τα παιδιά, τα μικρά παιδιά σε περιπτώσεις αναπηρίας τους θα ασχοληθούμε επίσης αλλά και γενικά με τα παιδιά και στο δεύτερο μέρος της συνάντησής μας θα ασχοληθούμε με ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα που έχει να κάνει με τη διατροφή και την υγεία και με τους γενετικά μεταλλαγμένους οργανισμούς και με τις συνήθειες της διατροφικές και το σημείο το 21 που έχει να κάνει με το σημείο που βλέπετε ε, για το Γιβραλτάρ μετά από το 26 θα στηθεί αύριο. Σήμερα και αύριο θα έχουμε άτομα που έχουν ε, προσυπογράψει το σημείο 5. Όπως σας είπα, κάθε Σινόθ και φορά και στο 7 και στο 8 επίσης ε, που ο κύριος Κατσιούλης θα μας παρουσιάσει το θέμα. Ο κύριος Κατσιούλης το σημείο 15 μετά που έχει να κάνει με την ανάγκη λήψης μέτρων σε Ευρωπαϊκή Ένωση για την κοτοπολεμήση τη σεξουαλικής εκμετάλλευση παιδιών, Ζακυλίν Ντεκρόι, μετά το 17 από τον Τζον Μπράιαν για την εξέταση των αιτήσεων για γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα και το σημείο 19 Ζιλ Μπέλ και Ρόμπερτ Φέρκερκ και το σημείο 28 που κανονικά θα έπρεπε να εξαρτηθεί από το πρωί που θα μας παρουσιάσει ο κ. Καρλ Βέτσελ και αύριο το πρωί μετά από συνάντηση των συντονιστών θα ασχοληθούν με την ετήσια έκθεση 2009 της Επιτροπής μας και το σύντομο γνωμοδότης για την Επιτροπή Περιβάλλοντος του κ. Μποστινάρο για την βιοπικιλότητα. Αυτά ήθελα να σας πω. Δεν ξέρω αν υπάρχει μια κάποια αντίρρηση για την ημερήσια διάταξη. Αν όχι, τότε εγκρίνεται. Να περάσω τώρα στο δεύτερο σημείο της ημερήσια διάταξης, έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων 23 ε, Φεβρουαρίου και 22 και 23 Μαρτίου του 2010 βέβαια. Και αν υπάρχει κάποια αντίρρηση, τότε εγκρίνονται και τα πρακτικά αυτών των δύο συνεδριάσεων, που είναι το δεύτερο σημείο της σημερινής διάταξης, τα πρακτικά αυτά. Να σα ανακοινώσω τώρα κάτι, ότι όπως κάθε φορά έχουμε το παράτημα εδώ με ένα κατάλογο αναφορών για το κλείσιμο ή το άνοιγμα αυτών των θεμάτων και έτσι οι συστάσει αυτές, αν δεν υπάρξει μια κάποια αντίρρηση μέχρι το τέλος της συνεδριασής μας, θα θεωρούν ότι εγκρίνονται. Να προχωρήσουμε τώρα, θα εξετάσουμε την πρώτη αναφορά έχει να κάνει με τα θεμελιώδη δικαιώματα την 306 του 2009 και τη ΣΥΝΟΤ. Τώρα το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Υπέβαλα την αναφορά αυτή από πραγματική εγανάκτηση το 2007 ξεκίνησε μια εκστρατεία ε, συλλογής υπογραφών από την ε, Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Αναπηρίας. Εγώ ήδη ασχολήθηκα με τη συλλογή αυτή ε, υπογραφών στην Ιρλανδία. Συγκεντρώσαμε τόσες πολλές υπογραφές που φτάσαμε τελικά στα 1,3 εκατομμύρια υπογραφές, πολύ παραπάνω δηλαδή από ό,τι χρειάζονται για την πρωτοβουλία των πολιτών. ζήτημα το οποίο είχαμε τόσο στο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα το αρχικό καθώς επίσης και στη συνθήκη τη Λισαβόνα, Έχουμε επίση και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα άτομα με αναπηρίε. και συλλέγοντα τι υπογραφέ αυτέ, γνωρίζαμε επίση ότι διανύαμε και το Ευρωπαϊκό Έτο για τι ίσες ευκαιρίε. Πολλοί χρειάστηκε να καταβάλουν πολύ μεγάλε προσπάθειε και να κάνουν θυσίε προκειμένου να συλλέξουν τι υπογραφέ αυτέ, Εγώ θυσίασα όλε τι καλοκαιρινέ μου διακοπέ. και κατάφερα να γεμίσω πάρα πολλές τέτοιες σελίδες, είναι αυτή που βλέπετε με υπογραφές. Όταν υποβάλαμε τις ε, υπογραφές αυτές ε, στην κυρία Μάλστρομ εξ ονόματος του Προέδρου Μπαρόσο, βγάλανε τότε καταπληκτικού λόγου οι τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λέγοντά μα ότι θα λάβουν υπόψη τι υπογραφέ αυτέ, ότι θα γίνουν πραγματικέ και σοβαρέ συζητήσει, ότι πραγματικά επρόκειτο να μπουν ε, στι ε, δύσκολε λεπτομέρειε του ζητήματο αυτού και ότι θα κατέβαλαν τελικά μία νομοθεσία. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια ζητάμε να υπάρχει μια συγκεκριμένη οδηγία για τα άτομα με τι αναπηρίες και να περιληφθεί επίση και το ζήτημα τη ηλικία. Και μπορώ να πω ότι η πρωτοβουλία αυτή που έλεγε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα αναλάβει εξαφανίστηκε στη συνέχεια από το πρόγραμμα εργασίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επέμενα τότε εγώ πάρα πολύ να μου πούνε τελικά πότε θα γίνει η οδηγία αυτή, πότε θα υποβληθεί η οδηγία αυτή, η πρόταση οδηγία. Και πολύ τότε, ακόμα και ο πρόεδρος Πέτερινγκ τότε μου είχε πει ότι δεν μπορούσαν να εντοπίσουν την πρόταση αυτή. Και κάποια στιγμή τελικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μου τηλεφώνησε και με ρώτησε τι πρέπει να κάνουν ε, με όλες αυτές οι υπογραφές, με όλα αυτά τα έγγραφα τα οποία είναι σε κάποια υπόγεια και μαζεύουν σκόνη. Μου είπαν τι πρέπει να κάνουμε τελικά με όλες αυτές τις υπογραφές. Θεωρώ λοιπόν ότι η δίδρασή τους είναι αρκετά προσβλητική στην αρχή. Την εποχή εκείνη συζητούσαμε μία οδηγία κατά των διακρίσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θελήσαμε τότε να καταφέρουμε να καταπολεμήσουμε κάθε μορφή ε, ε, προκατάληψης και γινόταν μια κάποια αναφορά στην ηλικία και στην αναπηρία, χωρίς όμως να είναι μια οδηγία η οποία θα κάλυπτε όλο το ζήτημα των ατόμων με αναπηρίες. Γιατί συνήθως ε, οι διακρίσεις σε βάρος των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία δεν είναι μια διάκριση που έχει να κάνει με την στάση που έχει κανείς Ανά πάσα στιγμή γνωρίζει κανείς ότι μπορεί να γίνει ανάπηρος και όλοι γνωρίζουμε ότι κάποια στιγμή θα φτάσουμε σε μια προχωρημένη ηλικία. Θεωρώ λοιπόν ότι ε, δεν μπορούμε να βάζουμε τις ε, διακρίσεις έναντι στα άτομα αυτά στην κατηγορία με τις υπόλοιπε διακρίσεις. Αυτό που είδαμε είναι ότι ε, δεν επιθυμούν οι θύνοντες να καταβάλουν τους απαραίτητους σπόρους. Αν αναλύσετε την κατάσταση θα δείτε τελικά ότι υπάρχουν ελάχιστοι πόροι προκειμένου να επιτευχθεί κοινωνική ένταξη και να εξασφαλιστούν ίσες ευκαιρίες για τα άτομα με αναπηρίες. Διάβασα και την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θεωρώ ότι η απάντηση που μας δίνουν, δηλαδή ότι η οδηγία κατά των διακρίσεων αρκεί η οδηγία διακρίσεων καλύπτει μερικό το όλο ζήτημα. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι θα πρέπει να ζητήσουμε πλήρω την αφορά αυτή, την οποία έχουν υποβάλει 1,3 εκατομμύρια πολίτε Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να έχουμε μια οδηγία για τα άτομα αναπηρίε και του ηλικιωμένου που θα εξασφαλίζει ότι θα παρέχονται οι απαραίτητοι πόροι για να προστατευτούν τα δικαιώματα των ανθρώπων αυτών. Και καταλαβαίνετε σε μια περίοδο οικονομική κρίση μια τέτοια οδηγία είναι απαραίτητη. Καταλαβαίνετε ότι στη δική μου τη χώρα, την Ιρλανδία, οι πρώτοι που πλήττονται από την οικονομική κρίση είναι οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με αναπηρίε. Και να κάνω και κάποιε παρατηρήσει και θα δώσω στη συνέχεια το λόγο στο Φόρουμ για την αναπηρία και στην Πρόεδρο. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη στην Βουλγαρία. Πάρα πολλέ υπογραφέ καταφέραμε να συλλέξουμε στη χώρα αυτή. Εργάστηκα για το ζήτημα αυτό, κυρίως για τα ορφανά παιδιά στη Βουλγαρία, τα οποία βρίσκονται σε διάφορα ιδρύματα περίθαλψης ή παιδικής φροντίδας. Η κατάσταση εκεί πέρα είναι πάρα πολύ δύσκολη και νομίζω ότι θα πρέπει να αντιδράσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενεργοποιώντας την διαδικασία της πρωτοβουλίας του πολίτη ειδικά για τη χώρα αυτή, για την Βουλγαρία. Σας ευχαριστώ πολύ. Λεμφόρε, Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Αναπήρων, που έχουμε 70 εκατομμύρια πολιτών με αναπηρίες ε, στα πλαίσια αυτού του φόρουμ, είναι 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και Νορβηγία, Ισλανδία, Αλβανία, πρώην Δημοκρατική Πρωτοδημοκρατία της Γερμανίας και με άτομα ακριβώ που έχουν αναπηρίες και το φόρουμ σήμερα είναι ε, ακριβώ ο οργανισμός που εκφράζει τις απόψεις των ατόμων αυτών. Είναι σημείο κλειδί διαπραγματεύσεις ε, με την Επιτροπή, με τον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών. 65 εκατομμύρια τουλάχιστον έχουν αναπηρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η επικίνδυνη κατάσταση σήμερα που μας ανησυχεί και δικαιολογείται μια οδηγία τα άτομα αναπηρίες καθημερινά αντιμετωπίζουν διακρίσεις ε, και προβλήματα σε κάθε τομέα και δεν έχουν ίση πρόσβαση στη μόρφωση, επίσης υψηλό ποσοστό ανεργίας και χαμηλό γενικά εισόδημα. Δεν μπορούν να μετακινηθούν ελεύθερα για διάφορες καθημερινές δραστηριότητες Ακριβώ επειδή υπάρχουν δυσκολίε στα πεζοδρόμια, στη λεωφορεία και παντού σε οποιαδήποτε άλλη δημόσια πρόσβαση. Και τα προβλήματα αυτά είναι μεγάλα γιατί έχουμε εμπόδια και νομοθετικά και δεν, έχουν, δεν είναι εύκολο να εγκατασταθούν σε άλλο κράτο. Ένα τουλάχιστον εκατομμύριο διακόσχε χιλιάδε ζουν σε ιδρύματα στην Ευρώπη η εκστρατεία ένα εκατομμύριο 400.000 δείχνει έτσι γιατί πρέπει να υπάρξει μια νομοθεσία για να μην έχουμε διακρίσεις για άτομα με αναπηρίες και να κινητοποιηθεί ε, να κινητοποιηθούν τα άτομα αυτά για να δείξουμε ακριβώς τον αθέατο πολίτη στους πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να δούμε πώς έχει προχωρήσει αυτό το φόρουμ από παντού σε όλες τις χώρες συλλέξαμε υπογραφές και το 90% ήταν από άτομο σε άτομο απευθείας και όχι με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και είχαμε ένα επίσημο δικαστικό κλητήρα που έκανε ακριβώς μια επαλήθευση των ατόμων αυτών των υπογραφών τους. 4 Οκτωβρίου του 2007, 2.000 ακριβώς άτομα γιόρτασαν στο Ρόπαν Σουμάν το 1 εκατομμύριο υπογραφέ. Η Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής από την Πορτογαλία, η Υπουργό Κοινωνικών Υποθέσεων, γιατί είχαμε τότε την Πορτογαλική Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ήρθαν ειδικά στις Βρυξέλλες για να γιορτάσουν το γεγονός αυτό. Έχουμε αυτή την μεγάλη απογοήτευση όμως ε, για τα άτομα αυτά γιατί δεν είναι καθόλου θετική η απάντηση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρά την κινητοποίηση δεν είχαμε ικανοποιητική απάντηση. Στο φόρουμ μας έστειλαν ακριβώς μια επιστολή ότι εντάξει πήραν αυτή την αναφορά. Καμία ανακοίνωση όμως στους πολίτες που συμμετείχαν σε αυτή την πρωτοβουλία και το, στο, με το φόρουμ επίση δεν συνεργάστηκαν στην προετοιμασία των ρυθμίσεων αυτών. Από κοινωνική πλευρά καθόλου στο κείμενο επίση που δεν ανταποκρίνεται το κείμενο αυτό στι ανάγκε των ατόμων με αναπηρίε παρόλο το εκατομμύριο και πάνω υπογραφέ. Ε, και η πρόταση αυτή δεν δείχνει το πώς γίνονται οι διακρίσεις απέναντι στα, παιδιά, στα άτομα με αναπηρίες. Η νομική βάση είναι ισχνή, το 3 της συνθήκης και όχι το 13 και 95. Το 4 είναι εντελώς λόγο και αποδυναμώνει τις πιο προχωρημένες εθνικές νομοθεσίες και δεν καθορίζει για κύριους τομείς όπως η μόρφωση και οι οικονομικές υπηρεσίες ένα πλαίσιο δεν υπάρχει μια αναλογία να μας στην πρόταση και στην βοήθεια που προσφέρουν τα κράτη-μέλη. Ε, στρατηγική δεν εμφανίζεται επίσης σχεδόν καθόλου στρατηγική του 2020. Η πολιτική αυτή Έχουμε λοιπόν ένα εκατομμύριο που έχουν προσυπογράψει και θα πρέπει να προσπαθήσουν τα θεσμικά όργανα για μια ε, πολύ καλύτερη οδηγία ανάλογα με τις απαιτήσει και τις ανάγκες όλου αυτού του κόσμου που έχει υπογράψει αυτές τις ε, αναφορές και επίσης πρόσβαση σύμφωνα με το άρθρο 95 και η συμφωνία ε, που υποστηρίζει το φόρουμ είναι στα πλαίσια επίσης της πολιτικής στρατηγικής του 2020. Αυτό και σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Μαρία Ζουμπέρ από την Επιτροπή. Ευχαριστώ. Το θέμα εδώ νομίζω ότι άπτεται δύο ερωτημάτων. Καταρχήν τον τρόπο και το περιεχόμενο όλης αυτής της εξτρατεία που ξεκίνησε με τη συλλογή υπογραφών. Καταρχήν, να ξεκινήσω με το είδο. Αυτό πρέπει να το δούμε με υπό το φω ε, τη ε, πρωτοβουλία των πολιτών. Να σα θυμίσω ότι οι υπογραφέ ε, αποδόθηκαν στην Κομισιόν στι 22 Νοεμβρίου 2007 πριν δηλαδή από την έναρξη ισχύω τη ε, συνθήκη τη Λισαβόνα. Οπότε οι διατάξει ε, τότε δεν ήταν δεσμευτικέ για την ε, πρωτοβουλία των πολιτών. Τώρα ισχύει η συνθήκη τη Λισαβόνα. Μπορούμε να δούμε ποιε είναι οι διατάξει που ισχύουν στο άρθρο 14 και υπάρχουν και κάποια ακόμη θέματα που πρέπει να εγκριθούν όταν μιλούμε για συνθήκες και για ε, όρου που πρέπει να ισχύουν για τέτοιες ε, πρωτοβουλίε. Οπότε ακόμη δεν είναι πλήρως εφαρμόσιμες και ανεπτυγμένε οι διατάξει. Παρ' όλα αυτά, για το περιεχόμενο πρέπει να πω ότι η Κομισιόν έχει δεσμευτεί να ενισχύσει τη συμμετοχή των πολιτών και παρόλο που τότε δεν ίσχυε η συνθήκη τη Λισαβόνα, η Κομισιόν προσπάθησε ήδη να απαντήσει, να ανταποκριθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και προσπάθησε να λάβει υπόψη και το περιεχόμενο αυτής τη της ω αναφοράς το δυνατόν περισσότερο. Τώρα ο κύριος Παρόσο έστειλε μια επιστολή για να δηλώσει ότι όντως έχει λάβει τις υπογραφές και τι είδαμε, τι αναλύσαμε και μπορούσαν να ληφθούν και υπόψη γιατί ήταν αρκετά έγκαιρη η υποβολή του. Ε, όταν δηλαδή η Κομισιόν υπέβαλε την πρότασή τη για την ε, οδηγία ε, για την μη διακριτική μεταχείριση. Το Νοέμβρη του 2007 έγινε αυτό. Η οδηγία εκδόθηκε τον Ιούλιο του 2008. Οπότε μπόρεσε να ληφθούν, μπόρεσαν να ληφθούν υπόψη οι υπογραφέ όταν έγινε η αξιολόγηση επιπτώσεων και όταν υπευλήθη το τελικό κείμενο. Η Κομισιόν λοιπόν θεωρεί ότι υπάρχουν κάποια ειδικά θέματα που άπτονται των αναπηριών και πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη. Η πρόταση με την οποία, την οποία επέβαλε η Κομισιόν τον Ιούλιο έχει ένα ειδικό άρθρο, ειδικέ διατάξεις δηλαδή που αφορούν τις αναπηρίες και είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτές οι διατάξεις που υπάρχουν στην πρόταση της Κομισιόν αυτό που κάνουν είναι να εγγυώνται το ίσο επίπεδο μεταχύ, ε, προστασίας ε, όπως ε, αυτές που υπάρχουν στις ειδικές, όπως αυτή που υπάρχει στις ειδικές οδηγίες που εκδίδονται. Λήφθηκαν λοιπόν υπόψη όλες αυτές οι ειδικέ διατάξεις, καθώς επίσης και το... και γι' αυτό υπάρχει και το ειδικό άρθρο στη συγκεκριμένη οδηγία. Τώρα, για το τι συμβαίνει και πού βρισκόμαστε. Το Κοινοβούλιο έχει ήδη εγκρίνει την νομοδότηση στις 2 Απριλίου 2009. Όπως ξέρετε το Συμβούλιο ακόμη εξετάζει την πρόταση και οι διαπραγματεύσει ακόμη συνεχίζονται. Εν τω μεταξύ, η συνθήκη τη Λισαβόνα άρχισε να ισχύει, οπότε το πρώην άρθρο 13 έγινε άρθρο 19 και οι διαδικασίε επίση άλλαξαν. Οπότε παραμένει η, ε, ομοφωνία, οπότε πρέπει να ε, συμφωνήσουν όλα τα μέλη για να εγκριθεί η πρόταση. Αλλά το Κοινοβούλιο θα πρέπει να δώσει και την σύμφωνη γνώμη του. Αυτή η συνθήκη υπευλήθη μέσω της, μέσω της συνθήκης της Θα σταματήσω εδώ γιατί τα θέματα ακόμα είναι εκκρεμή. Υπάρχει λοιπόν περιθώριο ελιγμών. Θα περιμένουμε πώς θα εξελιχθούν οι διαπραγματεύσεις. Στην πρόταση σας λέω και πάλι, στην πρόταση που υπευλήθη στις 2 Ιουλίου του 2008, η αναφορά που υπεγράφει από τόσους πολίτες ελήφθη υπόψη όπως έπρεπε να γίνει. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Κυρία Γκόμες. Σας ευχαριστώ. Να σας πω ότι είναι απίστευτη η ε, πρωτοβουλία αυτή να καταφέρει κανείς να συλλέξει πάνω από ένα εκατομμύριο υπογραφές προτού καν αρχίσει να ισχύει η συνθήκη της Λισαβόνας. Και νομίζω ότι πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτό το λόγο να δώσει και μια καλή απάντηση. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης υπόθηκε ότι ε, θα πρέπει να προωθηθούν κάποιες πρωτοβουλίες. Το Intergroup για τα άτομα με αναπηρίες άρχισε να ασχολείται με ένα σύμφωνο για τα άτομα με αναπηρίες, το οποίο, με το οποίο θα πρέπει να ενταχθεί στα πλαίσια της ε, στρατηγικής για την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το 2020. Επίσης, προσπαθούμε να ασκήσουμε πίεση στα κράτη-μέλη να συνάψουν την ε, Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα άτομα αναπηρίες Ορισμένα, ορισμένα κράτη-μέλη έχουν ε, συνάψει τη συμφωνία αυτή, έχουν επικυρώσει τη συμφωνία αυτή, αλλά πάλι όχι. Και έχουμε έπειτα και την οδηγία κατά της διακρατική μεταχείρισης, την οποία ψήφισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά το πρόβλημα είναι ότι όλη η διαδικασία έχει ε, συναντήσει εμπόδια στο Συμβούλιο. Θα θέλαμε λοιπόν το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πούνε πώς θα συνεχιστεί η διαδικασία αυτή, πώς δηλαδή θα προωθηθεί η ε, εξέταση της οδηγίας αυτής που όπως σας είπα έχει μπλοκαριστεί στο Συμβούλιο. Θα ήθελα λοιπόν να μας ε, δώσετε μία απάντηση και καταλαβαίνετε πλέον ότι υπάρχει πολύ μεγάλη στήριξη από τους Ευρωπαίους πολίτες. Θέλαμε λοιπόν να ευοδοθεί όλη η διαδικασία. Κυρία Ράπτη. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Δεν θα πάρω το χρόνο που μου δίνετε, γιατί η τοποθέτηση της ε, συναδέλφου της Κίνγκα ε, με κάλυψε απολύτως. Ήταν ακριβώς αυτά που ήθελα να πω. Θα προσθέσω μόνο ότι θα ήθελα πραγματικά να ακούσω από την πλευρά της Επιτροπής πώς βλέπει όλα αυτά που ανέπτυξε η Κίνγκα και με την οποία συμφωνώ απολύτως, αλλά επίσης και το θέμα της Ευρωπαϊκής Κάρτας Αναπηρίας, για την οποία έχουμε μιλήσει κατά καιρούς και που πιστεύουμε ότι η θέσπισή της θα βοηθήσει πάρα πολύ στην μετακίνηση των ανθρώπων με ειδικέ ανάγκες μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ασφαλώς τα κράτη-μέλη θα είναι αρμόδια να ορίσουν τι είναι αναπηρία, τι δικαιώματα θα έχουν οι ανάπηροι κλπ. Αλλά μέσω της Ευρωπαϊκής Κάρτας Αναπηρίας ε, θα δοθούν εγγυήσεις και θα μπορεί να διευκολυνθεί η μετακίνηση και τα δικαιώματά τους να έχουν ισχύ παντού. Ευχαριστώ. E, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν θα επαναλάβω αυτά που υπόθηκαν ε, από τους υπόλοιπους συναδέλφους. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπαν. Όντω είναι πολύ σημαντική η αναφορά αυτή. Είναι θεμελιώδου σημασία στα πλαίσια της πρωτοβουλίας για τους πολίτες. Εγώ είμαι υπεύθυνη για αυτή τη νέα πρωτοβουλία για το 2012 και μετά. Τότε ελπίζουμε οι πολίτες να μπορούν, σύμφωνα με τη συνθήκη της Λισαβόνας, να υποβάλουν τέτοιου είδους αναφορές. Ελπίζω να γίνει αυτό. Είναι εξαιρετική αυτή η προσπάθεια που έχει γίνει. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό και θα πρέπει να το δούμε όντως σε αυτό το πλαίσιο. Ακούσαμε ήδη την απάντηση της Κομισιόν, είπε ότι είναι ικανοποιημένη με τη δουλειά που έχει γίνει και όλες οι πτυχές που αναφέρονται στην στην αναφορά μας είπαν ότι συμπεριλαμβάνονται στην οδηγία για την διακριτική μεταχείριση. Βέβαια, οι πολίτε μα είπαν ότι κάποιε από τι ανησυχίε του δεν έχουν ληφθεί υπόψη. Η Κομισιόν θα θέλαμε να μα δώσει μια πιο περιεκτική απάντηση για να απαντήσει και στα επιχειρήματα που έθεσαν οι πολίτε που λένε ότι δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι ανησυχίε του στην οδηγία κατά τη διακριτική μεταχείριση. Υπάρχουν δηλαδή κάποια γενικά σχόλια στην οδηγία αυτή και όχι ε, πολύ ειδικά ώστε να καλύπτονται οι ανησυχίες των ε, όσων υπέγραψαν την ε, αναφορά για τους, κυρίως για, τους, για τα ατομαμένα πυρία αλλά και για τους ηλικιωμένους. Θα ήθελα λοιπόν μια πιο περιεκτική άποψη, απάντηση από την ε, Κομισιόν. Ο κύριος Κάσμαν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Χαίρομαι που βλέπω εδώ την πρώην Πρόεδρο. Χαίρομαι που είναι εδώ η κάθε σύνοτ. Θα προσθέσω και εγώ την ε, δική μου υποστήριξη στις αναφορές αυτές. Ε, η πρωτοβουλία αυτή είναι πολύ σημαντική γιατί στην πολιτική όσο πιο ενεργοί είναι οι πολίτες τόσο πιο υγιής είναι και η δημοκρατία μας. Γιατί όντω ε, αντικατοπτρίζουμε τι δικέ του ανησυχίε. Βέβαια, πολλέ φορέ δεν είμαστε σε θέση να πάρουμε τα κατάλληλα μέτρα και να καλύψουμε όλε τι ανησυχίε. σε αντίθεση με την κυρία Γκέριγκερ, ε, δεν θα συμφωνήσω με αυτά που είπε. Εγώ ε, δούλεψα πολύ στενά ε, για την οριζόντια οδηγία για, ε, τη διακριτική μεταχείριση και κάποιοι πάλι της Κομισιόν επίσης έχουν χρόνια που εργάζονται επί της οδηγίας αυτής και κάποιες από τις ασυνέπειες που υπάρχουν τώρα και τις ανεπάρκειες αντιμετωπίζονται πραγματικά με πολύ σωστό τρόπο σε αυτή την οριζόντια οδηγία και τόσο πολύ μάλιστα που η γερμανική κυβέρνηση ήταν αυτή που είπε ότι δεν μπορεί να το υποστηρίξει αυτό στο Συμβούλιο γιατί ε, κυρίως επί τη βάση του κόστους που έχει να κάνει με τις αναπηρίες. Και αυτό είναι ένα επιχείρημα το οποίο πρέπει να το δούμε σοβαρά. Οποιοδήποτε επιχείρημα που λέτε ότι υπάρχει κόστος όταν παρέχει μια υπηρεσία αυτό σημαίνει ότι δεν θέλετε να προσφέρετε την υπηρεσία για να ικανοποιήσετε τους ε, πολίτες που πάσχουν από κάποια αναπηρία. Οπότε αποδεσμευόμαστε ουσιαστικά από όλους όσους είτε συνδέονται, είτε είναι μέλη μιας οικογένειας που έχει κάποιο άτομο με αναπηρία, είτε που συμμερίζεται τις ανησυχίες αυτών των ατόμων με, των ναι, με αναπηρία. Όλες λοιπόν αυτές οι ανησυχίες νομίζω ότι καλύπτονται στην οριζόντια οδηγία. Υπάρχει και η οδηγία, η οριζόντια, και η οδηγία πλαίσιο για την, ε, ε, για την απασχόληση και οι υπόλοιπε τομεακές οδηγίε, οι οποίε πραγματικά δείχνουν πόσο μεγάλη διακριτική μεταχείριση υπάρχει ακόμη. Αν δηλαδή υπάρχει διακριτική μεταχείριση ε, έναντι, κάποιου αναπήρου, μπορεί κάποιο να πει ότι ναι, αλλά και εγώ είμαι θύμα διακριτική μεταχείριση λόγω τη εθνικότητά μου ή λόγω του χρωματό μου. Η οδηγία λοιπόν η οριζόντια το καλύπτει αυτό. Η Κομισιόν και ο πρόεδρος Μπαρόσο είπαν ότι δεν θα υπέβαλαν μία οδηγία που θα είχε να κάνει με τα όσα παραμένουν εκκρεμία από το παλιό άρθρο 13. Είχαμε δηλαδή τις ε, ομάδες ε, ε, ομοφιλοφίλων, θρησκευτικές ομάδες, όλοι αυτοί και η πίεση που άσκησαν ήταν αυτή που άλλαξαν την άποψη του Προέδρου και έχουμε αυτή την οδηγία τώρα. Τα περισσότερα λοιπόν από τα προβλήματα, νομίζω εγώ, για την ελεύθερη μετακίνηση, για την ελεύθερη πρόσβαση στις υπηρεσίες, υπάρχουν, αναφέρονται. Θα διαφωνήσω λοιπόν και με την ε, κάθε σε ένα σημείο για τις, ε, για τις ομάδες ομοφιλοφίλων, για τις εθνοτικές ε, μειονότητες, για τις θρησκευτικές μειονότητες. Δεν είναι ότι αδιαφορούμε ή δεν συμφωνούμε ή δεν μας αρέσουν αυτοί οι άνθρωποι. Κάποιοι όντως εξακολουθούν να, να ε, να δείχνουν διακριτική μεταχείριση εναντί αυτών των ανθρώπων. Έχω δει ανθρώπου να τους διώχνουν από τα αστιατόρια γιατί τους κάνουν κακή διαφήμιση. Αν λοιπόν δεν δεχτούμε τον κοινό παρονομαστή που υπάρχει σε οποιαδήποτε πτυχή διακριτική μεταχείριση δεν πρόκειται να την αντιμετωπίσουμε ποτέ. Η οδηγία λοιπόν αυτή τη Κομισιόν θεωρώ ότι είναι ο σωστό τρόπο για να το κάνουμε αυτό. Το Κοινοβούλιο αναθεωρεί στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ την οδηγία και εγώ στενά ε, συνεργάζομαι και με το Φόρουμ για τι Αναπηρίε και με όλους όσους ασχολούνται με το θέμα, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οτιδήποτε λείπει θα συμπεριληφθεί. Αλλά ας είμαστε συγκεκριμένοι, ας μην είμαστε γενικόλογοι, ας εξασφαλίσουμε ότι η νομοθεσία που προτείνουμε θα εγκριθεί από 27 κράτη-μέλη. Δεν υπάρχει δικαιολογία να παραμένει το θέμα αυτό έκρεμες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη που έφτασα καθυστερημένος. Συνάντησα κάποια, κάποια προβλήματα καθώς ερχόμουν. Παρ' όλα αυτά γνωρίζω πολύ καλά το περιεχόμενο της ε, αναφοράς και συμφωνώ 100% με τον κύριο Κάσμαν και συμφωνώ με την απάντηση που έδωσε. Η αναφορά αυτή αναφέρεται σε γνήσεις πραγματικές ανησυχίες και στην προηγούμενη θητεία του Κοινοβουλίου συζητήσαμε το ζήτημα αυτό, αν θα πρέπει να έχουμε μια οριζόντια οδηγία, αν θα πρέπει να έχουμε μια τομεακή οδηγία όσον αφορά συγκεκριμένε μορφέ αναπηρία ή αν θα πρέπει να καλύψουμε μορφέ αναπηρία που δεν καλύπτονται καθόλου από το κοινοτικό δίκαιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο παρελθόν είπε ότι προτιμά μια οριζόντια οδηγία μια οδηγία πλαίσιο για τις αναπηρίες και νομίζω ότι είναι σημαντικό να επιμείνουμε στη θέση αυτή. Σε καμία περίπτωση δεν θέλω να αντιταχθώ σε ανησυχίε που εκφράζονται από την αναφορά αυτή αυτό που λέω ουσιαστικά είναι ότι πολλέ από τι ανησυχίε αυτέ καλύπτονται ήδη από την ε, οδηγία που έχουμε. Αν παρόλα αυτά βέβαια υπάρχουν κάποιοι τομεί που δεν καλύπτονται, τότε θα πρέπει να καλύψουμε του τομεί αυτού, να δούμε πώ τα ζητήματα αυτά, τα πιο εξειδικευμένα, μπορούν να καλυφθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι δεν πρέπει να ξεκινήσουμε πάλι από το μηδέν, να ξεκινήσουμε πάλι από την αρχή μια ολόκληρη συζήτηση για το αν θα πρέπει να έχουμε τομεακή εξειδικευμένη οδηγία ή οριζόντια οδηγία. Και ένα ζήτημα τεχνικής φύσης. Μπροστά μας έχουμε μία αναφορά. Δεν είναι πρωτοβουλία των πολιτών αυτό ακόμα. Είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε τη διάκριση αυτή. Ανάμεσα στις αναφορές μπορεί οποιοδήποτε να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή ακόμα και ομάδα πολιτών είτε πρόκειται για ένα εκατομμύριο, είτε πρόκειται για πέντε εκατομμύρια, είτε πρόκειται για έναν μόνο αναφέροντα. Ένα πράγμα είναι αυτό, η αναφορά, που μπορεί να υποβάλει, όπω σα είπα, οποιοδήποτε πολίτη καλώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει δράση για παρατυπίες που έχουν συμβεί. Άλλο λοιπόν είναι αυτό και άλλο είναι η πρωτοβουλία των πολιτών που προβλέπει ότι ένα εκατομμύριο πολίτες και άνω από 7, 9 ενδεχομένως κράτη-μέλη μπορούν να ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ασχοληθεί με ένα συγκεκριμένο ζήτημα και να νομοθετήσει γι' αυτό. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να αντιδράσουν με επίσημο τρόπο στο αίτημα αυτό, όχι όμω μέσω τη Επιτροπή των Αφορών. Βέβαια, ελπίζω ότι η Επιτροπή των Αφορών θα εξακολουθήσει να δραματίζει σημαντικό ρόλο και στα πλαίσια τη διαδικασία πρωτοβουλία των πολιτών. Πάντω, θα πρέπει να τραβήξουμε μια διακριτική γραμμή ανάμεσα στι δύο αυτέ ε, μορφέ αίτηση. Από τη μια τι αναφορέ και από την άλλη την πρωτοβουλία των πολιτών. Σε κάθε περίπτωση θα λάβουμε υπόψη μα όλα τα ζητήματα τα οποία περιγράφονται στην αναφορά αυτή και εφόσον χρειαστεί θα δούμε πώς καλύπτονται από την ε, οδηγία πλαίσιο. Πάντως πιστεύω ότι θα πρέπει να μείνουμε στα πλαίσια της οδηγίας αυτής και να προσπαθήσουμε να καλύψουμε όλες τις μορφές ε, διακριτικής μεταχείρισης. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Higgins. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν, να ευχαριστήσω όλους τους εθελοντές και τις ομάδες εθελοντών που έκαναν πραγματικά εξαιρετική δουλειά και υπερασπίστηκαν τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Ε, όπως πάντα στους ε, εθελοντές καταλήγουμε για να κάνουν ε, την περισσότερη δουλειά, έδωσαν τον χρόνο τους, αφιέρωσαν τη ζωή του πολλέ φορέ για την βελτίωση των ανθρώπων με, της ζωής των άνθρωπων με αναπηρία. Παρόλο που έχουν γίνει αρκετή, έχει γίνει αρκετή πρόοδος. Δεν βλέπω εγώ κάποια αντίφαση μεταξύ της ε, νομοθεσίας για την ισότητα όπως είπαν εδώ τα οι συνάδελφοι σε όλους τους τομείς της ζωής που τους υποστηρίζω. Δεν βλέπω λοιπόν να υπάρχει αντίφαση μεταξύ αυτού και της εφαρμογής της νομοθεσίας που θα αφορά περισσότερο τα άτομα με αναπηρία στην Ορλανδία. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που συνεχίζει να υπάρχει. Μία από τις αναφορές στην ομάδα, δεν είναι εδώ αναφέρον, αλλά, ή αναφέρουσα μάλλον, αλλά μιλά για την ε, αμέλεια της, ε, ε, της κυβέρνησης στην παροχή πρόνοια σε παιδιά που πάσουν από αυτισμό. Το πρόβλημα αυτό υπάρχει στην, στην Ιρλανδία. Οι γονείς των παιδιών αυτών σωστά λένε κατά την άποψή μου ότι η εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας όπως εφαρμόζεται τώρα είναι κάτι γενικό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα παιδιά λαμβάνουν την ειδική θεραπεία ή την εκπαίδευση που χρειάζονται απεγνωσμένα. Οι γονείς τους λοιπόν κατέληξαν και το απέδειξαν ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν διαφορετικοί τρόποι εκπαίδευσης που θα έπρεπε να έχει δημιουργήσει η κυβέρνηση και που είναι πολύ πιο ωφέλιμοι για τα συγκεκριμένα παιδιά. Δεν μπορεί η πολιτεία να καλύπτει έτσι με μία, με ένα, νομοθεσία τους πάντες, τις ανάγκες όλων. Φυσικά δεν πρέπει να αποδυναμώσουμε τη γενική δέσμευση, είτε σχετίζεται με αυτό που είπε ο κύριος Κάσμαν, για, την, ε, για τις σεξουαλικές προτιμήσεις, είτε αφορά τις αναπηρίες. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει πιο συγκεκριμένη νομοθεσία. Καλή είναι και η γενική δέσμευση, αλλά και πιο συγκεκριμένη νομοθεσία θα βοηθούσε. Κυρία Τζανόκα. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα κι εγώ να υπογραμμίσω ότι ε, ανέκαθεν υποστήριζα την ιδέα της ε, οριζόντιας οδηγίας, όταν το ζήτημα αυτό το συζητούσαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όταν τελικά εγκρίναμε νομοθεσία το 2007. Ωστόσο, γνωρίζουμε τώρα ότι επανεξετάζουμε την οδηγία αυτή στα πλαίσια της συνθήκης της Λισαβόνας, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη σημασία, μεγαλύτερη προσοχή σε συγκεκριμένες ομάδες πολιτών στα πλαίσια της νομοθεσίας αυτής και ότι θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στα άτομα με ειδικέ ανάγκες, στα άτομα με αναπηρίε. Αν κατάλαβα καλά, η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αφορά μόνο κάποιες νομοθετικές πρωτοβουλίες αλλά σε θεωρητικό επίπεδο τουλάχιστον. Δεν φαίνεται, ότι η Ευρωπαϊκή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει εφαρμόσει στην πράξη την νομοθεσία αυτή. Και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πάρα πολύ αργή ακόμα και στην αξιολόγηση της πραγματικής εφαρμογής των νομοθεσιών κατά των διακριτικών μεταχειρήσεων και ότι δεν, έχουν, ε, δεν έχει ασχοληθεί ακόμη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τις διάφορες προσφυγές ε, επιπαραβάση που έχουν γίνει. Και νομίζω ότι και αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να εξετάσουμε. Το πώς δηλαδή τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν ή αν εφαρμόζουν τελικά στην πράξη την ε, κοινοτικέ οδηγίες όσον αφορά τη διακριτική μεταχείριση. Νομίζω ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσει στις ανησυχίες αυτές, να αξιολογήσει καλύτερα τις ε, εφαρμογή των κοινοτικών οδηγιών να δώσει μεγαλύτερη προσοχή στο ζήτημα αυτό και ζητώ ανοιχτά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας δώσει μια πιο περιστατωμένη απάντηση σχετικά με την αφορά αυτή. Κυρία Γιωτόβα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα μπορούσα να χωρίσω το θέμα σε δύο μέρη. Να δούμε πρώτα απ' όλα είναι η πρώτη σύνταξη για αυτή την πρωτοβουλία για τους πολίτες όπως προβλέπεται από τις συνδίκη της Αβώνας ή μια σκέτη αναφορά. Ε, το ουσιαστικό είναι ότι σε μια τόσο σημαντική υπόθεση μετά λίγους μήνες από τη συνθήκη της Αβώνας που τέθηκε σε ισχύ να συγκεντρώθηκαν ένα εκατομμύριο άτομα για να υποστηρίξουν τα δικαιώματα τους. Επίσης να το κάνουν και στο μέλλον. Έτσι ξεκίνησε η συζήτηση μέσω της δήλωσης Επιτροπής. Αλλά νομίζω ότι θα αποθαρρύνουμε ξεκινώντας τους πολίτες Ευρωπαίους. Από ό,τι άκουσα δεν είναι έτοιμοι με το κείμενο, με, τον κανον, με την ε, οδηγία αυτή, αλλά θα πρέπει να παροτρύνουμε τον κόσμο γιατί μετά από αυτή την πρωτοβουλία για τους πολίτες θα έχουμε και άλλες πρωτοβουλίες και εμείς σαν βουλευτές θα πρέπει να υποστηρίξουμε όλους τους πολίτες. Ελπίζω Ελπίζω και θέλω μετά από τόσα που είδαμε στις αναφορές αυτές, ελπίζω αυτή η ρύθμιση να ισχύσει για τα κράτη μέσα Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετά από τις αναφορές θα έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Εμείς χρειάζεται να δούμε εάν θα ψηφίσουμε μια ειδική ή γενικευμένη ε, οδηγία και πρέπει να δούμε την ουσία και όχι το ύφος ε, του θέματος ε, και αφού με την κυρία Σίνοτ συζητήσαμε για παιδιά και άλλα ανάπηρα άτομα η Βουλγαρία αναφέρθηκε σαν το χειρότερο παράδειγμα η κυρία Σίνοτ θα μπορούσε να πάει στη Βουλγαρία να την επισκεφθεί να δει τα πράγματα επιτόπου μετά από τη ζήτηση τότε και την ταινία του BBC ε, το ντοκιμαντέρ αυτό νομίζω ότι όλα αυτά έπαιξαν το ρόλο τους ε, παρότριναν. Βέβαια δεν θα έπρεπε να υποτιμήσω και ότι έχει γίνει μέχρι τώρα στη Βουλγαρία. Γιατί όλοι σας, όλοι σας γνωρίζετε ότι δεν γίνεται μετά από ένα σύστημα που ίσχυσε για 50 χρόνια με μία μορφή αντιμετώπιση, μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα ριζικά. Έχουν γίνει κάμποσα πράγματα βέβαια, συνεχίζεται η εργασία και τώρα αυτά τα τελευταία χρόνια, αυτού του τελευταίου μήνες ε, έγιναν πολλά για τα παιδιά από πλευράς Βουλγαρίας και δεν θα ήθελα έτσι να υποφελούνται και να κατηγορούν στα ελαφρά, ελαφρά την καρδία τη χώρα μου. Ευχαριστώ, ευχαριστώ την συνάδελφο. Η εκπρόσωπος της Επιτροπής κάτι θα ήθελε να προσθέσει γιατί αναφέρθηκε ακριβώς το όνομά της αρκετές φορές από όσους έχουν πάρει μέχρι τώρα τον λόγο σήμερα εδώ. Ευχαριστώ. Όντως κάποια πράγματα δεν τα ανέφερα. Γιατί αν οι υπογραφές μιλούν για την ε, πρόταση, για την οδηγία για, την, για τις Να τονίσω λοιπόν ότι η πρόταση ε, παρέχει το ίδιο επίπεδο προστασίας. Παρ' όλα αυτά, η Κομισιόν έχει δεσμευτεί όχι μόνο να αντιμετωπίσει τη διακριτική μεταχείριση, αλλά να εξασφαλίσει ότι τα άτομα με αναπηρία απολαμβάνουν των δικαιωμάτων τους και των θεμελιωδών ελευθεριών τους. Αναφέρθηκε κάτι και θα ήθελα να το σχολιάσω. Η σύμβαση του ΟΗΕ υπάρχει για, τα ανθρώπινα, για τις ε, αναπηρίες και ξέρετε ότι είναι η πρώτη διεθνή συνθήκη για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συμβαλόμενο μέρος στη σύμβαση αυτή. Και αυτό είναι κάτι ε, το οποίο τονίζει ιδιαίτερα έντονα η Κομισιόν. Η σύμβαση υπεγράφει και από την τότε κοινότητα και από όλα τα κράτη-μέλη και τώρα φτάνουμε στη χρονική στιγμή όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να ολοκληρώσει την, την ε, ένταξή της ως μέλος. 14 κρατημέλη ήδη έχουν, την έχουν υπογράψει και η Κομισιόν και το Συμβούλιο και τα κρατημέλη επίσης κατάφεραν να υιοθετήσουν την απόφαση και τα συμπεράσματα για την σύμβαση. Ακόμη μιλούμε για τον κώδικα διοντολογίας, ο οποίος πρέπει να εγκριθεί πριν από την τελική έγκριση των μέσων, των εργαλείων. Αυτό βέβαια θα μας ε, διευκολύνει σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της ε, σύμβασης. Η σύμβαση λοιπόν είναι το ορόσημο για την ε, πολιτική που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για τις αναπηρίες. Η σύμβαση λοιπόν είναι μια, ένα μεικτό εργαλείο. Κάποιες αρμοδιότητες εμπίπτουν στα κράτη-μέλη, κάποιες εμπίπτουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αυτό που προσπαθούμε εδώ να κάνουμε είναι να συνεργαστούμε σε διάφορα επίπεδα και να χρησιμοποιήσουμε όσα εργαλεία έχουμε περισσότερα. Και ένα από τα εργαλεία είναι η νομοθεσία. Τα άλλα είναι η συνεργασία. Συνεργασία σε, υψηλό επίπεδο για τις, με ομάδες που ασχολούνται με τις ε, αναπηρίες. Ομάδα υψηλού επίπεδου για τις ετήσιες εκθέσεις για την εφαρμογή. Δηλαδή ακόμη και χωρί αυτό το επίσημο βήμα τη ένταξη, α πούμε στην σύμβαση συνεργαζόμαστε όσο το δυνατόν περισσότερο και υπάρχουν πολλά θέματα όπω η, ανεξάρτητη, ε, η ζωή ανεξάρτητα των ατόμων αυτών. Άλλα θέματα. Είναι πολλέ από τι πρωτοβουλίε που έχουν αναφερθεί στην ομάδα του επίπεδου και στην έκθεση που έχει εκπονήσει για τι αναπηρίε. Και η Κομισιόν λοιπόν και τα κρατημέλη προσπαθούν να δώσουν μια πλατφόρμα για τα κρατημέλη, έτσι ώστε να μπορούμε να συζητήσουμε σε ένα, σε ένα επίπεδο ειδικά για, τα, για τους αρμοδιότητες που είναι μικτές. Η Κομισιόν τώρα εργάζεται σε ό,τι αφορά την ε, νέα πολιτική, νέα στρατηγική για τις αναπηρίες. Η παλιά μας ε, στρατηγική τελειώνει στο τέλος του 2010, οπότε τώρα η Κομισιόν θα υποβάλει μια νέα στρατηγική. Υπάρχει Σύμβαση για τα άτομα με αναπηρία του ΟΗΕ, που είναι, όπως σας είπα, το ορόσημο που μας εμπνέει για να εκπονήσουμε εμεί τη δική μας πολιτική. Είναι λοιπόν η αναφορά μας για την εκπόνηση της στρατηγικής μας και τη λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη. Τώρα, αναφέρθηκαν κάποιες ειδικέ ομάδες αναπήρων. Ίσως ε, να μην ε, ε, μακρηγορήσω επ' αυτού, αλλά να σας διαβεβαιώσω ότι η πρόταση αυτή και αυτή, αυτό, αυτή η έκκληση για την ενιαία οδηγία είναι θέμα με το οποίο ασχολείται η Κομισιόν και πρέπει να σας πω σε όλους ότι προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Μήπως ε, θα ήθελα να σας παρουσίασα το θέμα ή να πούν κάτι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ε, σαφώς συζητήσαμε για την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Πρόκειται όμως για μια σύμβαση η οποία είναι όντως εξειδικευμένη στα άτομα με αναπηρίες. Τα ίδια τα Ηνωμένα Έθνη έχουν συνειδητοποιήσει ότι χρειάζεται μια εξειδικευμένη σύμβαση. Σαφώς η ε, οριζόντια οδηγία μπορεί να έρθει να συμπληρώσει τα μέτρα τα οποία πρέπει να υπάρχουν για τα άτομα αναπηρίε. Δεν μπορεί όμως να αντικαταστήσει η οριζόντια αυτή οδηγία μια πιο εξειδικευμένη οδηγία και δεν μπορεί να καλύψει τα σημαντικά προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Και αν δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη νομοθεσία, οι άνθρωποι θα συνεχίσουν να υποφέρουν. Και υπογράφω τη λέξη, και υπογραμμίζω, με συγχωρείτε, τη λέξη αυτή, να υποφέρουν. Γιατί δεν θα υπάρχουν οι απαραίτητοι χρηματοοικονομικοί πόροι. Να σα δώσω ένα ακόμα παράδειγμα. στι ΗΠΑ Πολιτείες υπάρχει νομοθεσία για τις ίσες ευκαιρίες, για την ίση μεταχείριση. Υπάρχει όμως και μία συγκεκριμένη νομοθεσία για τα άτομα με αναπηρίες. Όταν εγκρίθηκε η νομοθεσία αυτή εξειδικευμένη στι ΗΠΑ, η ποιότητα ζωής των ανθρώπων με αναπηρίες τα δικαιώματά τους, η προστασία των ανθρώπων αυτών βελτιώθηκε πάρα πολύ σημαντικά. Πρόκειται λοιπόν για μια αμερικανική νομοθεσία η οποία είναι εξειδικευμένη στα άτομα με αναπηρίες και ακριβώς αυτό ζητάνε και τα 1,3 εκατομμύρια άτομα τα οποία υπέγραψαν την αναφορά. Είτε ονομάσετε την αφορά αυτή η πρωτοβουλία των πολιτών, είτε όχι, δεν έχει καμία σημασία. Ουδέποτε είχαμε μια τέτοια εκστρατεία, ουδέποτε είχαμε μια τέτοια συσπήρωση των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση για ένα συγκεκριμένο ζήτημα. Θεωρώ λοιπόν ότι η απάντηση που μα δίνεται αυτή τη στιγμή και η αντιμετώπιση που έχουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι προσβλητική. Ήρθα εδώ πέρα με ελπίδα και δεν θα ήθελα να φύγω αποθαρρυμένη. Πιστεύω ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε του πολίτε αυτού που υπέγραψαν. Αν εξετάσουμε τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών θα δούμε ότι η Σύμβαση αυτή λέει ότι πρέπει να ακούμε τα άτομα με αναπηρίε, να γνωρίζουμε ποιε είναι οι ανάγκε του. Και ακριβώ αυτό θέλουμε να προωθήσουμε και μέσω τη αναφορά αυτή. Να δούμε ποιε είναι οι πραγματικέ ανάγκε των ανθρώπων αυτών. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να μείνει ανοιχτή η αναφορά αυτή. Πρέπει να ασχοληθείτε περισσότερο με την, με την αναφορά αυτή. Δεν μπορεί να κλείσει τώρα εδώ. Θα ήθελα ειλικρινά να ευχαριστήσω την Επιτροπή Αναφορών γιατί ασχολείται με την αφορά αυτή για τα άτομα αναπηρίας και να μας βοηθήσει για να βελτιώσουμε την τύχη του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το φόρουμ είναι έτοιμο πάντα να συζητήσει για μια οδηγία. Όλες οι ανάγκες αυτών των ατόμων θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Ευχαριστούμε. Κάσμαν. Κάσμαν, ε, Ναι, Πρόεδρε. Για να προτείνω κι εγώ κάτι επικοδομητικό. Θα έλεγα να στείλουμε τις αναφορές στον Ραούλ Ρομέβα, που είναι ο εισηγητής για την οριζόντια οδηγία πλαίσιο στην ΛΥΜΠΕ και να ζητήσουμε σχόλια και ό,τι υπάρχει που, έχει, που δεν είναι ότι δεν υπάρχει μάλλον στην, στην οδηγία, να υπάρξει δυνατότητα να το συμπεριλάβουμε τώρα, στα πλαίσια της φάσης αυτής της προπαρασκευής δηλαδή. Ίσως να ήταν αυτός ο πιο γρήγορος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, παρά να περιμένουμε πότε θα μας έρθουν τα αποτελέσματα. Ε, Πιστεύω ότι έχει το, ε, την υποχρέωση αυτή η Επιτροπή, αφού ακούσαμε και τους συναδέλφους, να θεωρήσει ότι παραμένει ανοιχτή αυτή η αναφορά και περιμένουμε και ορισμένες νέες πρωτοβουλίες για τα θέματα αναπηριών. Και να διευκρινίσω κάτι επισήμως, όλοι το ανέφεραν για την πτυχή αυτή της αναφοράς Πάνω από ένα εκατομμύριο πολίτες προσυπέγραψαν. Θα ήθελα να πω λοιπόν ότι η Εκτριστική Επιτροπή τη θεώρησε σχεδόν σαν πρωτοβουλία νομοθετική και αυτό υποστηρίζει η Επιτροπή στην ε, απάντησή της. Δεν είναι όμως νομοθετική πρωτοβουλία αυτή δεν υπευλήθη τότε που είχα ίσχυε αυτή η νομοθετική πρωτοβουλία, ούτε και σήμερα δεν ε, έχει γίνει κάτι τέτοιο. Είναι απλά μία αναφορά. Άρα λοιπόν εδώ αυτή η Επιτροπή έχει την υποχρέωση να ανταποκριθεί, να δώσει συνέχεια σε αυτή την έκκληση, σε αυτή την καταγγελία μπορούμε να πούμε και θα πρέπει ακόμη περισσότερο να συμμετάσχουμε γιατί είδαμε ότι ένας πολύ μεγάλος αριθμός συμπολιτών μας ε, το υποστηρίζουν. Μια οδηγία για τις διακρίσεις απαιτείται είτε μια τομεακή ρυθμισή Έχω μια προσωπική μου άποψη, θα ήθελα να την εκφράσω. Η γενική οδηγία σίγουρα θα μπορούσε να καθορίσει αρχές ε, ενάντια σε οποιαδήποτε μορφή διακριτικής μεταχείρισης. Αλλά κατά την άποψή μου δεν νομίζω ότι συγκεκριμένα θα μπορούσε να μπει στον ειδικό χαρακτήρα ενός τομέα, του τομέα αυτού με τον οποίο τώρα ασχολούμεθα. Και όπως το είπαν ε, και σε άλλες χώρες συνάδελφοι για ειδικές ε, περιπτώσεις. Ε, θα πρέπει εδώ να έχουμε ένα διπλό εργαλείο, μια τομεακή οδηγία που πέρα από την γενική να μπορέσει να μπει σε για την προστασία των πολιτών. Θα πρέπει η Εκτελεστική Επιτροπή να προσφέρει ακόμα περισσότερες απαντήσεις ε, στους πολίτες ε, αυτούς. Γιατί? Για το πώς τέθηκε το πρόβλημα ήδη εδώ και αρκετά χρόνια και μετά από τόσα χρόνια μόνο σήμερα το συζητάμε αυτό και προσπαθώντας να δώσουμε μια μορφή απάντησης. Εδώ θα προσπαθούσαμε να προσφέρουμε προτάσεις και να αποδεχτούμε όσα είπε ο κύριος Κάσμαν, δηλαδή να έχουμε μια σωστά διαρθρωμένη πρόταση που να πάει και στην εισηγήτρια και στην ε, Επιτροπή Δημοσίων Ελευθεριών για να μπούμε σε λεπτομέρειες της όλης εργασίας και ακριβώς να δούμε αυτά ειδικά θέματα στην Επιτροπή αλλά και ταυτόχρονα να υποστηρίξουν όλοι μαζί μας την πρωτοβουλία αυτή για μια τομεακή οδηγία. Καλό και θετικό θα ήταν να συνεργαστούμε με την αρμόδια λοιπόν Επιτροπή και επίσης ε, να προσπαθήσουμε να παρετρύνουμε το Συμβούλιο για μια επικύρωση. Αυτό για το Συμβούλιο δηλαδή αναφέρθηκε ιδιαίτερα σχετικά με τη Συμφωνία και θα πρέπει να σπεύσουμε. Είναι σημαντικό όλα αυτά να γίνουν αποδεκτά από όλα τα κράτη-μέλη και στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι το τελευταίο και παράλληλα και μετά από τις, τα δύο δεχόμενα που είπαμε πριν, ίσως μια γνωμοδότηση, δεν ξέρω μήπως είναι αργά από διαδικαστικής πλευράς, αλλά μια γνωμοδότηση στην Επιτροπή Δημοσιονευθεριών ακριβώς για την εργασία της, ε, αυτή που διεξάγει τώρα, αυτή τη στιγμή. Αυτή η δέσμη προτάσεων βέβαια Παραμένει ανοιχτό το θέμα της αναφοράς αυτής. Δεν ξέρω αν το δέχεστε, αν δεν δέχεστε όλη αυτή τη δέσμη. Καμία αντίρρηση. Άρα λοιπόν εντάξει αυτές οι προτάσεις που μόλις εξέφρασα γίνονται δεκτές. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και όσους προσυπέγραψαν την αναφορά αυτή. Και... Για 3, 385 του 2008 η κυρία Σνέκερς ε, δεν είναι παρούσα και πρόσωπος της Επιτροπής που είχε λάβει ήδη το λόγο για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες έχει και πάλι το λόγο λοιπόν. Ε, thank Σας ευχαριστώ. Να σας υπενθυμίσω ότι ε, ο Ναφέρον επιθυμούσε να δημιουργηθεί μια ταυτότητα αναπηρίας ευρωπαϊκή που θα αναγνωρίζεται παντού στην Ευρώπη και θα έδινε ιδιαίτερα δικαιώματα στα άτομα αναπηρίας να χρησιμοποιούν δημόσια μέσα μεταφοράς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπέρ της ιδέας της αμοιβαίας αναγνώρισης του καθεστώτος αναπηρίας στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να παραχωρηθούν ε, περισσότερα δικαιώματα στους ανθρώπους αυτούς, ιδίως να χρησιμοποιούν τα δημόσια μέσα μεταφοράς. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή, μόλον ότι δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τον ορισμό της αναπηρίας και όσον αφορά τις διαβαθμίσεις αναπηρίας, καθώς επίσης και λόγω απροθυμίας των κρατών μελών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν προτίθεται να υποβάλει μια πρόταση για την δημιουργία εθνικής ταυτότητας αναπηρία με ευρωπαϊκή αναγνώριση. Το 2008 υπευλήθη αναφορά Έκτοτε είχαμε κάποιες εξελίξει οι οποίε θα ήθελα να σας παρουσιάσω. Όπως σας είπα, μολονότι αυτή τη στιγμή δεν παρουσιάζουμε ανάλογη νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καταβάλουμε ωστόσο κάποιες προσπάθειες προς τα επιθυμίε αστικά του αναφέροντος. Το Μάρτιο του 2008 ένα πρώτο σημαντικό βήμα έγινε μέσω της ε, τροπολογία της Ρύθμιση που υπάρχει για τα δελτία στάθμευσης των ατόμων με αναπηρίε προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό μοντέλο το οποίο θα αναγνωρίζεται σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε δηλαδή μια αμοιβαία αναγνώριση του καθεστώτος αναπηρίας όσον αφορά το δικαίωμα στάθμευσης και Ζητήθηκε τότε να επεκταθεί η αναγνώριση του δικαιώματο αυτού στα 12 κράτη-μέλη τα οποία προσχώρησαν στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση την εποχή εκείνη. Έχουμε λοιπόν το καθεστώς αυτό της αμοιβαία αναγνώρισης αλλά η αναγνώριση του καθεστώτος αναπηρίας εξαρτάται ακόμα από τις εθνικές νομοθεσίες. Δεν υπάρχει δηλαδή κοινοτική εναρμόνιση. Για την εφαρμογή λοιπόν της σύστασης αυτής η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε ένα εγχειρίδιο προκειμένου να εξηγήσει καλύτερα στα κράτη-μέλη πώς έχει αυτό το Ευρωπαϊκό Δελτίο Δικαιώματος Στάθμευσης και πώς θα πρέπει να εφαρμόζεται στα διάφορα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, στις ιστοσελίδες Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν περισσότερες πληροφορίες για το ποιο είναι αρμόδιο σε κάθε κράτος μέλος για το δικαίωμα αυτό, για το δελτίο αυτό της ε, στάθμευσης. Για ορισμένα ζητήματα ο αναφέρον θα μπορούσε να πάει κατευθείαν στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να δει ποιοι είναι οι θύνοντες σε κάθε κράτος μέλος όσον αφορά την χρησιμοποίηση των δημοσίων μέσων μεταφοράς και όσον αφορά την αγνώριση του δελτίου στάθμευσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σαφώς είναι υπέρ της αμοιβαίας αναγνώρισης σαφώς θέλει να προστατεύσει τα δικαιώματα και να δώσει περισσότερα δικαιώματα στους ανθρώπους με αναπηρίες και γι' αυτό το λόγο φέτος η ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέθεσε στο ακαδημαϊκό δίκτυο των ε, ειδικών σε θέματα αναπηρίας να ασχοληθούν με το ζήτημα αυτό. Το δίκτυο λοιπόν αυτόν μέχρι το τέλος του έτους θα υποβάλει μία συνθετική έκθεση όσον αφορά την ύπαρξη δικαιωμάτων ή την παραχώρηση διευκολύνσεων από το ένα κράτο μέλος στο άλλο, τα που θα απορρέουν από το καθεστώ τη αναπηρία και οι εμπειρογνώμονε επίση θα προσπαθούσουν να δούνε αν θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε μία εναρμόνιση του καθεστώτος αυτού αναπηρίας και των εναρμόνιση των διευκολύσεων και των δικαιωμάτων σε κοινοτικό επίπεδο. Πρόκειται δηλαδή για ένα αρχικό εγχείρημα το οποίο θα προσπαθήσει να, θα προσπαθήσει να εντοπίσει την αναγνώριση του καθεστώτος αναπηρίας στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από νομοθετικής πλευράς. Θα προσπαθήσει επίσης να εντοπίσει ποια τα δικαιώματα εκείνα και τις διευκολύνσεις που υπάρχουν από το ένα κράτος μέλος στο άλλο και σε ποιους συγκεκριμένους τομείς και στη συνέχεια θα προσπαθήσει να αξιολογήσει την δυνατότητα μεταφοράς των δικαιωμάτων αυτών, τη δυνατότητα αμοιβαίας αναγνώρισης αυτών των δικαιωμάτων Καταλαβαίνετε ότι ε, τα δικαιώματα αυτά, οι διευκολύνσει αυτέ μπορούν να εντοπίζονται σε διάφορου τομεί, όπω τον υγειονομικό τομέα ή τον πολιτιστικό τομέα ή στον τομέα των μεταφορών. Οι εμπειρογνώμονε θα προσπαθήσουν να συγκεντρώσουν στοιχεία από όλου αυτού του τομεί και θα προσπαθήσουν να αξιολογήσουν την δυνατότητα να προχωρήσουμε περισσότερο σε συγκεκριμένου ε, τομεί, που έχει σημειωθεί ουσιαστικά πρόοδο και που όχι και που υπάρχουν περιθώρια βελτίωση. Αυτά νομίζω ότι συνάδουν και με τα αιτήματα τα οποία έχει κάνει αναφέρον στην αναφορά του. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να πω απλώς ότι καλωσορίζω κι εγώ έτσι αυτή την ελαφριά πρωτοβουλία της Κομισιόν για την ε, ε, αμοιβή αναγνώριση. Φυσικά η αμοιβή αναγνώριση είναι μακρόχρονη διαδικασία, αλλά βασίζεται ε, και στο μοντέλο αυτό για την κάρτα στάθμευσης. Να υπάρχει δηλαδή η δυνατότητα να εισαχθεί μια τέτοια κάρτα, καθώς επίσης και η ταυτότητα για τα άτομα με αναπηρία. Έτσι ώστε όλα τα άτομα στα κράτη-μέλη να γνωρίζουν ποια είναι τα δικαιώματά τους. Νομίζω λοιπόν ότι είναι καλή η πρωτοβουλία αυτή. Ας ξεκινήσουμε και ας προχωρήσουμε μετά στην όλη διαδικασία εναρμόνισης. Ας ξεκινήσουμε δηλαδή ελαφρά και μετά μπορούμε να περάσουμε στο πιο έντονο ε, θέμα της εναρμόνισης. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κάσμαν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Συμφωνώ με την Κίνγκα. Αυτή η πρωτοβουλία είναι κάτι που θα πρέπει να ενθαρρυνθεί. Θα μπορούσαμε ίσως να αναλάβουμε και μια δράση Δηλαδή αν μπορεί να υπάρξει, να αποδειχθεί διακριτική μεταχείριση με βάση την εθνικότητα. Αν δηλαδή κάποιο είναι από κάποια άλλη χώρα και δεν μπορεί να έχει πρόσβαση ας πούμε στο, στο μουσείο επειδή είναι από άλλη χώρα και η χώρα που επισκέπτεται δεν τον αφήνει να μπει στο μουσείο δωρεάν. Θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι τέτοιο ή τέλο πάντων με κάποιο τρόπο να ενθαρρύνουμε όλο και περισσότερα κράτη-μέλη να έχουν μια, ένα είδος αμοιβαίας αναγνώρισης έστω και αν δεν είναι το απόλυτα επίσημο, ώστε να ξέρουν όλοι οι πολίτες τι δικαιώματα έχουν. Τώρα, στη φορά την ε, κάρτα που θα είναι νομικός ας πούμε εφαρμόσιμη γι' αυτό δεν ξέρω κατά πόσο έχουμε την αρμοδιότητα να το πούμε γιατί μπορούμε εμείς να πούμε ας πούμε ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να παράσχουν υπηρεσίες με τον ίδιο τρόπο όλα τα κράτη-μέλη γίνεται αυτό ας ξεκινήσουμε δεν νομίζω ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τα βασικά με την αμοιβαία αναγνώριση και έτσι με κοινή λογική πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε ένα σύστημα και για τα 27 κράτη-μέλη Ευχαριστώ Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, να προσθέσω και εγώ τη συμφωνία μου σε αυτά που είπαν οι δύο συνάδελφοι και η Κίνγκα και ο κύριος Κάσμαν και επειδή αναφέρθηκα και προηγουμένως στην Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας ε, θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό το ότι γίνεται μία πρώτη κίνηση από την πλευρά της Επιτροπής, αλλά νομίζω ότι έχει τη σημασία του να διευκρινίσουμε ότι ε, η Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας είναι κάτι πολύ πιο σημαντικό, πολύ πιο θεσμικό από την ε, Κάρτα αναπηρίας που έχει σχέση με τη στάθμευση. Το λέω αυτό γιατί η απάντηση από την πλευρά της Επιτροπής ήταν 9 δέκατα επιχειρηματολογία για την κάρτα στάθμευσης και ένα δέκατο για την ουσία του θέματος που αφορά η Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας. Εγώ μιλώντας για την Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας στην προηγούμενη τοποθέτησή μου είχα στο μυαλό μου ακριβώς αυτό που ανέπτυξε η Κίνγκα και ο κύριος Κάσμαν. Εδώ δεν μιλάμε μόνο για ζητήματα πρακτικής διευκόλυνσης. Μιλάμε για την ουσία. Μιλάμε ότι θα πρέπει να καταλάβουμε πως οι άνθρωποι με αναπηρία έχουν δικαιώματα, είναι άνθρωποι σαν όλους μας και ως κοινωνία οφείλουμε να τους διευκολύνουμε. Σε κάθε περίπτωση θέλω να ελπίζω ότι η Επιτροπή θα εργαστεί όχι μόνο έχοντας στο μυαλό της το τυπικό μέρος της υπόθεσης, αλλά το ουσιαστικό. Έχει σημασία. Ευχαριστώ. Κανείς άλλος δεν έχει ζητήσει το λόγο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα ήθελε να προσθέσει κάτι, δεν ζήτησε κανείς κάτι από την Επιτροπή. Νομίζω ότι όλοι συμμερίζονται αυτά που άκουσαν και από την Εκτελεστική Επιτροπή ακριβώς και ερμηνεύω σε αυτό που είπαν οι συνάδελφοι ότι υπάρχει πρόθεση να παραμείνει ανοιχτό το θέμα της ε, αναφοράς αυτής για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την όλη διαδικασία που νομίζω ότι φαίνεται και στα λόγια της ίδιας της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής μια πρακτική εναρμόνιση, μια πιστοποίηση, αναγνώριση παρομοίων γεγονότων και να μπορέσει κανείς να πετύχει το στόχο ακριβώς για πληρέστερη εναρμόνιση των νομοθεσιών σε θέματα αναπηριών για να φτάσουμε και σε μια αναγνώριση των δικαιωμάτων που έχουν να κάνουν με θέματα παρομοίων αναπηριών. Κανείς δεν είναι αντίθετος λοιπόν. Εγκρίνεται αυτό το να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά και να συνεχιστεί όλη η διαδικασία από πλευρά της Εκτελεστικής Επιτροπής. Κλείνει το θέμα εδώ λοιπόν προς το παρόν. Πάμε παρακάτω. David Λου μας είπε ναι πάμε στην αναφορά του 8 η 8 πριν από την 7 ο κύριος Κατσιούλης ε, έχει παρουσιάσει και την 7 και την 8 τι προτιμάει εντάξει συμφωνεί να παρουσιάσει πρώτα την 8. Ο κύριος Κατσιούλης λοιπόν για την 8. Ανεπαρκής ενίσχυση προ μαθητέ με σωματική διανοητική επιρρεπηρία στα ευρωπαϊκά σχολεία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλύτερα να τα πάρουμε όπω θα έχει η ημερήσια διάταξη. Α πούμε το 7 και μετά το 8. Πρώτα για τι ασφάλειε και μετά για τα σχολεία. Καταρχήν να πω ότι αυτά που είπε ο κύριος ε, Κάσμαν, ότι πρέπει δηλαδή να, υπάρχουν, ε, να υπάρχει περιεχόμενο στις οδηγίες που εγκρίνεται, είναι όντως θεμελιώδος σημασίας η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο. Πρέπει όντως να συμπεριλάβει τις ανάγκες αυτών ακριβώς των ανθρώπων. γιατί αυτοί είναι αυτοί που ξέρουν ε, στο πετσί τους τι σημαίνει να έχει κανείς αναπηρία και αυτοί μπορούν να δώσουν το σωστό υλικό ε, άλλο είναι να είναι κανεί ανάπηρο και άλλο είναι να έχει διαβάσει ένα βιβλίο για ανάπηρου. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Αγαπητά μέλη της Επιτροπής Αναφορών, Θέλετε να έχετε μια ευρωπαϊκή κοινότητα η οποία να συμπεριλαμβάνει τα άτομα με αναπηρία ή όχι. Θέλετε να τα κρατήσετε εντό τη κοινωνία ή εκτό αυτή. Θέλετε να υπάρχουν σχολεία ή όχι για του ανάπηρου. Φυσικά οι άνθρωποι αυτοί ανήκουν στην κοινωνία και φυσικά οι ασφάλειες, για παράδειγμα, θα πρέπει να λαμβάνουν τι ανάγκε του υπόψη. Είναι πολλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ένα ανάπηρο στην καθημερινή του ζωή, γιατί δεν λαμβάνονται ποτέ υπόψη οι, οι ιδιαιτερότητε τη φύση του. Οι άτομα με αναπηρία αντιμετωπίζονται σαν να μην αξίζει τον κόπο να ζουν. Το θέμα λοιπόν είναι να δούμε ποιε είναι αυτέ οι αλλαγέ που πρέπει να γίνουν, οι προσαρμογέ, έτσι ώστε να μπορεί κανεί να μιλά για εξίσωση των όρων ζωή των ατόμων με αναπηρία με όσου δεν έχουν αναπηρία. Πρέπει δηλαδή να υπάρξουν και νομοθετικά μέτρα. Άνθρωποι με αναπηρία θέλουν να συμπεριληφθούν στην κοινωνία. Τώρα, στις 5 ε, Μαΐου θα γίνει μια μεγάλη ε, διαμαρτυρία στο Βερολίνο ε, υπάρχει και η σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και μια δυνατή Ευρώπη μπορεί μόνο να αποτελείται από μια ε, κοινωνία η οποία συμπεριλαμβάνει όλους στους κόλπους της. Άτομα δηλαδή που, έχουν, ε, που πηγαίνουν, άτομα με αναπηρία ή παιδιά με αναπηρία που πηγαίνουν στο ίδιο σχολείο με παιδιά χωρίς αναπηρία και που δεν θεωρούνται παρείες της κοινωνίας. Πρέπει λοιπόν να τη χάνουν τις ίδιες αντιμετώπισης όπως και οι υπόλοιποι πολίτες. Η... Ε, ο παραγωνισμός των ανθρώπων αυτών μόνο ζημιά μπορεί να φέρει. Μέχρι σήμερα η Κομισιόν δεν έχει φροντίσει η... να γίνουν όλα αυτά. Και η κυβέρνηση της Γερμανίας δεν μπορούν να προστατευτούν ήδη από αύριο γιατί ακριβώς δεν υπάρχουν οι νομικές ε, διατάξεις οι κατάλληλες. Πρέπει λοιπόν να συμπεριληφθούν όλα αυτά και στην συγκεκριμένη οδηγία. Μόνο μία φωνή ακούστηκε στο Συμβούλιο αν μπορούσαμε να έχουμε ήδη από αύριο πιο αποτελεσματική προστασία των ατόμων αυτών, φυσικά θα ήταν ευχή ευχής έργων. Θα ήθελα τώρα να σας κάνω μια παρουσίαση PowerPoint. Μιλούμε για άτομα με ε, τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα χωρίς αναπηρία ε, έχουν να αντιμετωπίσουν τους ίδιους κινδύνους. Ένα ατύχημα, ας πούμε. Είτε είμαι εγώ ανάπηρος, είτε δεν είμαι τον ίδιο κίνδυνο διατρέχω αύριο να με πατήσει ένα αυτοκίνητο. Και για τον κίνδυνο αυτό, εγώ είμαι ίδιος με όλους τους υπόλοιπους σε ό,τι αφορά την ασφάλεια που πρέπει να λαμβάνω. Αν δηλαδή εγώ αύριο πάθω ένα καρδιακό επεισόδιο, ε, τον ίδιο κίνδυνο έχω να το πάθω με έναν άνθρωπο που, είναι, που δεν έχει αναπηρία. Πρέπει λοιπόν η ασφάλιση να είναι ίδια και για τους ανάπηρους και για τους ε, μη ανάπηρους πρέπει να υπάρχει ασφάλεια. Γιατί οι κίνδυνοι είναι οι ίδιοι. Πώς μπορούμε τώρα να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο ασφάλειας. Πρέπει να δούμε ποιο είναι ο κίνδυνο για τα άτομα με αναπηρία και αυτό να συμπεριληφθεί στα συμβόλαια, στι συμβάσει, τι ασφαλιστικέ. Αυτά πρέπει να συνυπολογιστούν στι κοινωνικέ ασφαλίσει. Θέλουμε να ασφαλίσουμε τα άτομα αυτά έτσι ώστε όλοι να λαμβάνουν την ίδια αποζημίωση. Είτε είναι ανάπηροι είτε δεν είναι ανάπηροι σε περίπτωση που πάθουν κάποιο ατύχημα. Το 2006 είχα στείλει στο Κοινοβούλιο μία αναφορά για την συμπερίληψη, το, για τη συμπερίληψη των ατόμων αυτών στις, ε, στις ε, ασφαλιστικές εταιρείες. Ε, η Κομισιόν το μελέτησε, το Κοινοβούλιο επίσης και προέβλεψαν κάποιες διατάξεις για τις περιπτώσεις αυτές. Βεβαίω, υπάρχουν, υπάρχουν ακόμα μεγάλα κενά. Υπάρχει και η σύμβαση του ΟΗΕ η οποία μιλά α, ειδικά και προβλέπει την συμπερίληψη των ατόμων αυτών σε ό,τι αφορά τις συμβάσεις τις ασφαλιστικές. Η Κομισιόν μέχρι τώρα έχει ένα εθελούσιο πρωτόκολλο προωθήσει για την... και πρέπει να το επικυρώσει ώστε η ανάπηροι, παρόλο που η οδηγία ακόμη δεν έχει εγκριθεί, είχε, έχει μπλοκαριστεί στο Συμβούλιο, μέσω της σύμβασης του ΟΗΕ να α, ε, προστατεύονται. Υπάρχουν λοιπόν αυτές οι δύο δυνατότητες. Είτε έχουμε την Ευρωπαϊκή Οδηγία για, την, ε, για, την, για τη διακριτική μεταχείριση ή έχουμε τη σύμβαση. Προς το παρόν και οι δύο έχουν μπλοκαριστεί. Και αυτό φυσικά είναι κάκιστο για τα άτομα με αναπηρία. Γιατί οποιαδήποτε στιγμή μπορεί κανεί να πάθει κάτι. Ένα ανάπηρο μπορεί να πάθει πολύ εύκολα ένα ατύχημα. Αν δεν ισχύει τίποτα από νομική πλευρά, ούτε η οδηγία είτε, ούτε η σύμβαση του ΟΗΕ, δεν μπορεί να προστατευτεί με κανέναν τρόπο. Ο πρόεδρο του IDF είπε ότι δεν μπορεί να περιμένει το μέλλον. Και εγώ πραγματικά θα, το, θα ήθελα να το επαναλάβω αυτό και προ την Κομισιόν Εντάξει, υπάρχει η οικονομική κρίση η οποία όμως ε, τώρα ε, χτυπά τους πάντες και κυρίως τους ανθρώπους με αναπηρία. Η Γερμανία λοιπόν έχει ζητήσει να συμπεριληφθούν όλες αυτές οι ε, διατάξεις σε νομοθεσία. Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλα δύο ή τρία χρόνια για να γίνει αυτό. Τώρα, να περάσω στην επόμενη αναφορά από το 2008, τη 1402 Αυτό που ε, γράφω είναι κάτι που συμβαίνει σε μένα. Μπορώ λοιπόν να σας το περιγράψω επακριβώς. Όταν δηλαδή κάποιος έχει ζήσει το πρόβλημα. Αυτό είναι που σας έλεγα πιο πριν. Όταν κάποιος έχει ζήσει το πρόβλημα μπορεί να το επεξεργαστεί και διαφορετικά. Γι' αυτό είναι σημαντικό να υπάρξουν, να υπάρξουν ανάπηρα, να μπορούν να συμπληρωθούν ανάπηρα άτομα και στην Κομισιόν. Δεν αρκεί να υπάρχουν μόνο στο Κοινοβούλιο. Γιατί πραγματικά την χάνουν σημαντική διακριτική μεταχείριση. Δεν λαμβάνονται καθόλου υπόψη τα δικαιώματα των αναπήρων. Για παράδειγμα, μετά από, τις, ε, μετά από ατυχήματα. Δεν ε, λαμβάνονται καθόλου υπόψη τα δικαιώματά τους. Επίσης, ε, προστασία στον τομέα της απασχόλησης. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει διακριτική μεταχείριση και δεν, δεν ισχύει τίποτα, ας πούμε, για τους ανάπηρους σε ό,τι αφορά το εργατικό δίκαιο. Γι' αυτό προτείνω να επεκταθούν οι διατάξεις και σε αυτή την οδηγία για την μετακίνηση των πολιτών. Γιατί όταν έγινε, ας πούμε, όταν έκανα εγώ την δική μου τη σύμβαση με την ασφάλεια, όλοι οι γιατροί θεώρησαν ότι το πρόβλημα που είχα εγώ τότε με το λαιμό μου είχε να κάνει με την αναπηρία μου και όχι με το ατύχημα που έπαθα. Οπότε τότε η σύγκριση φυσικά δεν ήταν υπέρ μου, και μετά από 8 χρόνια, όταν τελικά λύθηκε το πρόβλημά μου, το 96 ξεκίνησε η ιστορία αυτή και το 2004 διαπιστώθηκε ότι τελικά αυτό το πρόβλημα στην σπονδυλική μου στήλη ήταν ε, πρόβλημα που προέκυψε από το ατύχημα και τότε μου έδωσαν την κατάλληλη θεραπεία και δεν ήταν θέμα της αναπηρίας μου. Αλλά στην αρχή δεν είχε ληφθεί καθόλου αυτό υπόψη. Οπότε η αποζημίωση που, που, με βάση την αναπηρία μου που υπήρχε πριν από το ατύχημα ήταν πολύ πιο μικρή από το αν δεν ήμουν ανάπηρος όταν πάθαινα το ατύχημα. Γιατί τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στη σπονδυλική μου στήλη δεν λήφθηκαν υπόψη, δεν ε, θεωρήθηκαν ε, ε, συνέπειες του ατυχήματος. Γι' αυτό λοιπόν προτείνω να υπάρξει μία ε, ρύθμιση που να λέει ότι αν ακόμη και εκ των υστέρων προκύψει ότι κάποιος σε μία σύμβαση έχει τύχη διακριτικής μεταχείρισης, τότε είτε θα πρέπει να ακυρωθεί η σύμβαση, είτε θα πρέπει να επαναδιαπραγματευτεί. Ώστε να έχει τις ίδιες ευκαιρίες, να έχει την, ίδια, να έχει την δυνατότητα να λάβει την ε, αποζημίωση που θα ελάμβανε εάν δεν ήταν ανάπηρος πριν από το ατύχημα που του συνέβη. Εγώ μίλησα με την ασφαλιστική εταιρεία. Α, μου είπανε, εντάξει τώρα αυτό που λες, λίγο μας νοιάζει έγινε η σύμβαση, τελείωσε, δεν, έχω, δεν ε, ξαναδιαπραγματευόμαστε, τελειώσαμε. Πρέπει όμως ε, να υπάρξει κάτι, γιατί όπως βλέπετε συμβαίνουν αυτά τα πράγματα και πρέπει να υπάρχει μια νομική βάση που να μας προστατεύει. Αυτά. Αυτά είναι τα προβλήματα που έχουμε εμείς, τα ειδικά σε ό,τι αφορά τις αναπηρίες. Ε, εν τω μεταξύ βλέπατε όσο μιλούσα εγώ και τις διαφάνειες στο PowerPoint. Αν θέλετε τώρα να μπω σε λεπτομέρειες για την κάθε διαφάνεια, ευχαριστώ αλλά δεν νομίζω ότι έχουμε τόσο πολύ χρόνο. Οπότε μπορούμε να περάσουμε και στο επόμενο θέμα. Να μην σας φάω εγώ όλο το χρόνο. alla ναι, Για την 8 είναι αρμοδιότητα άλλης ε, υπηρεσίας της Επιτροπής. Άρα λοιπόν πρώτα να απαντήσει η Επιτροπή, ο αρμόδιος της Επιτροπής για το σημείο 7 και μετά θα πάμε στο σημείο 8. Στέφαν Όλσον από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και να ευχαριστήσω όλους ιδιαίτερως τον αναφέροντα με τον οποίο εργαζόμαστε εκ του συνήγης και τον οποίο γνωρίζω πλέον ε, προσωπικά. Θεωρώ ότι μας δίδαξε πάρα πολλά πράγματα και ότι η ιστορία του είναι ιδιαίτερα δυσάρεστη. Είμαστε αν μη τι άλλο ευγνώμονες για τα όσα μας δίδαξε, για όλες τις πληροφορίες που μας έδωσε. Όσον αφορά την νομική κατάσταση, το νομικό καθεστώς, η αναφορά αυτή καταδεικνύει πόσο σημαντική είναι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πρόταση που ε, υποστηρίχτηκε από το EDF και από τους πολίτες μέσω των υπογραφών τους και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδίως από συγκεκριμένου ευρωβουλευτές που ανέλαβαν πολύ ενεργή δράση. Η ε, πρόταση αυτή που συζητηθήκε στο σημείο 5 έχει να κάνει με την διακριτική μεταχείριση σε όλες τις ε, πτυχές κοινωνίας πέρα από την απασχόληση. Δηλαδή έχουμε την υγεία, την ε, κοινωνική ασφάλιση, την πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες όπως ασφαλίσεις. Σε όλους αυτούς τους τομείς θα υπάρξει απαγόρευση της διακριτικής μεταχείρισης λόγω αναπηρίας, λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού λόγω γύρατος και επιπλέον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβάλλει συγκεκριμένες ρυθμίσεις όσον αφορά την πρόσβαση, την ισότιμη πρόσβαση στις κοινωνικές υπηρεσίες. Θεωρώ λοιπόν ότι ε, η πρόταση αυτή θα πρέπει να εγκριθεί με την ε, μορφή που έχει υποβληθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εφόσον εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα απαντήσει σε πάρα πολλέ από τι ανησυχίε του αναφέροντο και σε πάρα πολλέ από τι ανησυχίε που έχουν και πολλοί άλλοι Ευρωπαίοι πολίτε, είμαι σίγουρο. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρώτο σημαντικό σημείο και θεωρώ ότι εδώ έχουμε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα και θα ήθελα να επιστήσω την ε, προσοχή της Επιτροπής Αναφορών στο εξή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντα μπορεί να κάνει περισσότερα πράγματα, αυτό είναι σίγουρο και εμείς θα προσπαθούμε πάντα να κάνουμε όσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα. Θα πρέπει όμως να συνειδητοποιήσουμε ότι είναι το Συμβούλιο αυτό το οποίο μπλοκάρει την πρόταση αυτή. Κατά τη διάρκεια τεσσάρων προεδριών του Συμβουλίου προσπαθούμε να συζητήσουμε το ζήτημα αυτό και δεν έχουμε καταφέρει να φτάσουμε την απαιτούμενη ομοφωνία ακόμα. Είναι πολύ σημαντικό να συνεργαστούμε λοιπόν με το Συμβούλιο. Πρέπει να πω ότι ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη συνεργάζεται πάρα πολύ καλά με το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τις Αναπηρίες και προσπαθούμε με τη βοήθεια του φόρουμ αυτού να πείσουμε τα κράτη-μέλη ότι πρέπει από κοινωνικής και οικονομικής πλευράς να βοηθήσουν τα άτομα με αναπηρίες. Γιατί τα άτομα με αναπηρίες, τα εκατομμύρια των ανθρώπων αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πέρα από πολίτε και καταναλωτέ και μπορούν να συμβάλλουν και αυτοί στην οικονομική ανάπτυξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε όλοι μαζί και θεωρώ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τόσο μέσω τη Επιτροπή Αναφορών όσο και μέσω τη Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, στην οποία αναφέρθηκε πριν από λίγο ο κύριο Κάσμαν, θα καταφέρουν να ασκήσουν πίεση στο Συμβούλιο. Αυτό όσον αφορά την πολιτική πλευρά, γιατί τέτοισαν κάποια τέτοια ερωτήματα που βρισκόμαστε από πολιτική πλευρά. Δυστυχώ δεν έχουμε ακόμα στο Συμβούλιο την απαιτούμενη ομοφωνία. Ερχόμενος τώρα πάλι στο ζήτημα του α, αναφέροντος. Δυστυχώς βάσει του κοινοτικού και εκτιμένου αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Αυτό το οποίο κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ακριβώς επειδή γνωρίζουμε το μέσο των ασφαλιών να ασφαλίσουν συγχωρείτε, ένα πολύ σημαντικό τομέα. Έχουμε ξεκινήσει ήδη ένα διάλογο με τον κλάδο των ασφαλίσεων και με όλου του ενδιαφερομένου. Συμμετέχει στο διάλογο αυτό και το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τι Αναπηρίε και στο διάλογο αυτό έχει συμβάλει πολύ με την εμπειρογνωμοσύνη του και ο αναφέρον. Προσπαθούμε εδώ πέρα να εντοπίσουμε τι πρακτικέ από το ένα κράτο μέλο στο άλλο. Και αυτό γιατί θεωρούμε ότι υπάρχουν κάποιε εταιρείε οι οποίε προσπαθούν να αποφύγουν να ασχοληθούν με τα ζητήματα αυτά που άπτονται της ναπηρίας. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να εστιαστούμε στις χώρες εκείνες και στις εταιρείε εκείνες που έχουν ασχοληθεί με τα ζητήματα αυτά και να χρησιμοποιήσουμε εθελουσίως αυτές τις βέλτιστες πρακτικές. Δηλαδή, παράλληλα με την οδηγία που έχουμε, να προσπαθήσουμε να πείσουμε τον κλάδο των ασφαλιστικών εταιριών να καταρρύψουν τα εμπόδια που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και όπου υπάρχουν για τα άτομα με αναπηρίες και γενικότερα για τους υπόλοιπους ενδιαφερομένους. Σας ευχαριστώ πολύ την προσοχή σας. Εμείς ευχαριστούμε κύριε Όλσον. Ο, η κυρία Γκόντς. Ε, Θέλετε να πάρετε το λόγο? Όχι. Ο κύριος Κάσμαν, ε, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Βασίλη, συγχαρητήρια για το καταπληκτικό έργο που έχεις κάνει. Πρέπει να πω βέβαια ότι μερικές φορές και εγώ ίδιος ε, δεν μπορώ να καταλάβω πολύ καλά πώς λειτουργούν όλα αυτά. Αστικό δίκαιο, ενοχικό δίκαιο, ανάλυση κινδύνου. Υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντε του οποίου πρέπει να λάβει κανεί υπόψη. Μόλον ότι δεν μπορώ να καταλάβω όλα αυτά πάρα πολύ καλά, καταλαβαίνω πότε πραγματικά υπάρχει αδικία. Βλέπουμε ότι η συζήτηση τη οδηγία έχει μπλοκαριστεί στο Συμβούλιο. Μα αν προχωρούσε στο Συμβούλιο η οδηγία αυτή, θα έχει επιλύσει πάρα πολλά από τα προβλήματα που ακούμε αυτή τη στιγμή. Και κυρία Πρόεδρε, ίσω ένα τρόπο να συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση στο Συμβούλιο, γιατί ξέρετε ότι στην ε, πολιτική χωρί πίεση τίποτα δεν γίνεται, ένας τρόπος λοιπόν θα ήταν να δούμε αν μπορούμε να υποβάλουμε μια προφορική ερώτηση στο Συμβούλιο. Δεδομένου του πολύ μεγάλου αριθμού αναφορών που λαμβάνουμε για το πρώην άρθρο 13 νυν άρθρο 19 για ζητήματα που έχουν να κάνουν με την θρησκεία, τις πεπιθήσεις, το σεξουαλικό προσανατολισμό, τα οφείλω και τις συναπηρίες Να υποβάλουμε σχετικά λοιπόν μια προφορική ερώτηση στο Συμβούλιο κατά τη διάρκεια της Συνόδου Λομελίας. Πρέπει να σας πω ότι πριν από αρκετά χρόνια, όταν ήμουν ηθοποιός, την εποχή εκείνη δεν ασφαλίζανε τους ηθοποιούς, γιατί μας θεωρούσαν τότε απατεώνες, κλέφτες. Βλέπω ότι μερικοί ακόμα συμφωνούν με αυτό το επιχείρημα. Και όταν άλλαξε η αντίληψή τους, τότε βρήκαν ένα άλλο επιχείρημα. Μας είπανε, αν είστε διάσημος, και αν παίζετε σε κάποιο θέατρο ή σε κάποιο έργο εκτός της χώρας σας, πάλι δεν μπορούμε να σας καλύψουμε γιατί ο κίνδυνος είναι πάρα πολύ μεγάλος. Και μετά από πολλή πίεση συνειδητοποίησαν ότι έχουν να κερδίσουν πάρα πολλά ασφαλή των ηθοποιούς. Και τώρα βέβαια τρέχουν να μας ασφαλίσουν. Ενδεχομένως αυτό να πρέπει να δούμε και σε κάποιες άλλες χώρες για το ζήτημα αυτό. Ιδίως να εντοπίζουμε αυτή την τόσο μεγάλη ανισότητα και αδικία. Στην Αυστραλία, για παράδειγμα, αν έχει κανεί ένα αυτοκίνητο, αυτόματα το αυτοκίνητο αυτό πρέπει να φορολογηθεί. Και με το αυτοκίνητο αυτό καταφέρνει κανεί να έχει μια ασφάλιση απέναντι σε τρίτον. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ο ιδιοκτήτη ενό αυτοκινήτου αναγκαστικά και αυτόματα είναι ασφαλισμένο για ζημία που μπορεί να προκαλέσει σε τρίτο. Ενδεχομένω και σε ορισμένα κράτη-μέλη θα μπορούσαμε αυτόματα να παρέχουμε μια τέτοια κάλυψη, μια τέτοια ασφάλιση. Αναφερθήκαμε νομίζω και σε μια μελέτη που έλαβε χώρα. Ας δούμε ποιε είναι οι πρακτικές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στα διάφορα κράτη-μέλη. Ας τι μελετήσουμε, αλλά δεν χρειάζεται να επινοήσουμε από την αρχή τον τροχό. Έχουμε ήδη στο Συμβούλιο αυτή την οδηγία πλαίσιο, Α ασκήσουμε πίεση στο Συμβούλιο προκειμένου να αναλάβει δράση. Και ας κρατήσουμε ουσιαστικά το Συμβούλιο υπόλογο για την απουσία αυτή δράσης. Ευχαριστώ. Ε, ναι, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Με όσα είπε ο φίλος Κάσμαν, συμφωνώ και εγώ, καλόδεχτα τα λόγια του αλλά με ανησυχούν τα λόγια της Επιτροπής γιατί το Συμβούλιο παγώνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια αυτό το θέμα πώς θα γίνει να βρούμε μια λύση και ε, ε, έχει το πράσινο φως η Επιτροπή γι' αυτό και η πρόταση του Μάικελ χρειάζεται μια επιστολή από εδώ στην ρεύοντα του Συμβουλίου για να ξεπαγώσει, να ξελιμνάσει αυτή η κατάσταση και ε, όπως είπε και ο Μάικελ Αυτές οι ερωτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο Συμβούλιο και να δούμε μέσω των δύο αυτών δών πώς θα έχει η κατάσταση, πώς θα ξεπαγώσει η κατάσταση από το Συμβούλιο που το εξήγησε και ο αναφέρον ε, πώς έχουν τα πράγματα και την χάνει υποστήριξής μας. Κυρία Ράπτη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είναι πάρα πολύ ξεκούραστο να μιλάει κανείς μετά τον κύριο Κάσμαν. Γιατί δεν μένει τίποτα να πει και έτσι μιλάει πάρα πολύ λίγο. Ε, θέλω λοιπόν να πω και κάτι ακόμη. Ο κύριος Κάσμαν είπε ότι είναι ηθοποιός και μας έδωσε μερικά παραδείγματα από αυτά που συμβαίνουν στο χώρο του. Ε, το δικό μου επάγγελμα πριν γίνω εθνική βουλευτής και τώρα ευρωβουλευτής ήταν δημοσιογράφος. Ως δημοσιογράφος λοιπόν θέλω να βλέπω τα πράγματα πρακτικά, να έχουμε αποτελέσματα. Έτσι λοιπόν, με δύο κουβέντες. Με βάση αυτά που είπε ο α, συνάδελφος κ. Κάσμαν και η προβληματική του αντιπροέδρου μας, θέλω δε σε αυτά να προσθέσω το τελευταίο κομμάτι που βλέπω και γραμμένο εδώ ως συμπέρασμα, αλλά και την επιχειρηματολογία στο πρώτο σκέλος του εκπροσώπου της Επιτροπής, θεωρώ αυτονόητο, για να αφήνω τα λόγια και να περνάω στην πράξη, ότι αυτή η αναφορά πρέπει να μείνει ανοιχτή, με την ελπίδα ότι θα βγει από την κατάψυξη του Συμβουλίου η υπόθεση της οδηγίας. Τελεία. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ράπτη και για μένα ήταν πολύ εύκολο να πάω σας παρακολουθήσω λόγω της γλώσσας βέβαια. Πού είναι? Α, there you are. Mr. Kasman Hadjio. Yeah. Uh, Michael. Yes. Just, just um, if we are... Λοιπόν, αν τίθεται όντω το ερώτημα αυτό προς το Συμβούλιο, όπως το είπε, το είπε ο κύριος Κάσμαν. Θα ήθελα να πω το και στην δική μου τη χώρα έχουμε πλέον μία ρύθμιση που επιτρέπει στις ε, ασφαλιστικές εταιρείες, επιτρέπει τόσο αγωγικών βέβαια, να κάνουν διακρίσεις εις βάρος των γυναικών, επειδή οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες, έτσι υπολόγισαν. Και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Ξέρω βέβαια ότι το ζήτημα της αναπηρίας είναι πάρα πολύ σημαντικό και σαφώς πολύ πιο πολύπλοκο. Αν τεθεί όμω το ζήτημα αυτό στο, στο Συμβούλιο, με συγχωρείτε, ότι να θέσουμε και το ζήτημα αυτό του φίλου, των γυναικών δηλαδή. Ευχαριστώ. Thank you, Chairman. Uh, I just wanted to... Ευχαριστώ να διαβεβαιώσω την Τατιάνα ότι εγώ είμαι απόλυτα δεσμευμένο στην ισότητα των δύο φίλων. Ο μόνος λόγος για τον οποίο δεν το ανέφερα ήταν ότι σε σχέση με το θέμα αυτό το φίλο δεν είναι κομμάτι του άρθρου 13, τώρα άρθρου 19. Καλύπτεται αλλού στη συνθήκη. Η δυνατότητα για την Ένωση δηλαδή να αναλάβει δράση για να αντιμετωπίσει τη διεκτική μεταχείριση με βάση το φύλλο. Φυσικά πρέπει να αναθεωρήσουμε τα όσα γίνονται, γιατί μία από τις οδηγίες για το φύλλο ε, θα έρθει πάλι στο Κοινοβούλιο για ε, μελέτη, οπότε ίσως τότε θα ήταν η καλή ευκαιρία να ξαναδούμε το θέμα της ισότητας και των ανισοτήτων που εξακολουθούν να υπάρχουν. Οι γυναίκες είναι πλειοψηφία έτσι, μην το ξεχνάτε αυτό. Κύριε, ευχαριστώ κύριε Κάσμα. <clears throat> Κύριε Σαλαβράκη, παρακαλώ. Εάν θέλουμε να συζητήσουμε, κυρία Πρόεδρε, στη βάση μιας λέσχης κοινωνικού προβληματισμού, όλοι φαντάζομαι βλέπουμε το πρόβλημα των αναπήρων με μεγάλη συμπάθεια. Το θέμα είναι να κάνουμε το επόμενο βήμα. Και το επόμενο βήμα είναι αυτό που έρχεται από την απάντηση της Επιτροπής. Ήδη έχει καθυστερήσει η λήψη του νομικού πλαισίου που θα μας οδηγήσει στις πράξεις εκείνες που θα κατογυρώσουν τα δικαιώματα που όλοι τα αναγνωρίζουμε. Και δεν μπορούμε να μην αναγνωρίσουμε δικαιώματα στο 12% του πληθυσμού. Είναι, ε, άκουσα μια στατιστική προηγούμενα που ήταν ε, όχι 50, 65 εκατομμύρια, είναι 12,5 εκατομμύρια δηλαδή του πληθυσμού. Δεν μπορούμε να πούμε πλέον ότι είναι, αποτελούν μειονότητα. Είναι μείζον πρόβλημα και είναι πρόβλημα μείζον διότι είναι και έκτακτον. Δηλαδή οφείλεται και σε έκτακτα περιστατικά η δημιουργία μιας αναπηρίας που μπορούν όπως ελέγχθη προηγουμένως να πλήξουν τον καθένα από εμά την επόμενη στιγμή, την επόμενη ώρα. Συνεπώς, εάν μείνουμε στο να εκφράσουμε τη συμπαθιά μας στους ανθρώπους που έχουν αναπηρία και έρχονται μπροστά μας με την αναφορά του συγκεκριμένου σημείου της αναπηρίας του δεν έχουμε κάνει τίποτα. Έχουμε μείνει στον καλό λόγο και ο καλός λόγος και η λύση του προβλήματος δεν γίνεται με equity όπως λένε οι Εγγλέζοι. Γίνεται με απόφαση. Θα έλεγα λοιπόν το εξή. Είτε μια απόφαση της Επιτροπής στην Ολομελιά της, είτε με ένα έγγραφο του Προεδρείου προς την Κομισιόν, εν μάλιστα και με τη λειτουργία της Επιτροπής μετά τη συνθήκη της, ε, ε, την οποία τώρα υπηρετούμε και τις αποφασιστικότερες σημασίες της στη διαρρύθμιση των αποφάσεων που θα ζητήσει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα από την Επιτροπή και, θα, και να το επιβάλλουμε αυτό και με ψηφίσματα και στην Ολομέλεια με χρονοδιαγράμματα. Δεν είναι δυνατόν να τους πηγαίνουμε και να τους φέρουμε τους ανθρώπους, να τους λέμε έχουμε ανοιχτή την αναφορά. Βλέπω η μία είναι το 2006, μπορεί να φτάσει το 2016 και να μην δίνουμε λύση στο πρόβλημα. Διότι το πρόβλημα συνδέεται και με οικονομική επιβάρυνση. Δεν μπορούμε να λέμε ότι θα επιβάλλουμε σε ασφαλιστικές εταιρείες κάτι ή να το εκφράζουμε σαν ευχή, διότι είναι εμπορικέ εταιρείε, βασίζονται στην αρχή τη ανταποδοτικότητα και αν δεν του ενισχύσουμε οικονομικά με, συγκεκριμένη, ε, με συγκεκριμένο επιμίσθιο, με συγκεκριμένο ασφάλιστρο για του ανθρώπου με ειδικέ ανάγκε, δεν θα το κάνουν ποτέ. Πολύ δε περισσότερο όταν τα πρόσωπα με αναπηρία δεν έχουν και τη δύναμη σαν κοινωνική ομάδα να επιβάλλουν ορισμένε καταστάσει. Θα έλεγα λοιπόν το εξή. Αφενό με να μείνει ανοιχτή η αναφορά, δεν περί αυτού Φαντάζομαι ότι όλοι μας συμφωνούμε. Αφετέρου όμως να λάβουμε μέτρα ουσιαστικότερου χαρακτήρα και να προχωρήσει είτε το Προεδρείο είτε η Επιτροπή σε διαβήματα προς τον Κομισιόν για να έχουμε επιτάχυνση αυτής της διαδικασίας της λύσεως του θέματος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, θέλετε κάτι να πείτε κύριε Κατσιούλη. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομα. Εγώ πήγα μέχρι το δικαστήριο στη χώρα μου, για τη δική μου την περίπτωση δηλαδή, και το δικαστήριο έκρινε ότι αυτό το θέμα μπορεί να ρυθμιστεί νομικά. Και τώρα προσπαθούν να βρούνε κάποιες νομικές δυνατότητες. Βέβαια το θέμα δεν είναι να το λύσουμε το θέμα πολιτικά μόνο, αλλά και νομικά. Ε, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πρέπει, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μάλλον, θα πρέπει να μας πει πώς μπορούμε εμείς να εξασφαλιστούμε από του κινδύνου που διατρέχουμε ως ανάπηροι. Εγώ δεν είμαι εξασφαλισμένο, δεν, ε, ε, σε σχέση με τους κινδύνου που διατρέχω, ενώ οι υπόλοιποι άνθρωποι που δεν είναι ανάπηροι είναι. Ε, να κλείσουμε την... Κρατάμε ανοιχτή την υπόθεση, δεν υπάρχει καμία, την αναφορά, δεν υπάρχει καμία ε, αμφιβολία περί αυτού ε, θεωρώ του κυρίου Κάσμαν η πρόταση για την προφορική ερώτηση και σας παρακαλώ να την, να κάνετε στην επόμενη Ολομέλεια, ε, κύριε Κάσμαν. Ε, και βεβαίως μια επιστολή προς το Συμβούλιο θα μπορούσε επίσης να γίνει, γιατί μοιάζει όλες αυτές οι τρεις υποθέσεις που ακούσαμε τώρα να κλειδώνουν ένα τεράστιο ζήτημα. Ότι εμείς εδώ, ανεξάρτητα από το αν ανήκουμε στην Επιτροπή Αναφορών, είμαστε μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έχουμε υποχρέωση να πιέσουμε το Συμβούλιο, την Επιτροπή να προχωρήσει σε τέτοια ζητήματα που εκπροσωπούν, που, με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωπα ένα μεγάλο μέρος αυτής της κοινωνίας που ονομάζουμε Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Θεωρώ μάλιστα ότι ίσως θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό αν στην ε, πρώτη αναφορά, όπου έχουμε ήδη μαζεμένες 1.250.000 ε, περίπου υπογραφές να δούμε στην ουσία την πρώτη ευκαιρία μας ως Ευρωκοινοβούλιο να ε, έχουμε τη δύναμη να την παρουσιάσουμε ως πρωτοβουλία πολιτών και να την αξιοποιήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Θεωρώ λοιπόν ότι ήρθε η στιγμή να πιέσουμε προς μια κοινωνικότερη Ευρώπη και χαίρομαι ότι ανήκω σε αυτή την Επιτροπή γιατί ίσως είναι από τις λίγες που θα μπορούσαν να πιέσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ. Ε, επειδή ο χρόνος είναι τρέχει πολύ δημοσιογραφικά κυρία Ράπτη. Ε, έχουμε την επόμενη ε, αναφορά πάλι από τον κύριο Κατσούλη που στην ουσία ε, θα έχει προβολή μιας μικρής ταινίας και αφορά ένα παρόμοιο ζήτημα, όχι ακριβώς το ίδιο. Κύριε Κατσούλη. Μιλούμε για την συμπερίληψη των ατόμων με αναπηρία στα σχολεία τα, των παιδιών με αναπηρία. Ε, το ίδιο πρόβλημα είναι θεωρητικά. Άνθρωποι με αναπηρία δεν έχουν καμία πρόσβαση σε υπηρεσίε, σε σχολεία. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει πάντα. Μιλούμε για αποκλεισμό. Το πρόβλημα αυτό αφορά το δικό μου το γιο, ο οποίος ε, είναι αυτιστικός. Από τον Οκτώβριο του 2008 έχω έρθει εδώ, στο Κοινοβούλιο και το είδα ότι στο Ευρωπαϊκό Σχολείο εδώ στις Βρυξέλλες συμβαίνουν σημεία και τέρατα. Μιλώ λοιπόν για τη συμπερίληψη των παιδιών με αναπηρία στα σχολεία. Είναι λίγο διαφορετικό αυτό από την ενσωμάτωση. Η συμπερίληψη, η ένταξη ε, ρυθμίζεται στο άρθρο 24 της Σύμβασης του ΟΗΕ. Εγγυάται, ε, εξασφαλίζεται συγγνώμη, εκεί η πλήρη κοινωνική συμμετοχή. Μιλούμε δηλαδή για κοινωνική συμμετοχή. Δεν μιλούμε για το ότι ο δικό μου γιο θα πάει σε μια τάξη ενό κανονικού σχολείου. Είναι να μπορεί να πάει σε ένα σχολείο το οποίο μπορεί να του προσφέρει όσα χρειάζεται και σε αυτόν και στα παιδιά τα υπόλοιπα, δημιουργώντας μια πιο κοινωνική, πιο κοινωνική κοινωνία, αν μπορώ να το πω έτσι. Ε, ο γιο μου πάει στο σχολείο αυτό λοιπόν, έχει ε, τους φίλους του και μια μέρα του είπαν ότι δεν μπορεί να πηγαίνει στο σχολείο πια, ε, έχασε τους φίλους του, καταλαβαίνετε τι, πόσο σημαντικό είναι αυτό για ένα μικρό παιδί. Υπήρξε και ένα ε, ντοκιμαντέρ στη γερμανική τηλεόραση για την περίπτωση αυτή και είδαμε πόσο σημαντικό είναι αυτό, πόσο σημαντική είναι η ένταξη γιατί η έννοια αυτή της ένταξης ε, είναι, είναι νέα και δεν πρέπει να τη συγχαίουμε με την ενσωμάτωση. Και αναφέρεται ότι κανένα παιδί και στην Σύμβαση ΙΕ δεν μπορεί να αποκλείεται από ένα σχολείο. Δηλαδή το σχολείο πρέπει να κάνει οτιδήποτε και μάλιστα στην Ισπανία υπάρχει ένα πολύ καλό παράδειγμα για το πώς λειτουργούν τα σχολεία. Υπάρχει μεγάλο ποσοστό ατόμων, παιδιών με αναπηρία που πάνε σχολείο στην Ισπανία και στην Ιταλία και στη Γερμανία έχουμε την το μεγαλύτερο διαχωρισμό. Δηλαδή ε, το 78% των παιδιών δεν πάνε σε ένα κανονικό σχολείο. Ε, στην, Ισπανία, στην Ισπανία και την Ιταλία συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Γιατί δηλαδή κάτι μπορεί να λειτουργήσει στην Ισπανία και την Ιταλία και δεν μπορεί να λειτουργήσει στη Γερμανία. Οπότε τώρα έχουμε τη σύμβαση για τα άτομα με αναπηρία που λέει σαφώ και μας δίνει το ε, δικαίωμα τα παιδιά μας, αν είναι παιδιά με αναπηρία, να μπορούν να πάνε σε ένα σχολείο που πάνε όλα τα παιδιά, να εντάσσονται κοινωνικά σε ένα σχολείο. Γιατί αν πάνε σε ένα ειδικό σχολείο, αυτά τα ειδικά σχολεία συνήθω είναι κάπου μακριά, πρέπει δηλαδή να κάνει κανεί ταξίδι 100 χιλιόμετρα να, βρει το σχολείο, χωρίζονται οικογένειε. Καταλαβαίνετε. Ο γιος μου μιλάει μόνο γερμανικά, οπότε μπορούσε να πάει μόνο στο ευρωπαϊκό σχολείο. Εγώ καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας είμαι χωριστά από τη γυναίκα μου είναι εδώ η γυναίκα μου σήμερα με την κόρη μου. Ε, Εμεί, εν πάση περιπτώσει, βρήκαμε μία, μία λύση. Γιατί ο γιο μου μιλάει μόνο γερμανικά. Οπότε, επειδή είμαστε και στην. μπορούσαμε να, πάμε, να πάει σε ένα σχολείο που βρίσκεται στα σύνορα με την Γερμανία. Τώρα, αν, ο γιος μου, αν το γιο μου τον είχα μεγαλώσει εγώ να μιλάει ελληνικά, τότε θα έπρεπε να ακυρώσω τη σύμβασή μου με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, γιατί ο γιο μου έχει, είναι παιδί με αναπηρία. Και η Κομισιόν μου λέει πράγματα που δεν ισχύουν, δεν λαμβάνει υπόψη της τις, τις συνθήκες που επικρατούν στις ζωές των ανθρώπων αυτών. Γιατί συγχαίει την ένταξη με την ενσωμάτωση. Η ένταξη είναι τελείως διαφορετική από την ενσωμάτωση. Ναι. Θα προβάλλουμε και το φιλμ γιατί δεν έχουμε πολύ ώρα. Ναι, ναι ε, τελειώνω Τελειώνω ε, Και πολύ σύντομα να προσθέσω ότι με τον αποκλεισμό αυτό και με τα σχολεία που δεν είναι προσαρμοσμένα, φυσικά δημιουργούνται περαιτέρω κόστη, η Κομισιόν αρνείται να καλύψει το κόστος, το δικό μου, δηλαδή εγώ έρχομαι εδώ για να δουλέψω και πραγματικά αντιμετωπίζω ένα τεράστιο στρες να είμαι, στο σχολείο, να είμαι στη δουλειά μου και να, έχω, να σκεφτώ μονίμως τι θα γίνει ο γιος μου στο σχολείο, αν θα τον διώξουν ή δεν θα τον διώξουν. Και η Κομισιόν έτσι μου το παίζει άνετη και λέει άμα τα έχουμε ρυθμίσει αυτά τα θέματα. Τίποτα δεν έχει ρυθμίσει. Ε, πραγματικά εκνευρίζομαι και συγγνώμη που εκνευρίζομαι, αλλά δεν γίνεται να συνεχιστεί άλλη αυτή η κατάσταση. Και αν θέλετε τώρα μπορούμε να δούμε και το φιλμ.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 ε, συμμερίζομαι τις απόψεις του κ. Κατσούλη, αλλά θα παρακαλούσα να μην ανοιχτή η αναφορά και να επανέλθει συνοδευομένη από μια έκθεση παιδοψυχιάτρου, εάν και κατά πόσον ε, το σχολικό περιβάλλον είναι κατάλληλο για το παιδί ή όχι, διότι όπως ξέρετε η παιδική ε, εγκληματικότητα έχει αυξηθεί, έχουμε φτάσει σε σημεία και βαρβαρότητος, έχουμε προβλήματα πάρα πολλά και πρέπει να δούμε αν το συγκεκριμένο σχολείο από πλευρά παιδοψυχιατρική είναι κατάλληλο για το παιδί για να το ενισχύσουμε ή όχι. Το αίτημα ή όχι. Ευχαριστούμε. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Ναι. Ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε. Η οχι το αιτημα η οχι ευχαριστουμε κυρια προεδρε σα Μπαρντού. Μέχρι. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Ε, είναι πολύ σημαντικό λεπτό το πρόβλημα αυτό που μας λέει ο αναφέρον ε, και αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή η Επιτροπή Ευρωπαϊκή και υποσχεθήκαμε την ένταξη παιδιών με προβλήματα στο Ευρωπαϊκό Σχολείο και εμείς επιμείναμε όλα αυτά τα χρόνια τα τελευταία ώστε να υπάρξουν τα απαραίτητα μέσα όταν ακριβώς υπάρχουν παιδιά με ιδιαίτερα προβλήματα που θα πρέπει να ενταχθούν στα Ευρωπαϊκό Σχολείο. Αυτό που είπε ο κύριος Κατσιούλη, ε, εκεί ε, απέδωσε ιδιαίτερη σημασία στα λόγια του κύριου Ματσιούλη και όσα μας είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είχαμε πολλέ ε, συναντήσεις, επαφές, η Επιτροπή γνωρίζει το πρόβλημα. Ο κύριος Κατσιούλη επίσης με τον πρόεδρο της Επιτροπής, τον κύριο Κάλλα, συναντήθηκε και η Επιτροπή μπορούμε να πούμε ότι ιδιαίτερα πρόσεξε το πρόβλημά του. Το Ευρωπαϊκό Σχολείο έχει μια πολιτική ένταξη για τα παιδιά ακριβώς που σημαίνει ότι δίδει τα απαραίτητα μέσα για τις ιδιαίτερες ανάγκες ενός μαθητή αλλά ο μαθητής θα πρέπει να μπορεί να συμμετέχει στα κύρια σημεία δραστηριότητες μαθήματα με τα περισσότερα παιδιά της ηλικίας του και είναι πολύ λεπτή αυτή η σημερινή περίπτωση το σχολείο, ανεξάρτητα από τα μέσα που διαθέτει κηρύσσει αυτό αναρμόδιο. Στην περίπτωση αυτή στο Βολιβέ υπήρξαν πολλές προσπάθειες για να ενταχθεί το παιδί αυτό. Δύο άτομα ειδικευμένα, γερμανόφωνα, δόθηκαν στη διάθεση αυτού του παιδιού για να το συντροφεύουν, για να το συνοδεύουν. Πήρε σημαντικά μέτρα το σχολείο, αλλά διαπίστωσε μια κάποια στιγμή ότι δεν είχε τις δυνατότητες για να εντάξει αυτό το παιδί και ότι δεν θα μπορούσε να ανταποκριθεί. Και σημαντικό είναι λοιπόν τώρα εδώ να τονίσουμε το τι μπορεί να προσφέρει το Ευρωπαϊκό Σχολείο σε σχέση με αυτό που μπορεί να προσφέρει το σύστημα εκπαίδευσης ενός κράτους μέλους. Σε ένα κράτος μέλος υπάρχουν πολλά πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα που θα μπορούσαν να προταθούν και κλασικής μορφής, ε, ακαδημαϊκής, επαγγελματικής μόρφωσης, ε, τεχνικής παρόμοιας, ε, για καλλιτεχνικά, αθλητικά, και πάρα πολλές δραστηριότητες. Λοιπόν, εκεί ανάμεσα πρέπει να υπάρχει και μια προσφορά για παιδιά που έχουν μια κάποια αναπηρία. Και το Ευρωπαϊκό Σχολείο δεν μοιάζει όμως με να, δεν εντάσσεται όπως πρέπει σε ένα εθνικό πλαίσιο εκπαίδευσης. Είναι κλασικής μορφής εκπαίδευση ακαδημαϊκής που έχει να κάνει και με το τελικό δίπλωμα στην τελευταία τάξη το πολιτήριο. Και αυτό σε όλες τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι σημαίνει αυτό οι μαθητές μερικές φορές δεν μπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους ε, στο ευρωπαϊκό σχολείο. Δεν πρόκειται όμως για διάκριση απέναντι σε παιδιά που έχουν ένα παρόμοιο πρόβλημα. Είναι ότι το παιδί δεν μπορεί να ενταχθεί όπως πρέπει σε ένα παρόμοιο σχολείο. Ένα παιδί ας πούμε που θέλει να, ακούσει, να ακολουθήσει καλλιτεχνική κατεύθυνση είτε να γίνει πρωταθετής κάπου είτε τεχνική εκπαίδευση δεν θα μπορέσει να ενταχθεί όπως πρέπει σε αυτό το σχολείο το ευρωπαϊκό και θα πρέπει να πάει σε άλλο σχολείο. Να σας τονίσουμε λοιπόν κάπως το στενό αυτό να αποκαλέσουμε χαρακτήρα του Ευρωπαϊκού Σχολείου και παρόλο που έχουμε μια εκπαίδευση όλες τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι πρόβλημα, ότι αρκετές φορές θα μπορούσε να κηρύξει αυτόν αρμόδιο ένας, το Ευρωπαϊκό Σχολείο. Στην περίπτωση αυτή η Επιτροπή Ευρωπαϊκή κατέβαλε κάθε την προσπάθεια να βοηθήσει την οικογένεια και η Επιτροπή βρήκε ένα σχολείο στο νότιο Βέλγιο ένα σχολείο ειδικό που μπορεί να δεχτεί ένα παιδί αυτιστικό και αυτά που είπε ο κ. Κατσιούλη σαν προβλήματα σχετικά με το σημεία τα σχετικά. Ήρθαν σε επαφή με τις κοινωνικές υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είναι οργοδότης του κ. Κατσιούλη ώστε να δοθούν όλα τα απαραίτητα μέσα, όλη η απαραίτητη βοήθεια ε, σύμφωνα και με την εργασία του. Και η Επιτροπή κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να προσφέρει βοήθεια, να ενημερώσει, να συνεργαστεί όσο μπορούσε με τις αντίστοιχες υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να βρεθούν οι καλύτεροι δυνατοί τρόποι. Επανέρχομαι στο γενικής φύσεως πρόβλημα. Βέβαια συνεχίζει να βελτιώνει ε, την δυνατότητα πρόσβασης στο Ευρωπαϊκό Σχολείο των παιδιών με προβλήματα ή με αναπηρίες ε, κάθε φορά στη Μεκτή Παιδαγωγική Επιτροπή, στον Ανώτατο Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Σχολείου. Κάθε φορά εμείς εκεί κάνουμε μια ανάλυση, επιμένουμε σε περιπτώσεις παιδιών που δεν μπορούν να παραμείνουν για να εξετάσουμε λοιπόν τι μπορεί να γίνει, τι μπορεί να βελτιωθεί στο σχολείο αυτό αλλά επαναλαμβάνουμε είναι θέμα ένταξης σε ένα γενικό σχολείο ακαδημαϊκής μόρφωσης που δεν μπορεί να προσφέρει βοήθεια σε κάθε ειδική περίπτωση. Γι' αυτό ακριβώς ε, επιμένει η Επιτροπή ε, στην ε, οικογένεια να την εμερώνει, τι μπορεί να προσφέρει το Ευρωπαϊκό Σχολείο και ενδεχόμενα τι δεν μπορεί να προσφέρει. Και ακριβώς όσο γίνεται περισσότερες πληροφορίες για τις δυνατότητες φοιτητήσεις ανάλογα με τις ειδικέ τους επαγγελματικές οικογενειακές ανάγκες. Ευχαριστώ. Κυρία Ράπτη, τώρα που θα μιλήσετε πριν από τον κύριο Κάσμαν, ίσως προλάβετε να πείτε αυτά που δεν θα μπορεί να πει εκείνος. Λοιπόν, ε, κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ και θα σας πω το εξής. Εάν είχα μιλήσει πριν την εκπρόσωπο της Επιτροπής, θα είχα πει μία φράση μόνο. Να μείνει ανοιχτή η αναφορά. Ε, με όλο το σεβασμό που έχω προς την Επιτροπή και προς τους εκπροσώπους της μετά τα όσα άκουσα από την εκπρόσωπο της Επιτροπής, είμαι υποχρεωμένη ε, απέναντι στη συνείδησή μου πρώτα και κύρια ε, να πω μερικά λόγια παραπάνω. Ε, καταρχήν ξεκινάω από το τελευταίο, ότι η Επιτροπή βρήκε ειδικό σχολείο και υπέδειξε στον αναφέροντα για να βάλει το παιδί του. Με συγχωρείτε, αλλά όταν ο αναφέρον έχει τέτοια επιμονή και υπομονή τόσων χρόνων. Έχει κάνει την ταινία που μόλις παρακολουθήσαμε. Έχει δείξει τέτοια επιμέλεια όλα αυτά τα χρόνια στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων του. Δεν είχε ανάγκη την Επιτροπή για να βρει το σωστό σχολείο. Μπορούσε να το κάνει και μόνος του. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, άκουσα να λέμε ότι το ευρωπαϊκό σχολείο, ο χαρακτήρας του ευρωπαϊκού σχολείου, αν σωστά μου μεταφράστηκε είναι στενός. Θεωρώ αδιανόητο το ευρωπαϊκό σχολείο μόνο και μόνο ως ευρωπαϊκό να έχει ένα στενό χαρακτήρα. Το ευρωπαϊκό σχολείο πρέπει να είναι παράδειγμα, πρέπει να είναι πρότυπο, να είναι ανοιχτό, να προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεύτερο κράτο. Τρίτο, άκουσα να γίνεται μία Αντιπαραβολή, μία παρομοίωση τα αθλητικά σχολεία, τα καλλιτεχνικά σχολεία και τα σχολεία για άτομα με ειδικές ανάγκες. Με συγχωρείτε, αλλά ή κάτι εγώ δεν κατάλαβα καλά ή κάτι άλλο συμβαίνει. Συγκρίνουμε ανώμια. Διότι ένα παιδί και στην Ελλάδα, στη χώρα μας, έχουμε αθλητικά σχολεία ένα παιδί που πηγαίνει στο αθλητικό σχολείο πηγαίνει όχι γιατί δεν μπορεί να ενταχθεί στο κανονικό σχολείο, αλλά γιατί θέλει να πάρει μια άλλη κατεύθυνση. Γιατί θέλει να, γίνει, να ακολουθήσει πρωταθλητισμό. Ένα, σχολείο πάει, ε, ένα παιδί πάει στο καλλιτεχνικό σχολείο όχι γιατί δεν μπορεί να ενταχθεί μέσα στο κανονικό σχολείο, αλλά για άλλο συγκεκριμένο λόγο. Έχει ένα ειδικό ταλέντο. Και έρχομαι στο συγκεκριμένο θέμα. Τον κύριο Κατσιούλη δεν τον γνωρίζω. Ούτε πρόκειται να του χαριστώ γιατί είναι Έλληνας. Δεν με αφορά αυτό. Οφείλω να τον αντιμετωπίζω και την αναφορά του όπως αντιμετώπιζα την αναφορά οποιοδήποτε από οποιοδήποτε κράτος. Και, σημειώνω, δεν είμαι βέβαιη, δεν είμαι βέβαιη, είναι δική μου άποψη αυτή, μπορεί να κάνω λάθος, δεν είμαι βέβαιη ότι η επιστροφή του παιδιού στο ευρωπαϊκό σχολείο θα του κάνει καλό. Δεν είμαι βέβαιη, αλλά δεν είμαι ειδική. Όμως, οφείλω να πω ότι από αυτά που διάβασα εδώ, εδώ είναι όλα γραμμένα και μεταφρασμένα σε όλες τις γλώσσες, αυτό που κατάλαβα είναι ότι υπήρχε από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Σχολείου μία, συγχωρήστε μου την έκφραση, ε, άρνηση να δεχτεί να κάνει στο μέγιστο βαθμό αυτό που πραγματικά θα έπρεπε να προσπαθήσει να κάνει. Μιλήσαμε προηγουμένως για αυτά που γράφουμε στα χαρτιά και για αυτά που υποστηρίζουμε στη θεωρία. Αυτά όμως πρέπει να τα κάνουμε πράξη. Η δική μου αίσθηση, και μπορεί να κάνω λάθος, είναι ότι δεν κατεβλήθη προσπάθεια τόση όση έπρεπε. Ένα. Δεύτερον, θα περίμενα να ζητηθεί μία ιατρικού τύπου γνωμάτευση από ειδικού, όχι μόνο εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτικός, παιδοψυχολόγος, γιατρός, μία τριπλέτα δηλαδή αρμοδίων και ειδικών, οι οποίοι να αποφασίσουν ότι ένα παιδί δεν μπορεί να ενταχθεί μέσα σε ένα σχολείο όταν μάλιστα αυτό το σχολείο είναι το Ευρωπαϊκό Σχολείο. Ε, με δεδομένα όλα αυτά και με δεδομένο επίσης ότι όταν συζητούμε εδώ αναφορές δεν συζητούμε μόνο για να ικανοποιήσουμε ή για να μην ικανοποιήσουμε κάποιον που κάνει μια αναφορά αλλά δίνεται η ευκαιρία να θίξουμε και να συζητήσουμε γενικότερα ζητήματα θεωρώ ότι σε κάθε περίπτωση αυτή εδώ η αναφορά πρέπει να παραμείνει όχι ανοιχτή, διάπλατη. Ευχαριστώ. Πολύ κύριε Ράπτη. Ο χρόνος περνάει. Η επόμενη παρακαλώ, ο κύριος Κάσμαν καταρχήν, αν μπορεί να μας μιλήσει λίγο σύντομα. Ευχαριστώ πολύ. Um, θα είμαι πολύ σύντομος. Με ιδιαίτερη χαρά παίρνω το λόγο μετά την κυρία Ράπτη, γιατί είπε τα περισσότερα από αυτά που θα ήθελα να πω. Σε ένα σημείο διαφέρω εγώ. Νομίζω ότι ο Βασίλης έκανε την αφορά αυτή γιατί θέλει να ασχοληθούμε με τις γενικές αρχές, δηλαδή με την διακριτική αυτή μεταχείριση την οποία δεν θέλει να επαναληφθεί. Δεν νομίζω λοιπόν θα πρέπει να μπούμε αυτή τη στιγμή σε συγκεκριμένε λεπτομέρειες. Γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να γίνεται αναφορά σε ψυχολογική ανάλυση κτλ. Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι υπάρχει κοινοτική χρηματοδότηση προς τα ευρωπαϊκά σχολεία. Επομένως τα σχολεία αυτά θα πρέπει να συμμορφώνται με τις θεμελιώδεις αρχές Ευρωπαϊκής Ένωσης αν μη τι άλλο. Αν λοιπόν αρνείται κανείς σε ένα παιδί πρόσβαση, σε παιδεία, σε εκπαίδευση και αυτό επηρεάζει την οικονομική ζωή, τότε σίγουρα αυτό πρέπει να χαρακτηριστεί ως κοινωνικός αποκλεισμός και ο κοινωνικός αποκλεισμός απαγορεύεται από τις ευρωπαϊκές συνθήκες. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να στείλουμε ένα ερωτηματολόγιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μάλλον να στείλει ένα ερωτηματολόγιο στα ευρωπαϊκά σχολεία, προκειμένου να ενημερωθούμε για τα επίπεδα αναπηρίας τα οποία δέχονται τα σχολεία αυτά στα... όσον αφορά τους μαθητές. Κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να συνειδητοποιήσουμε πόσο σημαντικό είναι το πρόβλημα και θα συνειδητοποιήσουμε επίσης και τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για να λύσουμε το πρόβλημα αυτό ενδεχομένως να πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη χρηματοδότηση προκειμένου να μπορούν τα σχολεία αυτά να δεχθούν περισσότερους μαθητές με αναπηρία και το πιο σημαντικό να καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα ασχοληθούμε με τις βασικές ανησυχίες και την κατάφορη παραβίαση των αρχών στις οποίες αναφέρεται ο Βασίλης σήμερα στην αφορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κάσμαν. Ε, το σημειώσαμε κιόλας. Η κυρία Βέθμαν. Ευχαριστώ. Θα συμφωνήσω σε πολλά με τους προλύσαντες, ειδικά για το ε, ειδικό καθεστώς που, ε, για το οποίο μιλούμε για τα παιδιά τα αυτιστικά. Ο αυτισμός είναι, χρειάζεται ειδική, ε, ειδική αντιμετώπιση εγώ ήμουν εκπαιδευτικό πριν, πριν μπω στην πολιτική και πραγματικά υπάρχουν, έχουν ακουστεί πάρα πολύ καλέ ιδέε. Είναι καλό αυτό που ακούστηκε από την Κομισιόν ότι υπήρξαν δύο καθηγητέ που συνόδευαν το παιδί για να μπορέσει το παιδί να τα καταφέρει. Όταν όμω και το παιδί ξέρει ότι, ποια είναι τα ε, όρια του, μπορούμε και εμεί να σεβαστούμε το δικαίωμά του στην εκπαίδευση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και μιλάω και ως μητέρα τώρα είναι σημαντικό να ενσωματώνονται τα παιδιά. Τα παιδιά με αυτισμό είναι εξαιρετικά παιδιά. Έχουν ε, ειδικά, ιδιαίτερα ταλέντα. Και το είπε η Κομισιόν, έχουν ε, ταλέντα στη, στα μαθηματικά, στα αθλητισμό, στην καλλιτεχνία. Οπότε δεν θα πρέπει να μιλούμε για αποκλεισμό ή για ένταξη, αλλά για ενσωμάτωση στην κοινωνία να χρησιμοποιήσουμε δηλαδή αυτές τις ειδικέ ποιότητες ε, προσόντα που έχουν αυτά τα παιδιά, όχι να τα βάζουμε στη γωνία. Φυσικά είναι πολύ δύσκολο γιατί αυτό που ζει η οικογένεια του Βασίλη, που είναι χωρισμένη όλη την εβδομάδα για να μπορεί το παιδί να πηγαίνει στο σχολείο. Πρέπει λοιπόν η οικογένεια αυτή να λαμβάνει την προστασία και την ε, ε, πρόνοια που χρειάζεται. Έτσι είναι δουλέψω στη δική μου την ε, πατρίδα και πραγματικά εγώ θα ε, ε, με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό που είπε και ο συνάδελφος για την επιστημονική ανάλυση. Βέβαια τώρα να μην περάσουμε στο πινκ πονγκ να μιλάει, να κάνει ο ένας κάτι, να πηγαίνει πίσω, να ξανααναλύεται κτλ. Να, γίνει, να αναλυθεί μια δράση που να βοηθήσει το παιδί γιατί πραγματικά αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα ήθελα λοιπόν όντω να το δούμε ο, τι χρειάζεται ο αυτισμός, τι, ποια είναι τα, τα βήματα που πρέπει να αναλυθούν, γιατί πραγματικά ε, εμείς οι ενήλικέ πρέπει να κάνουμε πολλά. Φυσικά είναι μεγάλο το βάρο που αντιμετωπίζει μια οικογένεια με παιδί με αυτισμό. Οπότε ό,τι μπορούμε να κάνουμε είναι καλό. Το να είναι κανεί εδώ πέρα και να είναι χωριστά από την οικογένειά του, ε, δεν είναι και πολύ εύκολο, σκεφτείτε το, αλλά πρέπει πάντα να έχουμε υπόψη μα τι ειδικέ, οι δυνατότητε που έχει το παιδί αυτό και ποιο είναι το καλό του και πώ αυτό μπορεί να ενσωματωθεί στην, στην κοινωνία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε εμεί κύριε Βέρτμαν. Ε, πολύ σύντομα κύριε Τουργκάη, παρακαλώ. Ναι, πολύ σύντομα κύριε Πρόεδρε. Ούτε και εγώ γνωρίζω, ούτε γνώριζα τον κύριο Κατσιούλη. Χαίρομαι που το γνωρίζω σήμερα εδώ. Αλλά τι γίνεται. Εάν, κύριε Πρόεδρε, έψαχνα θέση σε ένα σχολείο για τα παιδιά μου, αφού άκουγα την Επιτροπή, έκανατε την καλύτερη προπαγάνδα για να μην πάω σε αυτό το σχολείο τα παιδιά μου. Και είμαι καθηγητής ο ίδιος, ε, δάσκαλος. Και εάν ξέρουμε τι γίνεται για μια ένα έννοια τα υπερπαιδιά, τα καλύτερα σε μαθηματικά, φυσική, σε μουσική, σε σχολείο, σε ε, σπορ, ε, ε, τότε χρειάζεται το ειδικό σχολείο, αλλά τα παιδιά μου και τα δύο πάνε στο ίδιο σχολείο τα δύο παιδιά μου και το ένα έχει δυσκολίες εκεί στο σχολείο. Τι γίνεται, θα πρέπει να βγει από το σχολείο. Αντίθετα, θα πρέπει να μπει εκεί ένας καθηγητής, ένας δάσκαλος να μπορεί να παρακολουθήσει το παιδί σύμφωνα με τις δυνατότητές του. Αυτό μπορεί να παρακολουθήσει, αλλά όχι να φτιάξει κανείς ένα σχολείο με σούπερ παιδιά, με προσωπικότητες εδώ και εκεί. Εντάξει, αυτό θα ήταν και εύκολο αν θέλετε για το σχολείο. Ε, σας το λέω σύμφωνα και με την πείρα μου, εντάξει, καλό θα ήταν, αλλά τι γίνεται, το δύσκολο ποιο είναι να βρούμε ακριβώς τις λύσεις που λέει ο αναφέρον, ε, τα προβλήματα, να δούμε ποιες είναι αυτές οι λύσεις και στο σχολείο αυτό, για να μην ε, ε, διώξουν το παιδί και να το πάνε σε δεκάδες χιλιόμετρα απόσταση με προβλήματα για το παιδί και για την οικογένεια. Αυτά κύριε Πρόεδρε. Και ακούστε, εγώ άκουσα τις ε, εξηγήσεις που δόθηκαν, ε, συμφωνώ αυτό που η κυρία Ράπτη και ο κύριος Κάσμαν ε, και συνάδελφος εδώ και θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά. Αλλά το πιο δύσκολο εδώ, κύρια Πρόεδρε, είναι να δούμε πώς μπορούμε να βρούμε μια λύση σε αυτό το πρόβλημα. Δεν ξέρω, παραμένοντας ανοιχτή η υπόθεση αναφορά, θα είχαμε το χρόνο για να το μελετήσαμε ή ο ίδιος ο αναφέρον να μπορέσει να μας υποδείξει μια λύση για να δούμε κι εμείς, όπως το κάναμε και σε άλλες περιπτώσεις, πώς θα απευθυνθούμε στο Συμβούλιο, δεν ξέρω, μια επιστολή, κάτι να κάνουμε τέλος πάντων, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε το παιδί αυτό. Γκόντς, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ σύντομα. Μόλον ότι είμαι ψυχίατρος πρέπει να πω ότι το ζήτημα δεν είναι ψυχολογικής φύσης. Εδώ πέρα μιλάμε για τα καθήκοντα του σχολείου, του Ευρωπαϊκού Σχολείου. Επίση, θα ήθελα να επικρίνω την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέκρινε ένα παιδί με ειδικέ ανάγκες με τα παιδιά εκείνα που έχουν ιδιαίτερα ταλέντα και που θα πρέπει να κατευθυνθούν προς το ένα ή το άλλο εξειδικευμένο σχολείο. Νομίζω ότι δεν τίθεται τέτοια σύγκριση και νομίζω ότι θα αντιμετωπίσετε αρκετά προβλήματα με την προσέγγιση αυτή που έχετε. Θεωρώ ότι θα πρέπει να είμαστε απόλυτα σαφείς ότι τα ευρωπαϊκά σχολεία, καθήκον των ευρωπαϊκών σχολείων, να βρουν έναν τρόπο να εκπαιδεύσουν τα παιδιά είτε έχουν ειδικέ ανάγκε ή δεν έχουν ειδικέ ανάγκε. Να βρουν έναν τρόπο να του παρέχουν παιδεία, να βρουν έναν τρόπο να του παρέχουν του κατάλληλου καθηγητέ, έναν τρόπο προκειμένου να καταφέρουν να επιτύχουν την ενσωμάτωση. Νομίζω θα πρέπει να είμαστε απόλυτα ξεκάθαροι απέναντι σε αυτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Γκέντς. Ε, κύριε Ντερόσα. Ο κύριος Ντερόσα. Σας ευχαριστώ. Δεν σας άκουσα την πρώτη φορά σας, το συγγνώμη. Καταρχάς πρέπει να σας πω ότι έχω ξαναδεί το σκηνικό αυτό και στο παρελθόν. Γιατί το 2006 ήμουν εισηγητής για ένα ζήτημα το οποίο πήγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Πρόκειται για μια διαδικασία που είχε ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη από το 2003. Και ακούγοντας συζήτηση σήμερα και ξαναδιαβάζοντα την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τότε το 2003, όσον αφορά πάλι τότε έναν υπάλληλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είχε ανάλογα προβλήματα, μπορώ να σας πω ότι κατά λέξη σχεδόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε τα ίδια πράγματα. Είπε ότι ε, και τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι κάνει κάθε τι προκειμένου να βοηθήσει τα παιδιά με αναπηρίες για να ενσωματωθούν κτλ. Και έχουμε και μία έκθεση του συνηγόρου του πολίτη του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, ο οποίο είχε ταχθεί κατά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα επιχειρήματα που είχε εκφράσει τότε στο παρελθόν το 2003. Βάσει των πληροφοριών αυτών θεωρώ ότι δεν έχει σημειωθεί καμία πρόοδος καθότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για άλλη μια φορά ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ασχοληθεί με το ζήτημα αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Σχολείου, επομένω επηρεάζει και τον προπολογισμό των σχολείων αυτών αλλά και πάλι βλέπουμε ότι τα όσα μας λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σήμερα δεν μπορούν να είναι αποδεκτά. Δεν μπορούμε να δεχθούμε μια κατάσταση όπου τέσσερα χρόνια τελικά αργότερα πάλι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η δική μας Επιτροπή αναγκάζουν να ασχοληθούν με το ίδιο ζήτημα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το μόνο που κάνει είναι έρχεται εδώ πέρα και να επαναλαμβάνει την απάντηση που έδωσε στο παρελθόν. Δηλαδή ότι τα σχολεία αυτά είναι πρότυπα σχολεία τα οποία δεν ε, ε, είναι καταρτισμένα κατά τρόπον ώστε να δεχθούν ε, παιδιά με ειδικέ ανάγκες. Θεωρώ ότι τα σχολεία αυτά θα πρέπει να μπορούν να ενσωματώσουν τα παιδιά με ειδικέ ανάγκες και αν από οικονομικής πλευράς δεν είναι δυνατό να γίνει κάτι τέτοιο, τότε ξέρετε ότι όλοι οι γονεί έχουν το δικαίωμα να παρέχουν δωρεάν εκπαίδευση στα παιδιά του, αν μη τι άλλο στο Βέλγιο, και θα πρέπει αυτό να ληφθεί υπόψη από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Δηλαδή δεν μπορεί να ζημιώνεται ένας γονέας επειδή έχει ένα παιδί με ειδικέ ανάγκε και αναγκάζεται τελικά να πληρώνει χιλιάδες ευρώ ετησίως μόνο και μόνο για να παρέχει βασική εκπαίδευση στο παιδί του, ενώ έχει το βασικό δικαίωμα τη δωρεάν παιδείας Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Τιντερόσα. Ε, πάρα πολύ σύντομα κύριε Κατσιούλη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Χαίρομαι που άκουσα όλα αυτά τα σχόλια. Εμείς είχαμε πει σαφώς πριν υπογράψω εγώ τη σύμβαση με το Κοινοβούλιο, είχαμε πει στο Ευρωπαϊκό Σχολείο τι ακριβώ πρέπει να γίνει για να τύχει τι καλύτερε δυνατέ εκπαίδευση στο παιδί μου. Και είπαμε ότι ο Λούκα πρέπει να υπαχθεί στην μέθοδο ABA. Έτσι ώστε να μπορέσει να ενσωματωθεί στο σχολείο και να παρακολουθήσει. Εγώ συζήτησα με τον ε, αρμόδιο στην υπηρεσία μου το Ευρωπαϊκό, Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συγγνώμη, Σχολείο λαμβάνει κάτι 3,6 εκατομμύρια. Ε, τέσσερις μέρες πριν έρθουν αυτοί οι άνθρωποι για να ε, δώσουν την συμβουλή τους ας πούμε στο σχολείο, για τη δική μας την περίπτωση, το σχολείο μας απέρριψε. Και έρχονται τώρα εδώ πέρα άνετοι και Μάλιστα, μέχρι πριν, πριν από δύο μέρες έλαβα εγώ μια επιστολή που μου λέει ότι δεν μπορούμε να αναλάβουμε τα έξοδά σα. Ε, υπάρχει μέθοδος για το δικό μου το γιο. Αυτή η μέθοδος δεν έχει χρησιμοποιηθεί. Και με τη μέθοδο αυτή τα παιδιά που έχουν αυτισμό μπορούν να ε, λαμβάνουν εκπαίδευση μέσα στο σχολείο. Μέχρι στιγμής αυτό δεν έχει γίνει. Και γι' αυτό λέω, και πολύ σωστά το είπε ο κύριος ε, ε, Guys, ότι ναι εντάξει μπορεί να υπάρχουν προβλήματα κτλ αλλά θα μπορούσε κανείς έστω να προσπαθήσει να εισάγει αυτή την μέθοδο στο σχολείο για να δει δηλαδή ότι μπορεί να λειτουργήσει. Μέχρι στιγμής αυτό δεν έχει γίνει. Ε, αυτό είναι αυτό που λέω εγώ και ανεξάρτητα με την σύμβαση ε, του ΟΗΕ, η οποία ούτω ή άλλω εξασφαλίζει το ότι οποιοδήποτε παιδί έρθει στο σχολείο σα δεν μπορείτε να το αποκλείσετε. Ευχαριστώ και συγγνώμη που έτσι αγανάχτησα λίγο, αλλά καταλαβαίνετε είναι πολύ προσωπικό το θέμα. Σα ευχαριστούμε, δεν είναι προσωπικό τελικά, φαίνεται ότι είναι πολύ πιο γενικό και σας ευχαριστούμε για αυτό το δυνατότητα που μας δίνετε να σκεφτούμε ξανά μερικά πράγματα. Πριν, ναι, παρακαλώ κυρία Μπαρντού. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Ορισμένα συγκεκριμένα στοιχεία για παρατηρήσεις που ακούστηκαν, οι σχόλια που έγιναν, ε, είπαν αρκετοί ότι χρειάζονται ειδικοί και παιδοψυχίατροι κλπ. Να διευκρινίσω κάτι σε ευρωπαϊκό σχολείο. Όταν αναλαμβάνεται ένα παιδί με πρόβλημα, Έχουμε μία ομάδα επαγγελματιών που μελετάει την υπόθεση, βλέπει ποιες ανάγκες του παιδιού, τι γίνεται, πώς έχει κατάσταση και αυτή η επιτροπή ειδικών παίρνει την απόφαση σε τελικό στη τελική φάση αν το σχολείο μπορεί να εντάξει το παιδί. Κάθε φορά που λαμβάνεται μια απόφαση αφού το σχολείο λέει ότι δεν είναι το αρμόδιο για να εντάξει αυτό το παιδί υπάρχει μια απόφαση με μια ομάδα ειδικευμένη σε παρόμοια θέματα. Δεν είναι ότι ο διευθυντής μόνος το αποφασίζει μετά από μια συγκεκριμένη λύση από αρμόδια εξειδικευμένα άτομα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, χρειάζεται να το διευκρινίσουμε. Και ακόμα κάποιο μίλησε για παιδιά, με σούπερ παιδιά που θα πρέπει να πάρουμε τα καλύτερα εμείς εκεί. Όχι, δεν είναι αυτό για το Ευρωπαϊκό Σχολείο. Πολλά παιδιά έχουν δυσκολίες εκμάθησης, είτε υπάρχουν συμφωνίες λόγω ειδικών αναγκών και ιδιαίτερα βοηθούνται αυτά τα παιδιά η πραγματικότητα ποια είναι. Υπάρχουν και ορισμένε περιπτώσει που κηρύσσει αυτό αρμόδιο το σχολείο. Δεν μπορεί να αντιμετωπίσει. Δεν είναι σημαίνει ότι όποια παιδιά δεν μπορούν να μάθουν, ε, αποκλείονται, διώχνονται. Υπάρχει και ειδικό λογαριασμό για αυτό το learning support, για την στήριξη, για την εκμάθηση και πολλά παιδιά έχουν βοηθηθεί από αυτό. Είναι πάντως ένα παράδειγμα που δείχνει πόσο βοηθούνται τα παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίε. Ίσως δεν ήμουν σαφής στην επαχειροτομαλογία μου για κάθε τι που δεν προτείνεται σαν εκπαίδευση στο Ευρωπαϊκό Σχολείο για άλλους τομείς. Τι μπορεί να κάνω, κανεί τι μπορεί να προσφέρει, ιδιαίτερα διαφοροποιημένο. Μπορεί να υπάρχουν σχολεία με διάφορες προφορές, προσφορές εξειδικευμένες σε πολλούς τομείς. Το ευρωπαϊκό σχολείο είναι κάτι περισσότερο ομοιόμορφο, α το πούμε έτσι. Δεν μπορεί να διαφοροποιηθεί τόσο όπω εθνικό επίπεδο μπορεί να γίνει στα σχολεία. Και σε ορισμένε περιπτώσει ακριβώ ε, μα περιορίζει η κατάσταση σε σχέση με άλλα σχολεία Και γι' αυτό μερικέ φορέ ε, κηρύσσουμε αυτού αναρμόδιου για να αντιμετωπίσουν μια παρόμοια κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι είναι καιρό ίσω να ξανασκεφτούμε το ρόλο των ευρωπαϊκών σχολείων. Ίσως είναι ο μόνος τρόπος για να δούμε αν στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε να κάνουμε με μια διάκριση, ε, ε, μια κοινωνική διάκριση ή για μια επιστημονικά επιβεβλημένη απόφαση που, οδήγησε στην περίπτωση του κ. Κατσούλη στο ότι για το καλό του παιδιού έπρεπε να φύγει από αυτό το σχολείο και να πάει καλό. Όχι για το καλό του, του, του διδακτικού προσωπικού ή οποιοδήποτε άλλου που δηλώνει αναρμόδιο να αντιμετωπίσει δικές περιπτώσεις. Πραγματικά νομίζω ότι τώρα περισσότερο από ποτέ πρέπει να ξαναδούμε το ρόλο και την ε, αποστολή των ευρωπαϊκών σχολείων στη γενικότητά του. Συμφωνώ με τον κύριο Κάσμαν για την έρευνα που θα έπρεπε να γίνει και αφορά τη λειτουργία ε, των ευρωπαϊκών σχολείων γενικότερα παράλληλα με το ότι αυτή η αναφορά δεν το συζητάμε ότι πρέπει να παραμείνει ανοιχτή και ίσως πραγματικά ακολουθώντας και την προηγούμενη περίπτωση να προτείνουμε μια ακόμη προφορική ερώτηση στην ολομέλεια όπως και για την προηγούμενη περίπτωση πάλι του κ. κατσούλη. σε αυτή την περίπτωση θα με να την, θα μπορούσα να την κάνω εγώ. ευχαριστώ πολύ. Και τώρα το σημείο 9 της ημερήσιας διάταξης είναι παρόμοιο θέμα με το προηγούμενο και έτσι συμπληρώνουμε την όλη συζήτηση. Είναι 840 του 2007, η Τρεζαχέης είναι απούσα και ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Σιλβιο Γκρέκο, έχει το λόγο για να μας πει πώς έχουν τα πράγματα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μια που δεν είναι εδώ η αναφέρουσα να σας αναφέρω εγώ κάποια στοιχεία της ε, αναφοράς και να κάνω και τα σχόλια εκ μέρους της Επιτροπής. Η αναφορά αφορά ε, την ε, αμέλεια για, την, για τα παιδιά που πάσουν από αυτισμό στην Ιρλανδία. Η αναφέρουσα λέει ότι το παιδί της δεν έχει λάβει ποτέ πρωτογενή, πρωτοβάθμια συγγνώμη, εκπαίδευση την οποία δικαιούται σύμφωνα με το Σύνταγμα. Υπάρχουν και κάποια άλλα σημεία τα οποία επίσης ε, σχετίζονται με την αναφορά για δυσκολίες δηλαδή που αντιμετωπίζει η οικογένεια αλλά και άλλες οικογένειες για, την, για τα σχολεία αυτά ABA, τις εφαρμοσμένες ανάλυσης συμπεριφοράς δηλαδή τα οποία δικαιονται σε τέτοιου είδους εκπαίδευση για παιδιά δηλαδή με αυτισμό. Τώρα, σύντομα να αναφερθώ σε δύο εργαλεία τα οποία ήδη ε, ακούστηκαν από τους συναδέλφους μου. Υπάρχει το σχέδιο οδηγίας για την ίση μεταχείριση και στο χώρο εργασία και η σύμβαση των, του ΟΗΕ για, τα παιδιά με, για τους ανθρώπους με αναπηρίες. Να πω απλώς ότι το, ε, το θέμα αυτό είναι διαδικαστικό, δεν θα το σχολιάσω γιατί το είπαν ήδη οι υπόλοιποι. Ε, η έκθεση λοιπόν καλύπτει, η αναφορά καλύπτει και τον τομέα της εκπαίδευσης και σύμφωνα με την οδηγία τα κράτη-μέλη θα πρέπει να παράσχουν τα μέτρα που είναι απαραίτητα ώστε να διευκολύνουν τα άτομα με αναπηρία να έχουν μια αποτελεσματική και χωρίς διακριτική μεταχείριση πρόσβαση στην εκπαίδευση και χρειάζεται να παράσχουν και την, τις εύκολες προσαρμογές, εκτός αν αυτές συνεπάγονται δυσανάλογη επιβάρυνση. Uh, Αυτά για, την, ε, για το σχέδιο οδηγία. Σε κάθε περίπτωση αυτή η πρόταση ε, Φυσικά λαμβάνει υπόψη και τις αρμοδιότητες των κρατών μελών, ειδικά σε ό,τι αφορά την οργάνωση και το περιεχόμενο του, ε, του συστήματος εκπαίδευσής τους. Και βέβαια υπάρχουν και αναφορές για την εκπαίδευση για παιδιά με αναπηρία. Ακόμη αυτή η οδηγία δεν έχει εγκριθεί. και το θέμα που αναφέρει η αναφέρουσα πρέπει να ε, υπαχθεί στους, ε, στο Ιρλανδικό δίκαιο. Επίσης, να αναφερθώ στις διατάξεις που αφορούν την, ε, που αναφέρονται, περιλαμβάνονται συγγνώμη, στην σύμβαση του ΟΗΕ Ειδικά το άρθρο 7 και το 24 που αναφέρονται στα δικαιώματα των παιδιών με αναπηρία και στα δικαιώματα που έχουν αυτά στην εκπαίδευση. Η σύμβαση ε, λέει ότι τα συμβαλόμενα μέρη εξασφαλίζουν ένα εκπαιδευτικό σύστημα χωρίς εκποκλισμούς σε όλα τα επίπεδα και με βάση τις ίσες ευκαιρίες η Ιρλανδία, όπω όλα τα υπόλοιπα 27 κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει επικυρώσει τη σύμβαση, αλλά ακόμη δεν την έχει, ε, την έχει υπογράψει, δεν την έχει επικυρώσει. Οπότε, όταν επικυρωθεί η σύμβαση, θα ισχύσουν και θα είναι δεσμευτικέ και οι διατάξει τη. Προ το παρόν όμω αυτό δεν έχει γίνει. Δεν έχει εγκριθεί η σύμβαση από την Ιρλανδία. Τώρα, για τα πιο σκληρά μέτρα για τα πιο ήπια μέτρα. Εντάξει, η Κομισιόν αυτό που κάνει είναι να υποστηρίζει το δικαίωμα των ανθρώπων με αναπηρία στην ε, εκπαίδευση. Πριν η συνάδελφος μίλησε για το ακαδημαϊκό δίκτυο για των εμπειρογνωμόνων για ανθρώπους με αναπηρίες μίλησε για τη μελέτη για την ε, κάρτα ε, για, την αναπηρία και τα ωφέλη. Ε, τώρα κάτι παρόμοιο γίνεται φέτος στον τομέα της εκπαίδευσης με ακαδημαϊκούς που κάνουν μια, ένα εγχείρημα και στα πλαίσια της οδηγίας πλαίσιο για όλα τα κράτη-μέλη ειδικά για τα παιδιά με αναπηρία και την εκπαίδευση των παιδιών αυτών και βεβαίω αυτό έχει να κάνει και με τους πόρους που δαπανούν τα κράτη-μέλη ώστε να εφαρμόσουν και να εξασφαλίσουν ότι τα παιδιά αυτά θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα σχολεία και στην εκπαίδευση με βάση την ίση μεταχείριση. Ιδού. Λοιπόν, η βασική απάντηση στην αναφορά αυτή είναι ότι η δυνάμη του κεκτημένου αυτό εμπίπτει στην εθνική αρμοδιότητα και όχι στην ευρωπαϊκή. Σας ευχαριστούμε. Κάποιος θα επιθυμούσε να λάβει το λόγο παρακαλώ. Κανείς. Ναι, εσείς. Νομίζω ότι θα πρέπει να γίνουν κάποιες παρατηρήσεις. Όπως είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ζήτημα εμπίπτει στην εθνική νομοθεσία. Αυτό όμως το λέει ήδη και η αναφέρουσα. Είπε ότι προσπάθησε να δικαιωθεί μέσω των Ιρλανδικών δικαστηρίων, αλλά απέτυχε στην προσπάθειά της αυτή, γι' αυτό απευθύνεται σε εμά τώρα. Νομίζω ότι ε, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι ε, οι αναφέροντες αν μη τι άλλο πρέπει να έχουν μια απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της δικής μας Επιτροπής και εφόσον ε, έχουν έρθει σε επαφή με ευρωβουλευτές από την εκλογική τους περιφέρεια, τότε θα πρέπει να δοθεί ενδεχομένω και μια συνέχεια, να έχουν το δικαίωμα δηλαδή να λάβουν από τους βουλευτές αυτούς κάποιες περισσότερες πληροφορίες. Σε κάθε περίπτωση πάντως και η περίπτωση αυτή ενδυναμώνει το επιχείρημα για την οδηγία πλαίσιο για τη διακριτική μεταχείριση, για την καταπολέμηση διακριτική μεταχείρισης. καταλαβαίνετε ότι δεν είναι δυνατόν να έχουμε οδηγίες, ε, κοινοτικέ ρυθμίσεις που θα απευθύνονται σε κάθε μία περίπτωση ξεχωριστά. Θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει μία κοινοτική οδηγία σφαιρική η οποία θα καταπολεμά κάθε διακριτική μεταχείριση. Το πρόβλημα βέβαια είναι ότι το σχέδιο αυτοδηγίας έχει ε, μπλοκαριστεί στο Συμβούλιο, συναντά εμπόδια εκεί και το πρόβλημα είναι ότι ε, και αυτή η αναφορά και οι προηγούμενες αναφορές αναφέρονται σε προβλήματα τα οποία δεν θα ίσχυαν αν η οδηγία αυτή την είχε μπλοκαριστεί. Πρέπει να γράψουμε λοιπόν στο Συμβούλιο και να του ζητήσουμε να λάβει τι ευθύνε του. Uh, θα είμαι πολύ σύντομο, Πρόεδρε. Σε προηγούμενη αναφορά μου αναφέρθηκα στην uh, αναφορά αυτή. Θα ήθελα να πω ότι uh, η συγκεκριμένη αναφορά τονίζει για άλλη μια φορά ότι, δεν υπάρχουν, ότι κάποιες συγκεκριμένε αρχές που δεν τυχαίνουν σεβασμού όσον αφορά τα άτομα με ανάγκες και πιο συγκεκριμένα την εκπαίδευση των παιδιών με αυτισμό. Το ζήτημα αυτό είναι πολύ δύσκολο και ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο στην ε, Ιρλανδία. Υπάρχουν πάρα πολλοί γονείς οι οποίοι συνειδητοποίησαν ότι η Ιρλανδική κυβέρνηση έθελε τυφλή απέντη στις πραγματικές αυτές τρανταχτές ανάγκες των παιδιών τους και προσπαθεί ουσιαστικά να προτείνει κάποιες γενικές λύσεις που δεν είναι λύσεις και που έχουν αναγκάσει τελικά γονείς να προχωρήσουν σε τεράστιες θυσίε. Υπάρχουν γονείς που έχουν ιδρύσει σχεδόν ολόκληρο σχολείο μέσα στο σπίτι για να προσφέρουν κατοίκον εκπαίδευση με συγχωρείτε στα παιδιά τους. Γονείς οι οποίοι πληρώνουν πάρα πολλά χρήματα προκειμένου να καταφέρουν να παρέχουν μια στοιχειώδη παιδεία στα παιδιά τους. Και αυτό γιατί δεν μπορούν να σωματωθούν τα παιδιά τους στο γενικότερο σύστημα παιδείας στην Ιρλανδία. Πρέπει λοιπόν το κράτος να φουγκραστεί πραγματικά τους γονείς, να ακούσει την εμπειρία που έχουν συσσωρεύσει οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι ασχολούνται σε καθημερινή βάση, στακτική βάση, με θέματα αναπηρίας. Ακόμα και στα πλαίσια του συντάγματος κατοχυρώνεται το δικαίωμα της ε, παιδείας. Το πρόβλημα όμως δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι η φύση της εκπαίδευσης που παρέχεται προς το παιδί αυτό. Και βλέπουμε τελικά ότι ακόμα και η Ιρλανδία πρέπει ακόμα να κάνει σπουδαία βήματα και υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Χριστό, Το κείμενο της αναφοράς αυτής και θα μπορούσαμε να πούμε ότι ακούσαμε προτάσεις εδώ που θα μπορούσαν να συνδυαστούν με άλλες αναφορές όπως ακριβώς να ζητήσουμε την επικύρωση της σύμβασης και να έρθουμε και σε άλλο θέμα παρότριση στην Επιτροπή να προχωρήσει καλύτερα για μια συμφωνία, για μια καλύτερη παρέμβαση σε παρόμοιες περιπτώσεις μέχρι και το ερώτημα που θα έπρεπε να υποβάλλουμε στην Επιτροπή, όπως είπε η συνάδελφος, για να επισπεύσουμε την διαδικασία. Παραμένει ανοιχτή η αναφορά. Έτσι λοιπόν συνεχίζουμε και εφαρμόζουμε αυτά που είπαμε ότι θα ακολουθήσουμε. Και τώρα η επόμενη, η 15. 15. Το είχαμε κάνει και σε άλλες περιπτώσεις και επειδή έχουμε καθυστερήσει θα πρέπει να δούμε τις ε, αναφορές που είναι παρόντες ή αναφέροντες. Ε, είναι οι 15 η αναφέρουσα είναι παρούσα, είναι 1696 του 2008. Η Ζακλίν Ντεκρουά έχει το λόγο. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για την υποδοχή σας, για την προσκλησή σας θα σας μιλήσω για ένα πρόβλημα που λαμβάνει τεράστιες διαστάσεις στη Γαλλία και στον κόσμο ολόκληρο για τις ε, εικόνες ε, πραγματικών εγκλημάτων ε, σχετικά με παιδιά και 3% του πληθυσμού αφορά από τη λένε οι γαλλικές στατιστικές και στο Βέλγιο Έχουμε 300.000 άτομα που αφορά το θέματα και 22 εκατομμύρια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Είναι θέμα πάρα πολύ ευαίσθητο και φοβίζει και τις κυβερνήσεις γιατί σημαίνει η διαφθορά και της αστυνομίας και τα κύρια θύματα είναι παιδιά. Παιδιά σε διάφορα ιδρύματα και που θα πρέπει να υπάρχει μια κατάλληλη αντιμετώπιση για να σωθούν αυτά τα παιδιά, κάτι που δεν γίνεται. Και αυτές οι περιπτώσεις ε, κλείνουν και θεωρούνται και κρατικά απόρριτο σε ξεχωριστούς φακέλους ε, και πήγα μια φορά εγώ στην ε, αστυνομία, δεν μπορούσα να με ικανοποιήσει, μου είπε η αστυνομία ότι ήταν κωδικοποιημένο σε φάκελο το θέμα έχει να κάνει με θέματα ακριβώ που τραντάζουν τα θεμέλια του κράτους. Και από ό,τι είδαμε έκπληξη, ε, η προσφυγή μου δεν έγινε δεκτή λόγω έλλειψη στοιχείων. Ποια ακριβώ στοιχεία θα μπορούσα εγώ να επικαλεστώ για να ταράξω τα θεμέλια του κράτους. Δεν ήξερα. Ε, περιπτώσει περιπτώσεις ε, συναντάμε παντού στην Ευρώπη. Ποιο είναι το χειρότερο τώρα ότι όσοι προσφεύγουν, όσοι διαμαρτύρονται, όταν δεν σωπαίνουν μια κάποια στιγμή υπάρχουν και αποφάσεις δικαστικές λανθασμένες. Παιδιά που κλείνονται στη φυλακή ενώ υπάρχουν ιατρικές αποδείξεις ότι δεν μπορούσαν τα παιδιά αυτά να διαπράξουν το έγκλημα για το οποίο έχουν κατηγορηθεί και βλέπουμε ότι επίσης καταδικάζονται ουσιαστικά σε θάνατο επειδή υπάρχουν συνθήκες κράτησης τρομερές και απέσιες, χειροτερεύει η υγεία τους, επιδεινώνεται η κατάστασή της, και πολλά τρομερά πράγματα συμβαίνουν και στο Βέλγιο ακόμα που πιστεύουμε ότι πρόκειται για ένα κράτος δικαίου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σεβασμού τους και όταν κάποιος ε, εδώ και τρία χρόνια έχει ένα καρκίνο και μπαίνει στη φυλακή και κανείς δεν τον προσέχει, κανείς δεν παρακολουθεί την υγεία του, καταλαβαίνετε τι γίνεται. και καποιο ηταν ήταν 590-600 ε, ώρες ε, με χειροπέδες κανονικά. Όταν μπαίνει κάποιο στη φυλακή δεν πρέπει να διατηρηθούν οι χειροπέδες και αυτό ε, βάσει... Αυτό είχε γίνει το 1998 και μάλιστα με ένα δελτίο που έδειξε ότι υπάρχει αυτή η σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών δόθηκε και ε, συγχαρτήρια για τη διαλεύκαση αυτού εγκλήματο από το του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά παντού εδώ και εκεί ε, μπήκαν ε, στο αρχείο διάφορες περιπτώσεις, ποτέ δεν έγινε μια έρευνα εκτός από δύο-τρεις φορές 88.500 φωτογραφίες υπάρχουν θυμάτων και βλέπουμε παντού ότι είναι και θύματα η κυρία εδώ δίπλα σε μένα ας πούμε βρέθηκε στη φυλακή, κλείστηκε στη φυλακή γιατί δεν αναγνώρισαν μια εργαστηριακή ανάλυση που έλεγε ότι είχε μια σεξουαλική αφροδίσια, ένα αφροδίσιο νόημα, ε, νόσημα, συγγνώμη, σε, σε, ηλικία 7 ετών. Και τα κυρία δεν ήξερε την περίπτωση, εγώ το βρήκα στο ίντερνετ, δεν ήξερε την ίδια την περίπτωσή της, καταλαβαίνετε. Εδώ αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση τρομερή και ο τύπος δεν δείχνει καθαρά τα γεγονότα όπως συμβαίνουν. Ο εισαγγελέα δίνει τη δική του εκδοχή χωρίς τίποτα το πιο συγκεκριμένο και το 1998 υπόθεση αυτή έχουμε ένα και ένα παράρτημα με 40 εκατομμύρια φωτογραφίες. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Και όλα και χειρότερα προβλήματα θα αντιμετωπίζουμε από τη στιγμή που κάθε χώρα παραβιάζει τον νόμο, τον εθνικό και το διεθνή όμως. Αυτό συμβαίνει. Και κάποιος συνάδελφος είναι στη φυλακή και είναι το δικαστικό συμβούλιο υπάρχει απόδειξη ότι εξαφανίστηκαν στοιχεία από το φάκελό του. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι σε μια τσέπη αν τα έχω θα μπορούν να μου τα πάρουν κιόλας να τα χάσω, αλλά όχι σε ένα φάκελο και αναγνωρίστηκε ότι είχε δικαστεί, καταδικαστεί βάσει μη πλήρους φακέλου και στοιχείων και παντού έχουμε παρόμοιες περιπτώσεις που συμβαίνουν και βλέπουμε πολλές φορές ότι δεν δημοσιεύει εύονται αυτές οι περιπτώσεις. Ξέρουμε ότι είναι και στημένε υποθέσει μερικές φορές. Τα βλέπουμε στο ίντερνετ ε, όταν έχουμε παρόμοιες δραματικές περιπτώσεις και υπάρχουν παιδιά στην όλη περίπτωση. Ακούμε 3% του παγκόσμιου πληθυσμού. Έχουμε 180 εκατομμύρια άτομα. Είναι άτομα αυτά που θα πρέπει να καταλάβουμε ότι οι παιδιά που έχουν ζήσει παρόμοιες καταστάσεις είναι καταδικασμένα να φέρουν τραύματα σε όλη τη ζωή ψυχολογικά και για να μπορέσει να μεγαλώσει ένα παιδί χρειάζεται δικαιοσύνη και όμως δείχνουν όλες οι στατιστικές ότι το 100% των κατ' δολοφόνων είναι παιδιά που έχουν προβλήματα μικρά, ποτέ τους αποδόθηκε δικαιοσύνη. Πολλοί κατ' επανάληψη δολοφόνοι, κανείς όμως δεν ψάχνει το φάκελό τους, λένε «Α, είναι τέρατα αυτός, αυτά τα άτομα και υπάρχουν και κόσμος, υπάρχουν άτομα, παιδιά που ε, εκπορνευόταν, ε, πολλά προβλήματα, κανείς όμως από δικαιοσύνη δεν παρενέβη υπέρ αυτών των παιδιών. Ναι, ναι, ναι, ναι, αυτό που λένε είναι τέρας αυτό το άτομο, αλλά ποιος είναι το τέρας, είναι η δικαιοσύνη η ίδια που δεν έριξε μια ματιά στην περίπτωση αυτών των παιδιών. Εμείς όταν, όταν ε, καταγγέλουμε τις περιπτώσεις αυτές ε, μας φέρονται σαν να είμαστε σκουπίδι, σκουπίδια οι αρχές και η δικαιοσύνη. Εντάξει, πρώτη φορά τώρα εδώ. Όταν μιλάμε για ένα κρατούμενο ναι, και ρωτάμε ότι κάποιο που, που ε, κάποιον που υποφέρει από μια καρδική πάθηση. Γιατί τον ξυπνάτε κάτι ταρτάκι. μα, λένε, αν δεν τον ξυπνάμε, πάμε να δούμε, τον ενοχλούμε για να δούμε αν είναι ζωντανός ακόμα ή όχι. Και πολλά πράγματα βλέπουμε παρόμοια και έχουν να κάνουν ε, με περιπτώσεις που δεν τους αρέσει στο κράτος ε, παρόμοιε. Έχουμε στην Ολλανδία, στο Βέλγιο, πολλέ στη Γαλλία, Πολλέ περιπτώσει και τι διαπιστώνουμε εκεί που οι δικαστική. Όταν έχουμε στο εφετείο, πολλές, όταν έχουν στο εφετείο πολλές περιπτώσεις, ε, οι δικαστές των οποίων οι περιπτώσεις ε, συστηματικά αυτών των δικαστών πηγαίνουν σε εφετείο τιμωρούνται, κρίνονται μάλλον σε μας τίποτα ε, ο κράτος ε, την πληρώνει όχι ο δικαστικός Καθώς τη βγάζει ωραία. Αλλάζουν τα στοιχεία, εξαφανίζεται το θύμα, αυτή που δεν υπάρχει θύμα, δεν υπάρχει και κύκλωμα εγκληματικό. λοιπόν ο εγκληματία παραμένει ατιμόρυτος. Ε, εντάξει, δεν ασκούμε κριτική τους νόμους είναι για την προστασία των παιδιών. Είναι καλοσυνταγμένοι οι νόμοι, αλλά είναι και καλοί από τη στιγμή που εφαρμόζονται σωστά. Αν έχουμε τώρα εμείς νόμους που δεν, υποχρε... δεν ε, σε... εφαρμόζονται υποχρεωτικά γιατί αποτελούν κρατικό απόρριτο, τότε υπέροχος ο νόμος χωρίς νόμο όμως ουσιαστικά. ρωτιέται κανείς πώς θα μπορούν να εφαρμόζονται αυτοί οι νόμοι. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς μπορούν να υποχρεώσουν ε, τα κράτη να εφαρμόζουν τους νόμους αυτούς ε, και επίσης αντιμετωπίζουμε διάφορα προβλήματα σε παιδικά εγκλήματα ε, τα έχουμε μερικές φορές αλλά το ίντερνετ ε, ε ε, έχουν ρίξει τα σύνορα το ίντερνετ, ε, ξέρω δεν υπάρχουν πια σύνορα, η παραγωγή γίνεται τόπου όμως ε, και έχουμε και θέματα που αφορούν 36 χώρες ας πούμε. Μας χάρη το Βέλγιο που είναι ένα σκάνδαλο για την Ευρώπη. Όταν εκεί βλέπουμε η γαλλική πτυχή του εγκλήματος δικάστηκε βάσει έλλειψης όμως 1.800 πιστηρίων. Ε, ξέρουμε ότι υπάρχουν τόσοι, αλλά τόσα... Όχι 1.800, συγγνώμη, 80.000 λέει τώρα. Ε, και καταδικάστηκε όμως. Αγνοούν ότι δεν υπάρχουν πια αυτά τα στοιχεία. Τι γίνεται, τι χρησιμεύει τότε ένας φάκελος, τι χρησιμεύουν αυτά τα πιστήρια. Και επίσης δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στο φάκελό της γιατί επαναλαμβάνομαι είναι απόρριτο Α, λοιπόν, 80.000 ε, ενδείξεις, πιστήρια κλπ. Δεν υπάρχουν πια στο φάκελό της, δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στο φάκελό της. Τι κάνουμε εδώ, τους κλείνουμε έτσι στη φυλακή. Αυτό στη Γαλλία. Και μια περίπτωση παρόμοια στο Βέλγιο, αλλά οι βελγικές αρχές ε, ουσιαστικά θέλουν να δολοφονήσουν το άτομο αυτό και ο υπουργό δικαιοσύνη του πρότεινε ο ίδιος ε, να πάρει ένα χάπι που θα προκαλέσει ε, προσβολή και προσπάθησαν και οι γιατροί να τον ξεκάνουν και μετά μια περίπτωση ε, επέζησε 42 μέρες αλλά 42 μέρες μετά αποφάσισε ο Υπουργός Δικαιοσύνη εντάξει ε, περισσότερο ανθρώπινες συνθήκες κράτησης. Βλέπουμε παρόμοιες περιπτώσεις, βλέπουμε παρόμοιες εγκλήματα, υπάρχει κόσμος πολλής που διαμαρτύρεται. Εντάξει, ολοκλήρωσα κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Για να απαντήσει η Επιτροπή τώρα. Σέζαρ Αλόνσο Ριάρτε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Τρία διαφορετικά ζητήματα έχουμε στην αφορά αυτή και διαφορετική απάντηση πρέπει να δώσουμε στο καθένα. Το πρώτο αφορά ένα αριθμό υποθέσεων όπου η αναφέρουσα λέει ότι αθώοι άνθρωποι ουσιαστικά έχουν καταδικαστεί και ένοχοι έχουν απελευθερωθεί, έχουν αθώθει. Το δεύτερο ζήτημα έχει να κάνει με τη λειτουργία του δικαστικού συστήματος, το οποίο υπολειτουργεί ή δεν λειτουργεί σωστά σε διάφορα κράτη-μέλη ιδίως το πολύ σοβαρό ζήτημα της σεξουαλικής εκμετάλλευσης των παιδιών. Νομίζω λοιπόν ότι τα ζητήματα αυτά θα πρέπει να αναλυθούν ξεχωριστά. Ξεχωριστές δηλαδή περιπτώσεις όπου ένοχοι έχουν ε, καταδικαστεί, συγγνώμη, ένοχοι έχουν αθωωθεί και αθώοι έχουν καταδικαστεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προς το πρώτο αυτό ζήτημα, ως πρώτη αυτή υπόθεση δεν μπορεί να πει τίποτα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι, θετικό, δεν είναι ε, δικαστήριο στο οποίο μπορεί να κάνει κανείς έφεση και δεν μπορούμε εμείς να θεωρήσουμε καμία τέτοια δικαστική υπόθεση. Το ζήτημα αυτό βρίσκεται εντελώ εκτός των αρμοδιοτήτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με το άρθρο 72 της ε, ισχύουσα συνθήκη. Καμία δράση δεν μπορεί να ληφθεί εξ ονόματο Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το δεύτερο τώρα ζήτημα, την μη λειτουργία δηλαδή του δικαστικού συστήματο σε ορισμένα κράτη-μέλη τη Ένωση, σίγουρα η αιτία σε αυτή είναι πάρα πολύ σοβαρή. Γιατί ουσιαστικά παραβαίνει το άρθρο 6 τη Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου τη Ευρώπη και στην περίπτωση αυτή θα ξεκινούσε μια διαδικασία που προβλέπεται συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν υπάρχουν σοβαρές και επανειλημμένες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εμείς όμως θεωρούμε ότι βάσει των ισχυρισμών της αναφέρουσας δεν μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει σοβαρή ε, επαναλαμβανόμενη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλες αυτές τις χώρες, δηλαδή στην, στο Βέλγιο, τις κάτω χώρες, στη Γαλλία, την Πορτογαλία. Δεν υπάρχουν ε, τα αποδεκτικά στοιχεία προκειμένου να πούμε ότι το δικαστικό σύστημα δεν λειτουργεί στις ε, χώρες αυτές και ότι παραβιάζονται κατά αυτόν τον τρόπο τα κατοχυρωμένα δικαιώματα. Και το τρίτο τώρα ζήτημα – η ανάγκη καταπολέμησης, καταπολέμησης της σεξουαλικής εκμετάλλευσης ε, των παιδιών. Ενδεχομένω τα πράγματα εδώ είναι ακόμα πιο σοβαρά από ό,τι έχει πει η αναφέρουσα. Διάφορα επιστημονικά στοιχεία μας λένε ότι ε, ένα 10 με 20% των παιδιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικία κινδυνεύουν να πέσουν θύμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Αυτό βάσει στοιχείων που έχουμε από το 2003. Η σεξουαλική εκμετάλλευση είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό έγκλημα το οποίο αφήνει βαθιά τραύματα στο παιδί και μπορεί να εκδηλωθεί με διάφορους τρόπους. Υπάρχουν νέες μορφές ε, εγκλήματος όπως το διαδίκτυο βέβαια και η παιδική πορνογραφία ή ακόμα και ο σεξουαλικός ε, τουρισμός. Δεν έχουμε όμως ακόμα μία σαφή απάντηση αυτή τη στιγμή και το κοινοτικό δίκαιο δεν μας δίνει μία σαφή απάντηση. Έχουμε μία απόφαση πλαίσιο από το 2004 η οποία θέτει ελάχιστα επίπεδα ε, προσέγγισης των εθνικών νομοθεσιών όσον αφορά αυτό το ζήτημα της σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Πρόκειται όμως απλώς για μια απόφαση πλαίσιο, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ανα πάσα στιγμή οποιοδήποτε κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει να μην την εφαρμόσει. Δεν μπορεί να προσφύγει δηλαδή κάποιος στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο βάσει αυτής της απόφασης πλαίσιο. Και για αυτό το λόγο, μετά την ε, θέση σε ισχύ της ε, συνθήκης της Αβώνης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ένα σχέδιο οδηγίας προκειμένου να έχουμε τα απαραίτητα νομοθετικά μέτρα για να καταπολεμήσουμε πιο αποτελεσματικά την ε, σεξουαλική κακοποίηση, σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών. Η πρόταση αυτή υποβλήθηκε στις 25 Μαρτίου του 2009 και ακολουθείται πλέον η νέα νομοθετική διαδικασία, δηλαδή έχουμε ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο και συναπόφαση μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και δημόσιος διάλογος για το ζήτημα αυτό. Προσπαθούμε να καλύψουμε στο σχέδιο αυτό όλες τις μορφές σεξουαλικής εκμετάλλευσης των ε, παιδιών και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η προστασία του θύματος, η προσφυγή κατά του εγκληματία και η πρόληψη όπου αυτό είναι δυνατό θα παρουσιαστεί αύριο με περισσότερε λεπτομέρειε στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και γνωρίζουμε ότι οι προσδοκίε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πολύ υψηλέ. Υπήρχε και μια σύσταση από το Κοινοβούλιο πέρυσι προ το Συμβούλιο προκειμένου να προσαρμοστεί νομοθεσία και πιστεύουμε ότι τα αιτήματα τα οποία εξέφρασε πέρυσι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν ληφθεί υπόψη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εμείς προσπαθούμε ως Επιτροπή να προωθήσουμε το φάκελο αυτό προκειμένου να έχουμε μια πολύ ποιοτική νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα, μπορεί, θα μπορέσει να εφαρμοστεί πιο αποτελεσματικά μέσω της νέας συνθήκης. Σας ευχαριστούμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτρόπης που νομίζω ότι η απάντησή του ήταν αρκετά λεπτομεριακή και δεν ακούσαμε παρεμβάσεις μετάλλες από τους συναδέλφους. Έδειξε όμως τη διάθεση της Επιτροπής για το θέμα αυτό της αναφοράς για τις ε, υπερβολές παραβάσεις κλπ. εις βάρος παιδιών για την εξέταση του θέματος αυτού. Η αναφορά Νομίζω ότι περάτωσε την πορεία της ε, και θα μπορούσαμε να δούμε τι θα γίνει με την οδηγία. Μπορούμε να την αφήσουμε ανοιχτή ακόμα και να παροτρύνουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βιαστεί κάπως ε, για να εφαρμοστούν όλα αυτά που αναφέρονται στην ε, οδηγία. Εντάξει, συμφωνείτε, εγκρίνεται. Πάμε τώρα στο σημείο 17 με την ίδια λογική. Ποιοι είναι παρόντες από τους αναφέροντες. Είναι 813 του 2008 αναφορά. Είναι John Bryan παρόν, ο οποίος έχει και το λόγο. Sorry. Uh, thank you, Chair, for the... Ευχαριστώ, Πρόεδρε, που μου δίνετε την ευκαιρία να σας υποβάλω την ε, αναφορά μου. Έχει να κάνει με την υγεία όλων των πολιτών της Ευρώπης. Η ανησυχία μου προκύπτει από το εξής. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων ε, και το σχετικό πάνελ ε, κάνει κάποιες εκδίδει κάποιες αποφάσεις οι οποίε μπορούν να αποβούν ε, μοιραίε για την υγεία εκατομμυρίων ε, Ευρωπαίων πολιτών. Ε, το πάνελ αυτό δεν είναι εκλεγμένο και κάνει αξιολογήσει κινδύνου. Δεν, κάνει, δεν αναλαμβάνει όμως την, την ευθύνη για την ανάλυση κινδύνου και δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε νομική ευθύνη για τι αποφάσει του. Οπότε πραγματικά ε, ενίσταμε σε ό,τι αφορά την, τον τρόπο με τον οποίο η ΕΦΣΑ διεκπεραιώνει και αξιολογεί αυτέ τι επιστημονικέ αποδείξει καθορίζει την, ε, τις νομοδοτήσεις για τα γενετικώς τροποποιημένα προϊόντα. Αυτές είναι οι βασικές μου ανησυχίες ε, που αναφέρονται και με συγκεκριμένες αναφορές στην ε, αναφορά μου που σας έχω υποβάλει. Καταρχήν, η ΕΦΣΑ ε, συνήθως εκδίδει θετικές γνωμοδοτήσεις για, τις, για τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς που βασίζονται σε επιλεγμένα δεδομένα που, παρέχονται από τους ετούντες. Αυτές οι μελέτες δεν είναι αξιόπιστες γιατί αυτός που έχει την, το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας δεν θα, δεν θα επιτρέψει να γίνει ανεξάρτητη ανεξάρτητη, δεν θα επιτρέψει ανεξάρτητους ε, ε, επιστήμονες να ε, έχουν πρόσβαση στα προϊόντα του. Επίσης, δεν, οι, επιστημονικά, επιστημονικά, οι επιστημονικές μελέτες που γίνονται πρέπει να είναι επαναλαμβανόμενες εάν θέλουμε να, τις να θέλουμε να είναι αξιόπιστες. Η σύνθεση τώρα της ΕΦΣΑ και του σχετικού πάνελ δεν είναι επαρκής για να αντιμετωπίσει τις, τα αιτήματα που δέχεται. Ε, θα πρέπει να υπάρξουν επιστήμονες εκπρόσωποι από ευρωπαϊκές μη κυβερνητικές οργανώσεις και ομάδες καταναλωτών. Το πάνελ έχει μια ιστορία στενών δεσμών με την βιομηχανία γενετικώς προϊόντων και κάποιοι από τους συμπληρωμένο στο πάνελ εμπλέκονται και σε εθνικέ συμβουλευτικέ επιτροπέ, οπότε έχουν δύο δυνατότητε να επηρεάσουν τι αποφάσει. Το μεγαλύτερο πρόβλημα με την ΕΦΣΑ είναι ότι οι απαιτήσει για, για τι αιτήσει για, για γενετικώ τροποποιημένου οργανισμού δεν είναι αρκετά συγκεκριμένε ώστε να επιτρέπουν κανονικέ αξιολογήσει κινδύνου. Επίση, η Κομισιόν που έχει εκδώσει τον, το σχέδιο του εφαρμοστικού κανονισμού ε, και το έχει στείλει και στον ΠΟΕ, κάνει τα πράγματα ακόμη χειρότερα. Πρέπει λοιπόν να υπάρξουν σαφή ε, ερευνητικά πρότυπα. Πρέπει να, υπάρξουν, να είναι σαφή οι παράμετροι. Ε, μετά η έρευνα πρέπει να γίνεται όπω ακριβώ απαιτείται. Δηλαδή είναι ε, παράδεκτο να, να, να εξετάζουμε με μονομένε πρωτενε και όχι ολόκληρα τα φυτά. Να θεωρούμε ότι κάποια, κάποια, δεδομένα, κάποια προϊόντα είναι ασφαλή επειδή τα προϊόντα του είναι ασφαλή. Να ξεχνούμε επιδράσεις που έχουν ε, όλες αυτές οι ουσίες στον οργανισμό. Ο εφαρμοστικό κανονισμό θα μπορούσε να λύσει αυτά τα προβλήματα, αλλά με την παρούσα ε, μορφή του πραγματικά βάζει πολύ νερό στις ε, κατευθυντήριε γραμμέ τη ΕΦΣΑ η ΕΦΣΑ δεν κάνει πλήρη και δεν εκδίδει πλήρω και εγκαίρω τα δεδομένα που υπάρχουν μέσα στι αιτήσει για του γενετικού οποποιημένου οργανισμού. Οι ανεξάρτητε αυτέ έρευνε μπορούν να ε, γίνουν μόνο μετά από την δημοσίευση ε, λόγω τη χρήση ε, του δικαιώματο τη εμπιστευτικότητα. Η ΕΦΣΑ αναγκάστηκε μόνο σε μία περίπτωση να δημοσιεύσει την απόφασή της. Ε, και θα ήθελα να ζητήσω επίσης και κάποιες ε, δράσεις που θα πρέπει να αναλυφθούν. Πέρα από τα πολλά σοβαρά προβλήματα που έχω, σας έχω αναφέρει, θεωρώ ότι δεν είναι πολύ αργά για το Κοινοβούλιο να αναλάβει δράση για να αυξήσει την εξουσία του σε ό,τι αφορά την πολιτική για του γενετικώ οπημένου οργανισμούς και να ενισχύσει την προστασία των Ευρωπαίων πολιτών. Η Κομισιόν και η ΕΦΣΑ φαίνεται ότι έχουν κάνει ελάχιστα πράγματα για να εφαρμόσουν τι συστάσει του, Ευρω... του Συμβουλίου περιβάλλοντο τη 4 η Δεκεμβρίου του 2008. Οπότε ζητώ από την Επιτροπή να υποβάλει τις, ε, τις ε, ε, στο Κοινοβούλιο. Να, μπει στο, να καταγραφεί στα πρακτικά ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να επιμείνει η ΕΦΣΑ και το συγκεκριμένο πάνελ να αναθεωρηθεί ώστε να υπάρχει καλύτερη εκπροσώπηση. Ε, να, επίσης όλες οι, ε, θα πρέπει να υπάρχουν αντίτυπα όλων των αιτήσεων και οι ετούντε θα πρέπει να μπορούν να ε, επιβεβαιώνουν γραπτό ότι θα δώσουν τα, ότι θα δώσουν τα, τα πρωτότυπα προϊόντα στους ε, ανεξάρτητους ε, ερευνητές. Ε, εάν αυτό είναι απαραίτητο. Επίση, ζητώ το, το Κοινοβούλιο να, καταψηφίσει με, να καταδικάσει με ψήφισμα το εξή. Την ε, υπερβολική εξάρτηση από τι επιστημονικέ αποδείξει που, που βρίσκονται στον έλεγχο του ετούντο. Η χρήση των αποτελεσμάτων από, από επιστημονικά ε, πειράματα τα οποία για οποιοδήποτε λόγο δεν, δεν υπάρχουν αντίτυπα να μπλοκαριστεί η ανεξάρτητη έρευνα μέσω μη ε, συνεργασίας ε, με, τους, ε, με όσους έχουν τις, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Επίσης, οποιαδήποτε, δυνατότητα της, οποιαδήποτε προσπάθεια της ΕΦΣΑ να βάλει νερό ή να ε, ε, επιταχύνει τη διαδικασία για την έγκριση των μελλοντικών προϊόντων ή των ελληνικών τροποποιημένων προϊόντων. Να καταδικαστεί επίσης οποιαδήποτε προσπάθεια να, απλοποιηθεί, να απλοποιηθούν οι απαιτήσει για την ασφάλεια. Ζητώ από το Κοινοβούλιο να επιμείνει ότι οι ε, κατεξοχήν ανεξάρτητε μελέτε που σχετίζονται με την ασφάλεια των υγειονομικών τροποποιημένων οργανισμών να υποβάλλονται πάντα στην διαδικασία αξιολόγηση κινδύνων και να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Ζητώ από το Κοινοβούλιο να υπάρξει μεγαλύτερη εμπλοκή των, των κρατών μελών στι αξιολογήσει κινδύνου και να θυμίσετε στην ΕΦΣΑ και στην Κομισιόν ότι όπου υπάρχει αβεβαιότητα και διαφωνία η αρχή τη ε, ε θα πρέπει να ε, μπαίνει στο παιχνίδι έτσι ώστε να υπάρχει υπάρχει μεγαλύτερη δυνατή προστασία για του Ευρωπαίους πολίτες. Χαίρομαι που μου δώσατε την ε, δυνατότητα να μιλήσω στην Επιτροπή σα και ζητώ να, την μελετήσετε, να μελετήσετε όλα αυτά τα σημεία που σα ανέφερα προσεκτικά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Εκπρόσωπο τη Επιτροπή, Σεβαστιαν Γκουκ. Κύριε Πρόεδρε, σα ευχαριστώ. Να σας επαναλάβουμε ότι το θεωρούμε το θέμα αυτό σαν ε, απόλυτη προτεραιότητα και ότι θα επαγρυπνούμε ώστε οι σπόροι και διάφορα αυτών των οργανισμών να διατίθενται στην αγορά παρά μόνο αν δεν είναι επιβλαβή για την υγεία των ζώνη ή των ανθρώπων. Και εμείς εμπιστευόμαστε την εργασία της ΕΦΣΑ και θα συνεχίσουμε την εργασία μας ακριβώς βάσει των νομοδοτήσεών της. Τώρα για την εξοδότηση πιστοποίηση για τη διαδικασία τα κράτη-μέλη και η ΕΦΣΑ καταβάλουν προσπάθειε που έχουν σημασία ώστε αυτοί οι τροπημένοι οργανισμοί να διατίθενται μόνο αφού εξεταστούν λεπτόμερος με ιδιαίτερη προσοχή. Αυτά τελευταία χρόνια οι προσπάθειε, ε, οι εξή έγιναν και οι πρωτοβουλίες οι εξή. Πρώτα απ' όλα για οποιαδήποτε άδεια από την ΕΦΣΑ ένα αίτημα υποβάλλεται στο κράτος μέλος ε, που μπορεί να κάνει τα σχόλια όπως προβλέπεται από τον εγγονισμό. Τα σχόλια αυτά αναλύονται από πλάση της ΕΦΣΑ και στη συνέχεια εντάσσονται στη γνωμοδότηση της ΕΨΑ με ένα ειδικό παράρτημα που τα συμπεριλαμβάνει αυτά τα σχόλια και τον τρόπο με τον οποίο η ειδική ομάδα που ασχολείται με του τροπομένου οργανισμού τα έχει λάβει υπόψη και ακόμα για την σχετική άδεια. Ε, χρειάζεται χρόνο από πλευρά ΕΦΣΑ για να κάνει την εκτίμηση αυτών των θεμάτων ε, αρκετές φορές και άλλοι συμβαλόμενοι θεωρούν ότι χρειάζεται πολύς χρόνος για αυτή τη διαδικασία και ένας από τους λόγους είναι ότι η ΕΦΣΑ απαιτεί από όσου υποβάλλουν την αίτηση συμπληρωματικέ πληροφορίες πολλές φορές σχετικά με το πόσο ασφαλής είναι αυτοί οι τροποποιημένοι οργανισμοί, δηλαδή διάφορε πληροφορίε, διάφορες δοκιμές συμπληρωματικέ και η γνωμοδότηση δίδεται μόνο από τη στιγμή που θα υπάρχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θεωρεί η ΕΦΣΑ ότι χρειάζεται να διαθέτει για να είναι ασφαλές το προϊόν όπως θα κριθεί στην γνωμοδότηση αυτή και θα μπορούσε να βελτιωθεί το σύστημα με την πρόταση κανονισμού ας πούμε που έχει να κάνει με την άδεια που σε αυτούς τους τροπικούς και για το, την αίτημα που θα πρέπει να υποβάλει κάποιος η πρόταση αυτή θα βελτιώσει ιδιαίτερα ακόμα περισσότερο την όλη διαδικασία για την έκδοση άδεια. Βασίζεται στι κατευθυντήρε γραμμέ που έχει η ΕΦΣΑ και τώρα εδώ και δύο χρόνια είναι αντικείμενο λεπτομερών συζητήσεων με τα κράτη-μέλη και με τις ε, διάφορες επιστημονικές επιτροπές των κρατών μελών που συμμετέχουν στην σύνταξη του λόγου κανονισμού που προχωράει και σε ένα δις πρωτοκόλλου που δεν υπάρχει σε, εθνικό επίπεδο και λέει ποιο πρωτόκολλο θα πρέπει να ισχύει και σε ποια ακριβώς κατάσταση. Συνεχίζουμε την εργασία μας πάνω σε αυτόν τον κανονισμό, συνεργάζονται όλα τα κράτη-μέλη, λαμβάνονται υπόψη μας βέβαια τα διάφορα σχόλια τα οποία γίνονται από άλλους με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Σας ευχαριστώ, λέει πρόεδρος Μπελιέ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η αναφορά αυτή μας καλεί να προσέξουμε τρεις βασικές αρχές στον τομέα της ε, υγείας των καταναλωτών και ουσιαστικά μας, μας ζητά ουσιαστικά να δούμε ποια είναι η πρόσβαση πληροφορίες και πόσο διαφανείς είναι οι πληροφορίες αυτές όσον αφορά την αξιολόγηση των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών και μας καλεί επίσης να εξετάσουμε την πολυεπιστημονικότητα και την μεροληπτικότητα ή όχι των μελετών που γίνονται και που επηρεάζουν πολύ τις επιλογές που κάνουν οι ευρωπαϊκές κοινωνίες και μας ε, καλεί επίσης η αναφορά αυτή να δούμε πώς εφαρμόζεται η αρχή της ε, πρόληψης. Συμφωνώ με τα όσα είπε ο Ναφέρον και θα ήθελα να πω ότι στα πλαίσια της Επιτροπής Περιβάλλοντος στις 5 Οκτωβρίου 2009 είχα τη δυνατότητα να μιλήσω με τη Διευθύντρια της ΕΦΣΑ για ζητήματα που είχαν να κάνουν με το καλαμπόκι της Μονσάντο 810 και την ε, ρώτησε αν ήταν σε θέση πραγματικά να μας πει με σιγουριά ότι οι έρευνες που κάνει η ΕΦΣΑ για τον περιβαλλοντικό και υγειονομικό αντίκτυπο των ε, τροφίμων αυτών ήταν ουσιαστικά βιώσιμες, αν μπορούσαν ουσιαστικά να δώσουν αποτελέσματα μακροπρόθεσμα. Η διευθύντρια της ΕΦΣΑ αναγνώρισε τότε με απόλυτη ειλικρίνη ότι δεν ίσχυε κάτι τέτοιο και ότι οι αξιολογήσεις όσοι έχουν σήμερα και ως γίνονται σήμερα από την ΕΦΣΑ δεν μας επιτρέπουν να έχουμε μια αξιολόγηση των υγειονομικών και περιβαλλοντικών κινδύνων μακροπρόθεσμα. Το δεύτερο ερώτημα είχε να κάνει με το καλαμπόκι 810 και πιο συγκεκριμένα με τις αναλύσεις που γίνονται από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, αναλύσεις που είναι πολλές φορές αντιφατικές σε σχέση με τις αναλύσεις της ΕΦΣΑ. Και πάλι η Διευθύντρια της ΕΦΣΑ αναγνώρισε ότι όντως οι αναλύσεις αυτές από εξωτερικούς αναλυτές, συμπληρωματικές δηλαδή σε σχέση με την ΕΦΣΑ, δεν είχαν ληφθεί υπόψη. Σα τα λέω όλα αυτά για να σας πω ότι σήμερα σε απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις, στα σημαντικά αυτά ζητήματα τα οποία έθεσε ο αναφέρον, στα τρία αυτά ζητήματα διαφάνεια, πρόσβαση πληροφορίες, επιστημονική αξιολόγηση και εφαρμογή της αρχής της πρόληψης σε περίπτωση αφιβολίας, Υφίστανται λοιπόν τα ζητήματα αυτά, υφίστανται τα προβλήματα αυτά και απαντήσεις μας δίνει προς αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αρκούν. Δεν μπορούμε δεδομένων των όσων διακυβεύονται για το ενηγεία και το περιβάλλον από τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς να ακολουθήσουμε μια διαφορετική στάση, στάση δηλαδή η οποία δεν θα είναι η απόλυτη επιμονή προκειμένου να έχουμε πλήρες πληροφορίες. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να λέμε ότι όλα βαίνουν αισίως. Έχουμε σε εξέλιξη έναν κανονισμό ο οποίος αργότερα θα μας δώσει κάποιες απαντήσεις. Ολοκληρώνοντας θα ήθελα να πω ότι ε, πρέπει η αναφορά αυτή να μείνει ανοιχτή προκειμένου να καταφέρουμε να εξετάσουμε και εμείς περισσότερο το, το περίφημο αυτό κανονισμό που επεξεργάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δούμε τελικά αν ο νέος, κανονισμός μπορεί να απαντήσει τις ανησυχίες του αναφέροντος. Ευχαριστώ. Thank you, President. Ευχαριστώ, Πρόεδρε τεράστιο το θέμα αυτό. Και πολλοί, όπως και εγώ φαντάζομαι, πιέζονται από τους ψηφοφόρους τους. Για πολλά χρόνια ήμασταν σε διέξοδο για τις εγκρίσεις των γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών, κάτι που δείχνει την ευαισθησία που υπάρχει γύρω από αυτό το θέμα. Φυσικά υπάρχει θέμα εμπιστοσύνης των καταναλωτών, διαφάνειας, ασφάλειας, αξιοπιστίας ο αναφέρον αναφέρει πολύ συγκεκριμένα ζητήματα, θέτει πολύ βασικά ερωτήματα που δεν έχουν απαντηθεί από την Κομισιόν. Εγώ έχω διαβάσει την απάντηση της Κομισιόν και άκουσα και σήμερα πολύ προσεκτικά τι είπε, αλλά εξακολουθούν να μην έχουν απαντήσει στα συγκεκριμένα θέματα. Πολύ συχνά όταν συζητούμε τέτοια θέματα όπως οι γενετικώ τροποποιημένοι οργανισμοί, πολλοί μιλούν για την ανάγκη τη επιστήμης, ότι δηλαδή δεν πρέπει να βασίζουμε τι αποφάσει ε, στη... δική μα αίσθηση, αλλά σε επιστημονικά δεδομένα. Θέλουμε αξιόπιστα, αμερόληπτα, επιστημονικά δεδομένα και πληροφορίε που να βασίζονται σε έρευνα. Όχι μόνο έρευνα που κάνουν οι εταιρείε και οι ετούντε, εντάξει να λαμβάνεται και αυτή η υπόψη, αλλά και έρευνα που να γίνεται από άλλου έρευνα που να γίνεται από ανεξάρτητους φορείς. Ξέρω ότι ο Dr. Brian John έχει αποστείλει πολλές πληροφορίες και στο παρελθόν και δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν μπορεί να γίνει, δεν μπορεί να μοιραστούν αυτές οι πληροφορίες ή να είναι δημόσιες αυτές οι πληροφορίες που βασίζονται σε επιστημονικές έρευνες. Αυτό που λέει η Κομισιόν σήμερα, για τον τρόπο δηλαδή που προχωράει όλη η διαδικασία, εξακολουθεί να μην απαντάει στο ερώτημα που έχει τεθεί για το πώς, αν δηλαδή, τα τεστ μπορούν να ε, δημοσιεύονται, μπορούν να δημιουργούνται αντίγραφα, να υπάρχουν πληροφορίες. Εμείς ως Κοινοβουλίο έχουμε ε, ευθύνη να οι πληροφορίες που δίνουμε να είναι αμερόληπτες, να είναι αποδεδειγμένες και τώρα εντάξει γίνονται και συζητήσεις για, τους, ε, για τον κανονισμό. Νομίζω όμως ότι Είναι επιτέλους η στιγμή να το δούμε το θέμα αυτό, να το μελετήσουμε πιο προσεκτικά, ώστε ίσως να καταλήξουμε και σε ένα ψήφισμα, όπως ζητά ο, ε, το, ο αναφέρον. Και να δούμε ποιοι είναι οι τρόποι με τους οποίους οι καταναλωτές, οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις μπορούν να, λάβουν, ε, να συμμετάσχουν ε, και ίσως στην έρευνα. Οπότε υποστηρίζω την ομιλήτρια που μίλησε πιο πριν Όντω είναι η σωστή στιγμή για να μπούμε στο βάθος του... της υπόθεσης, γιατί πραγματικά αυτό το θέμα αφορά πολλού. Um, Κυρία Πρόεδρε, θα είμαι πολύ σύντομος, γιατί ξέρω ότι ακολουθούν και άλλες αναφορές. Το ζήτημα πάντως είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας είπε ότι ε, ανέκαθεν έθετε τις ε, περιβαλλοντικές ανησυχίες ως μία από τις πιο βασικές της προτεραιότητες. Αντίθετα, εγώ πιστεύω ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επηρεαστεί πάρα πολύ από τις, ε, μεγαλο, από τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, οι οποίες προωθούν τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα σε διάφορες χώρε χώρες και σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Το ζήτημα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχει να κάνει με την ακαιρεότητα των οικοσυστημάτων μας, του περιβάλλοντός μας, έχει να κάνει με την ασφάλεια των τροφίμων και τώρα και στο μέλλον. Θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα υπεροπτικό να θεωρούν οι επιχειρήσεις αυτές ότι μπορούν να μετατρέψουν ουσιαστικά το οικοσύστημά μας, το οποίο διαμορφώθηκε μετά από εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια. Χρειάστηκε κανείς, μάλλον χρειάστηκε να περάσουν πάρα πολλά χρόνια προκειμένου τα φυτά αυτά να προσαρμοστούν στο περιβάλλον το οποίο έχουμε και να μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι απαράδεκτο αυτή τη στιγμή να καλλιεργούνται τεράστιες εκτάσεις με γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς για τους οποίους δεν γνωρίζουμε πώς θα εξελιχθούν μακροπρόθεσμα. Δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσουν σε σχέση με τις κλιματικές αλλαγές ή σε σχέση με άλλες περιβαλλοντικές δραματικές αλλαγές που μπορούν να γίνουν στο μέλλον. Συμφωνώ λοιπόν με τον αναφέροντα όσον αφορά την ανεξαρτησία, τη διαφάνεια, την δυνατότητα εξακρίβωσης των επιστημονικών αποτελεσμάτων, των δοκιμών και μία από τις ε, επιχειρήσεις αυτές που μας έδωσε γενικά τροποποιημένους οργανισμούς ε, και ουσιαστικά ελέγχει πάρα πολλές ε, πρωτεύουσες, μας έδωσε το παρελθόν και το το πορτοκαλί παράγοντα. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει το Orange Agent. Πρέπει να είμαστε πάρα, πολύ προσεκτικοί λοιπόν. Briefly, first. Σύντομα, Πρόεδρε. Ναι, να προτείνουμε ψήφισμα του Κοινοβουλίου για να πιέσουμε την Κομισιόν να υποβάλει μια συνεκτική πρόταση. Δεύτερον, θα πρέπει η αναφορά αυτή να πάει στην Επιτροπή ΕΝΒΗ για να μας πούν την άποψή του πριν λάβουμε οποιαδήποτε άλλη απόφαση και γιατί όχι να ε, οργανώσουμε μια ακρόαση στο Κοινοβούλιο. Γιατί το θέμα αυτό δεν είναι απλώς αντιφατικό, είναι ένα από τα θέματα κλειδιά που υπάρχουν στην ατζέντα της Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Είχαμε αρκετέ ε, περιπτώσεις ε, σημαντικής κριτικής από την ΕΦΣΑ Είναι πραγματικά πολύ ανησυχητικό το γεγονός και να προσθέσω εδώ ότι ειλικρινά αρνήθηκαν να χρησιμοποιήσουν την αρχή της ε, πρόληψης. Στον δανεικό τύπο λένε ότι η νανοτεχνολογία δημιουργεί προβλήματα όπως αυτά που δημιουργούσε ε, ο αμίαντος. Δεν το υπιέψα αυτό αλλά ακούγεται και αυτό. Και αυτό είναι ένα επιχείρημα για να μην χρησιμοποιηθεί η αρχή της πρόληψης. Νομίζω ότι πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ώστε να χρησιμοποιείται αυτή η αρχή. Η Μονσάντο είναι από τα πιο ε, οργανωμένα λόμπι που έχουμε εδώ στην ε, Ευρώπη. Μετά από τους πυρηνικούς νομίζω είναι οι πιο... αυτοί που κάνουν την πιο εντατική δουλειά ό,τι αφορά το λόμπι στην Ευρώπη. Eh, Σας ευχαριστούμε. Θα μπορούσαμε να ζητήσουμε από την Επιτροπή Περιβάλλοντος για την αναφορά αυτή να μας πει μερικά πράγματα για την δική τους εργασία εκεί σε αυτή την Επιτροπή και μετά με την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή και μετά και από την αυριανή συζήτηση με, για την βιοπικιλότητα να δούμε την τροπή περιβάλλοντος τι θα μπορούσε να γίνει και ορισμένες υποδείξεις για την κατάσταση αυτή την οποία αντιμετωπίζουμε. και μετά να οργανώσουμε μια κοινή ακρόαση με την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Θα ζητήσουμε λοιπόν να συνεργαστούμε με την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Αυτά. Τελευταίες ε, δύο αναφορές είναι παρόντες οι αναφέροντες. Παρακαλώ σύντομα, σύντομα το 19... 1037 Τζιλμπέλ Ιρλανδικής Ιθαγένειας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την Επιτροπή σας. Θα, αναφέρω και τις, θα παρουσιάσω και τις δύο αναφορές ε, εκ μέρους του Τζιλ Μπελ. Ρόμπερτ Βέκερ ονομάζομαι εγώ. Υπάρχει μεγάλη σύνδεση μεταξύ της τελευταίας αναφοράς που ακούσαμε και της δικής μας. Τα θέματα αυτά σχετίζονται με αξιολογήσεις κινδύνων που κάνει η ΕΦΣΑ. Και με πολλούς τρόπους βλέπουμε γενετικώς αποποιημένους οργανισμούς που έχουν ε, πολλά ερωτηματικά και σε, πολλούς, σε πολλές περιπτώσεις παίρνουν το πράσινο φως. Βλέπουμε ακόμη και η ΕΦΣΑ στις πρόσθετα, στα πρόσθετα τροφίμων να εγκρίνει τέτοια, α, τέτοιες ουσίες. Ε, ουσίες που ουσιαστικά αποτελούν φάρμακα. Και αυτό που λέμε είναι ότι όταν γίνονται αξιολογήσεις ε, κινδύνων και αναλύσεις κινδύνων, ή διαχειρήσεις κινδύνων από την Κομισιόν, τα δύο πρώτα από την ΕΦΣΑ, όταν λοιπόν γίνονται και ισχύουν ή ε, λαμβάνονται υπόψη για τις ε, έρευνες που κάνει η Κομισιόν, για τα ανώτατα ή ελάχιστα επίπεδα ύπαρξη αυτών των ουσιών στα προϊόντα, ε, βλέπουμε πολύ περιοριστικό καθεστώς να επικρατεί. Τέσσερα προβλήματα θα σας αναφέρω. Και δίνουμε και τέσσερις πιθανές λύσεις στην Επιτροπή. Και θα το κάνω αυτό σε λιγότερο από πέντε λεπτά. Πάνω από 100 εκατομμύρια άνθρωποι, περίπου 20% του ευρωπαϊκού πληθυσμού που λαμβάνει πρόσθετα τροφίμων. Αντίθετα σε ό,τι λέγεται, αυτό σχετίζεται με άτομα που έχουν υγιή διατροφή και όχι με όσους τρώνε ό,τι να είναι. Βεβαίω η χρήση του είναι διαφορετική ανάλογα με τα κράτη-μέλη και ανάλογα με τι διάφορε πληθυσμιακέ ομάδε. Υπάρχουν πολλέ ανησυχίε γιατί κινούμαστε προς την παγκοσμιοποίηση της παροχής τροφίμων και στην διαθεσιμότητα των τροφίμων που τα μικροθρεπτικά επίπεδα αυξάνονται επικίνδυνα. Για να ενισχύσουμε λοιπόν την ε, δυνατότητα επιλογής θα πρέπει να δημιουργήσουμε έναν καθεστοτικό περιορισμό, αν μπορώ να το πω έτσι, ε, από την Κομισιόν δυνάμει του άρθρου 5 για την οδηγία, τις οδηγίες για τα προστάτα τροφίμων. Βέβαια αυτός δεν είναι ο μοναδικός τρόπος για να αντιμετωπίσουμε διάφορες ασθένειες. Γιατί περίπου 12% ε, της, ε, του πληθυσμού της Ευρώπης ας πούμε έχουν δυσαναξία στη γλουτένη. και πρέπει να ή μπορεί να, υπάρξουν, ή μπορεί να ομάδες που έχουν ε, δυσανεξία στη λακτόζη και απαγορεύεται να προσλάβουν οποιαδήποτε ε, γαλακτοκομικά προϊόντα. Ήδη από το 80 ξεκίνησε στις ε, είπα ε, το, η τάση αυτή και θα δείτε εδώ στη μέση αυτού του διπλού μοντέλου ένα αποδεκτό ρυθμό πρόσληψης το πάνω κομμάτι είναι αυτό που ισχύει και το υπόλοιπο είναι αυτό που είναι επιβλαβές. If you like, versions of no adverse effect Υπάρχουν τα όρια λοιπόν, τα κατώτερα αποδεκτά όρια, τα οποία παρόλα αυτά δεν είναι απολύτως αποδεδειγμένα. Τα υψηλά όρια βρίσκονται στα πλαίσια του, των αποδεκτών ορίων. Η Κομισιόν αυτή τη στιγμή προσπαθεί να αφαιρέσει, να μειώσει το, ε, και να, να βγάλει αυτά τα επίπεδα από το γενικό επίπεδο, ώστε να αυξηθούν τα γενικώ επιτροπόμενα επίπεδα. Τέσσερα βασικά σημεία θέλω να σας πω. Υπάρχουν πολλά ακόμη. Τα ανώτατα όρια της ΕΦΣΑ είναι το σημείο εκκίνησης για, την, για τον καθορισμό των, των ανώτατων όριων και το αποτέλεσμα είναι ότι δεν είναι ε, αποδεκτά. Για τις βιταμίνες και τα μέταλλα, ε, η ομάδα υπεργνωμόνων από, από τις 32 είπε ότι μόνο 8 μπορούν να υπολογιστούν ε, αξιόπιστα. Όλα τα υπόλοιπα είναι σε επίπεδο καθοδήγησης. Και μάλιστα λέει η έρευνα, ότι αυτό δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως ασφαλή άνωτα όρια και αυτό δημιουργεί πρόβλημα για τον τρόπο με τον οποίο η ΕΦΣΑ χρησιμοποιεί τα όρια. Δεύτερον, δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψη η εξαίρεση της βιταμίνης Β3 και η τοξικότητα που υπάρχει μεταξύ των διαφόρων ομάδων θρεπτικών ουσιών. Αυτό που, που γίνεται είναι ότι χρησιμοποιείται ο, πιο, πλέον τοξικός, η πλέον τοξική μορφή του κάποια θρεπτικής ουσίας. Τρίτον, τα βασικά συστήματα ή μοντέλα τα οποία μελετάει η Κομισιόν θεωρούν ότι το όριο μεταξύ του επιτρεπτού και του ανώτατου ορίου αντικατοπτρίζει το σχετικό κίνδυνο. Και αυτό δεν συμβαίνει. Γιατί εξαρτάται από το ποιο είναι ο κίνδυνο. Αν ο κίνδυνο είναι ε, η πατική ανεπάρκεια, ε, πρέπει να ληφθεί υπόψη ο κίνδυνο για να οριστεί και το όριο. Και τέταρτον, αυτό που καταδεικνύουμε μέσω των αξιολογήσεων ομοτήμων είναι ότι οι κίνδυνοι και τα ωφέλη συνήθω επικαλύπτουν ένα τον άλλον. Οπότε αν υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι προορισμοί πρέπει, μπορεί να σημαίνει αυτό ότι πρέπει να αφαιρέσουμε, να επαλείψουμε οποιοδήποτε κίνδυνο για όλο τον πληθυσμό. Θα δείτε ότι η πλειοψηφία δεν απολαμβάνει των ωφελημάτων αυτών των μελετών. Και βλέπετε εδώ στην διαφάνεια μια πολύ τυπική παρουσίαση και θα δείτε ότι αν αποτρέψετε κάποιον να φτάσει στο ανώτατο επιτρεπτό η πλειοψηφία δεν θα έχει να ωφεληθεί καθόλου. Τους τελευταίους μήνες δημοσιεύσαμε δύο μελέτες στην εφημερίδα ε, τοξικολογίας που είναι επίσημη ε, η επίσημη εφημερίδα και της Βρετανικής και της ε, Γερμανικής κοινότητας τοξικολογίας και καταλήγουμε ότι αυτά τα έγγραφα θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως βάση για να καθοριστεί το πώς θα προχωρήσουν οι προτάσεις της Κομισιόν και πώς το Κοινοβούλιο όταν του, δοθεί η δυνατότητα μελέτης για οποιαδήποτε πράξη, θα ορίσει ή θα συμπεριλάβει στην νομοθεσία αυτά τα ε, ανώτατα όρια και θα πρέπει να σκεφτεί πολύ προσεκτικά το πώς θα διαχειριστεί τα θέματα αυτά. Η Κομισιόν τον Ιούλιο του 2009 απέτυχε να απαντήσει στις βασικές μας ανησυχίες. Εντάξει, όλα αυτά που μας είπανε καλά ήτανε, αλλά δεν μας καθησύχασαν σε αυτά που είχαμε εμείς ως ανησυχίες. Δεύτερον, το βασικό παράπονο της Κομισιόν στην απάντησή της ήταν ότι η αξιολόγηση επιπτώσεων για τα, για τα, ήταν για τα, για τα καταστήματα που πολλούν υγιεινές τροφές. Δεν έχει δώσει όμως καθόλου ρυθμιτικά στοιχεία ώστε να χρησιμοποιηθούν για καλύτερε και πιο αξιόπιστες αξιολογήσεις επιπτώσεων. Οπότε η Κομισιόν όταν δημοσιεύει τις συστάσει της, καλό θα ήταν τότε να ξεκινούν και οι αξιολογήσεις επιπτώσεων. Και είναι σημαντικό το Κοινοβούλιο να μην θεωρεί ότι είναι κάτι δεδομένο, ότι τελεσμένο το... η δημοσίευση αυτή. Και τέλος, Επαναλαμβάνω ότι αυτά τα δύο έγγραφα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εκπρόσωπο των, της Επιτροπής ε, που θα πάρει ο τον κ. Μαθιουδάκη. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρέπει να σημειώσουμε ότι έχουμε τέσσερις αναφορές στο συγκεκριμένο σημείο που έχουν ομαδοποιηθεί Και αυτό που βλέπουμε ουσιαστικά είναι να γίνονται επικρίσεις όσον αφορά τη στρατηγική που ακολουθούμε για τη θέσπιση των ανωτάτων ορίων για βιταμίνες και ανόργανα στοιχεία σε συμπληρώματα διατροφής, ανώτατα όρια που βασίζονται σε έρευνες που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, όπως απαιτούν οι σχετικές οδηγίες. Θα ήθελα να κάνω κάποιες ε, παρατηρήσεις σχετικές με την παρέμβαση του κυρίου Βέρκερκ. Πρέπει να δούμε ότι μία από τις αναφορές εδώ είναι από έναν διατροφολόγο και στην αφορά του κυρίου Βέρκερκ γίνεται μία αναφορά στις ε, διατροφικές ιδιότητες και λέγεται επίσης ότι βασικές ανησυχίες υπάρχουν από αυτούς που χρησιμοποιούν ε, συμπληρώματα διατροφής στην ε, υγειονομική περίθαλψη που προτείνουν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν θεωρούνται φάρμακα, και επομένως εμπίπτουν στους κανονισμούς για τα τρόφιμα. Δεν θεωρούνται φάρμακα, δεν θεωρούνται μέρο ε, μια μιας θεραπεία. Ε, ε, θεραπείας. Πολλές επικρίσεις γίνονται στην αναφορά αυτή, στις οποίες βέβαια δεν έγινε αναφορά στο ότι οι βιταμίνες και την όργανα στοιχεία είναι θρεπτικά συστατικά, σημαντικά για την ανάπτυξη. αλλά λέγεται στι αναφορέ ότι θα πρέπει να γίνεται διαφορετική εξολόγηση κινδύνου. Όντω, κυρία Πρόεδρε, βιταμίνε και τα ανόργανα στοιχεία είναι βασικά τραπτικά στοιχεία και ορισμένα μπορούν όντω να παρουσιάζουν κάποιου κινδύνου αν καταναλωθούν σε υψηλέ δόσει. Συνεπώ, στόχο εδώ πέρα είναι ο στόχος της θέσπισης των ορίων είναι να εξασφαλίσουμε ότι τα προϊόντα τα οποία προσφέρονται στον καταναλωτή είναι ασφαλή και αυτό ελήφθη υπόψη από τα θεσμικά όργανα συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όταν ε, ενέκριναν τις ε, αρχές αυτές ζητώντας τα ανώτατα όρια να θεσπιστούν μέσω συγκεκριμένων κριτηρίων τα οποία αναφέρονται στην οδηγία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ως στόχο να εφαρμόσει πλήρως τα κριτήρια αυτά και όπως σας είπα ένα από τα κριτήρια είναι η χρήση των ανωτάτων ορίων όπως αυτά απορρέουν από επιστημονικές μελέτες που έχει ζητήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια Τροφίμων. Λάβαμε λοιπόν τις μελέτες αυτές και λάβαμε τις σχετικές γνωμοδοτήσεις. Ο κύριος Βέρκερ, το ακούσατε, πιστεύει ότι τα επίπεδα της ΕΦΣΑ δεν είναι αξιόπιστα. Νομίζω ότι η καταγγελία αυτή είναι πολύ σοβαρή, κυρία Πρόεδρε, και νομίζω ότι έχει και πολύ σοβαρές συνέπειες, αν γίνει δεκτή. Θα έχει πολύ σοβαρές συνέπειες όσον αφορά τις διαδικασίες που ακολουθούμε για την αξιολόγηση του κινδύνου και τη διαχείριση του κινδύνου. Οι επιπτώσεις, όπως σας είπα, θα είναι πάρα πολύ σοβαρές εφόσον δεχθούμε την καταγγελία αυτή και συνεπώς δεν μπορούμε να αποδεχθούμε την κριτική αυτή όσον αφορά την αξιολόγηση που γίνεται από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων